Συνάδελφοι, αυτό που ξεκινάμε τις συνεδριάσεις μας στις 2.30 μάλλον δεν μας βολεύει και πολύ, ίσως το ξαναλλάξουμε. Παρ' όλα αυτά, με μεγάλη μου χαρά υποδέχομαι εδώ την Επίτροπο Γκάμπριελ για πρώτη φορά από τον διορισμό της και όπως θα γνωρίζετε βεβαίως από τη θητεία σας εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, κάθε επιτροπή διοργανώνει ανταλλαγή απόψεων ε, με τους αρμόδιους επιτρόπους ε, στο πλαίσιο αυτού που ονομάζουμε διαρθρωμένο διάλογο και μιας και τελειώνει η θητεία σιγά σιγά και επίκυνται οι νέες εκλογές ε, έχουμε όπως καταλαβαίνετε πάρα πολλή δουλειά έχουμε τις προτάσεις για την ε, νέα γενιά χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Ε, προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε τη δουλειά για την αναθεώρηση της οδηγίας για τις ε, οπτικοακουστικές υπηρεσίες. Επίσης, το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2018 περιλαμβάνει μια σειρά από πρωτοβουλίες σε τομείς που είναι σχετικά νέοι για την ενωσιακή πολιτική και που αποτελούν, ε, ε, που αποτελούν προκλήσεις για την κοινωνία, σχετικά νέες. Κατά νου έχω βεβαίως τα fake news, τις ψευδείς ειδήσει και την ανάγκη να αυξήσουμε και να βελτιώσουμε τις ε, ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών. Ξέρω ότι τα θέματα αυτά σας απασχολούν και εσάς και θέλουμε χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή να σας δώσουμε το λόγο για να μας ενημερώσετε ποιε είναι οι θέσει σα, ποιε πρωτοβουλίε ε, σκοπεύετε να λάβετε. Σα παρακαλώ όμω όχι πάνω από 10 λεπτά για να έχουμε χρόνο και για ερωταπαντήσει μετά και στι προηγούμενε συνεδριάσει, ε, συζητήσει, ανταλλαγέ απόψεων είχαμε ε, δοκιμάσει αυτό το σύστημα του ping-pong που θεωρήσαμε ότι είναι και πολύ καλό ώστε μετά την εισήγησή σας οι συντονιστές να πάρουν το λόγο δύο λεπτά, τα μέλη της Επιτροπής για ένα λεπτό να μπορούν να θέτουν τα ερωτήματά σας, τους και εσείς να απαντάτε. Κάπως έτσι νομίζω ότι καθίσταται λίγο πιο ζωηρή η συζήτηση και λιγότερο, ε, παρά, παρά, λιγότερο παίρνει τη μορφή παράλληλων μονολόγων. Θα το κάνουμε έτσι λοιπόν και σήμερα. Σας ευχαριστώ και πάλι που βρίσκεστε εδώ μαζί μας. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου απευθύνατε να συμμετάσχω σε αυτό το διάλογο. Είναι πολύ σημαντικό να συμπορευόμαστε εμείς με τη δική σας Επιτροπή Πολιτισμού και Εκπαίδευσης για να ολοκληρώσουμε μαζί την, για να ενοποιήσουμε μαζί την ψηφιακή Ευρωπαϊκή αγορά. Να σας ευχαριστήσω θερμά για τον υπεκοδομητικό σας ρόλο. Σήμερα η ψηφιακή ανάπτυξη έχει τεράστιο αντίκτυπο σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου και του πολιτισμού. Και εσείς, όπως και εγώ, αναγνωρίζουμε όλοι πόσες δυνατότητες έχει ο ψηφιακός κόσμος για να ενισχύσει την επίδραση του πολιτισμού στην οικονομία και στην κοινωνία. Είναι ισχυρό μέσο για να έχουμε πρόσβαση ευρεία και πιο δημοκρατική στην κουλτούρα και στον πολιτισμό. Χάρη στη συνεργασία μας μπορούμε να τα καταφέρουμε έτσι ώστε περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες να έχουν την απαραίτητη κατάρτιση, εκπαίδευση και να έχουν πρόσβαση στα ευρωπαϊκά πολιτιστικά αγαθάτε και υπηρεσίες. Έρχομαι και παρουσιάζομαι μπροστά σας σε μια πολύ σημαντική στιγμή γιατί μένει λίγος χρόνος να μεταφράσουμε στην πράξη τις δεσμεύσεις μας για την ολοκλήρωση της ενοποίησης της ψηφιακής αγοράς. Τα τρία θεσμικά όργανα έχουν δεσμευτεί να δώσουν προτεραιότητα σε συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες τις οποίες θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας να μοιραστώ μαζί σας. Ας αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία να σεβαστούμε τις πολιτικές προτεραιότητες και να τις ακολουθήσουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόοδο, για τη δουλειά που έχει γίνει, για την οδηγία SMA, για τα ακουστικά. Θα ήθελα λοιπόν να ε, γίνει περισσότερη δουλειά σε αυτές τις νομοθετικές πρωτοβουλίες. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά ε, για τη δουλειά που κάνατε για την οδηγία DSM. Και υιοθετούμε τις προτάσεις σας πριν προχωρήσουμε πάνω στο θέμα των συγγραφικών δικαιωμάτων. Ως προς το SAPCAP, χθες έγινε ο πρώτος τριμερής διάλογος για αυτό το φάκελο με επικοδομητικό κλίμα και πνεύμα και θέλω να παρακολουθήσω την συνεργασία με τους συνομοθέτες, με τον συνομοθέτη. Επιτρέψτε μου λοιπόν τώρα να έρθω αμέσως, ευθύς αμέσως, σε ένα θέμα που με αγγίζει πολύ και με ενδιαφέρει τα μάλα, τις ψηφιακές δεξιότητες. Έχει μπει ο ψηφιακός κόσμος σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Άρα είναι απαραίτητο να αποκτηθούν νέες δεξιότητες και η πλειονότητα των εργαζομένων θα πρέπει να μπορεί να τις έχει, να τις κατέχει αυτές τις δεξιότητες. Και όχι μόνο των εργαζομένων. Τον Ιανουάριο θετήσαμε ως Κομισιόν ένα σχέδιο δράσης για την ψηφιακή δράση μέτρα για να βοηθήσουμε τα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών να προσαρμοστούν στις μεταστροφές και μετεξελίξεις στη ψηφιακή εποχή προβλέπεται ανάπτυξη απαραίτητων ψηφιακών δεξιοτήτων για να μπορεί κανείς να ζήσει και να εργαστεί σε αυτόν τον κόσμο που γίνεται όλο και περισσότερο ψηφιακός. Ωστόσο, σήμερα, αυτή τη στιγμή, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις λένε ότι οι νέοι που φεύγουν από το σχολείο δεν έχουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες. Το 40% των επιχειρήσεων στην Ευρώπη που αναζητούν ειδικού στο TIC λένε ότι δυσκολεύονται στην τεχνολογία δηλαδή, της πληροφορικής και των επικοινωνιών, δυσκολεύονται να βρουν άτομα με προσόντα. Ε, έχουμε το Digital Opportunity, ψηφιακές ευκαιρίες, μία, ένα πρόγραμμα για διασυνοριακά στάζ, μαθητείες για χιλιάδες νέους, σύμφωνα, ακολουθώντας το μοντέλο Εράσμους για την τριετία 18 με 20. Πάρα πολλές επιχειρήσεις ε, που έχουν ε, προσχωρήσει στη Συμμαχία για τις ψηφιακές δεξιότητες και, τις απασχολ... και την απασχόληση. Έχουν πει ότι είναι δεκτικές να υποδεχθούν μαθητευόμενους σε αυτό το πλαίσιο και ελπίζουμε ότι όλο και περισσότεροι νέοι θα μπορέσουν να υποφεληθούν από τέτοια προγράμματα. Από εκεί και πέρα, ένα άλλο θέμα που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερος και το οποίο θα συζητείτε όλο και περισσότερο έχει να κάνει με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το επόμενο. Είμαι πεπισμένη ότι η ευρωπαϊκή προσπάθεια δίν, παίζει σημαντικά ρόλο. Μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να αποκτήσουν καλύτερες δεξιότητες και προσόντα και να έχουν έτσι περισσότερη απασχολησιμότητα και να είναι πιο ανταγωνιστικά, να παραμείνουν πιο ανταγωνιστικά στην αγορά εργασίας. Δεν θα πρέπει όμως να αφήσουμε ανθρώπους ε, ε, στο περιθώριο. Και έρχομαι λοιπόν στο πρόγραμμα στήριξης Media. Το οπτικοακουστικό οποίο έχει αλλάξει το κοινό είναι πολύ πιο νέο και θέλει περισσότερο να έχει κατανάλωση εξατομικευμένη και διαδικτυακή. Οι πλατφόρμες διάδοσης ε, περιεχομένου οπτικοακουστικού ε, και γενικά ο χώρος των οπτικοακουστικών θα πρέπει να απεικονίζει την, τις αξίες και την κοινωνία μας. Έχουμε το βίντεο on demand, έχουμε πλατφόρμες διαμοιράσματος, έχουμε κοινωνικά μηνδία, κοινωνικά δίκτυα. Όλα αυτά δημιουργούνται από ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και πρέπει να ε, τύχουν τη στήριξή μας. Προετοιμάζουμε τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές μετά το 2020 και μετά το πρόγραμμα που θα διαδεχθεί το πρόγραμμα Media. Ε, όλα αυτά είναι πολύ λεπτά ζητήματα, τα παρακολουθούμε του σύνεγγυς και θέλω θα ήθελα να σας ζητήσω να στηρίξετε το πρόγραμμα και τις αξίες που ενσαρκώνει. Είναι η ίδια η στρατηγική στόχη για την πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία, για ανταγωνιστικότητα, για ανάγκη αναθεώρησης των δράσεων υπό το φως των νέων εξελίξεων στον νεοπτικοακουστικό τομέα και νέων προκλήσεων. Άρα χρειάζεται και προϋπολογισμός αντίστοιχος και ανάλογος με τις υψηλές μας φιλοδοξίες. Από τότε που ανέλαβα το χαρτοφυλάκιό μου, ξεκίνησα τη θητεία μου, δεσμεύθηκα όλη η ομάδα μου να συστρατευτεί και εγώ προσωπικά να αφιερώσουμε κάθε ε, δυνατή ε, προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Οι ευρωπαϊκές ταινίες κυκλοφορούν λιγότερο ε, από και διασχίζουν λιγότερο τα σύνορα από ότι οι αμερικανικές ταινίε προωθούνται λιγότερο και είναι λιγότερο ορατές στην αγορά. Η προσφορά δεν είναι αρκετά προσβάσιμη. Άρα πρέπει να ανταποκριθούμε σε κάποιες από αυτές τις προκλήσεις και γι' αυτό θα ήθελα να γίνει ένα ευρωπαϊκό ρεπερτόριο ευρωπαϊκών ταινιών. Δηλαδή, στόχος μας είναι να ξεκινήσει ένα πρωτότυπο πριν το τέλος του 2018, που είναι Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, και για να το πράξουμε αυτό θα οργανώσω μια σειρά συναντήσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς του κλάδου. Η πρώτη συνάντηση στρογγυλής τραπέζης έγινε στην Παρλινάλε του Βερολίνου, στο Βερολίνο, για να ε, εμπλέξουμε όσο να τον περισσότερους ενδιαφερομένους και να δημιουργήσουμε συνέργειες και να δώσουμε δυναμική σε όλα αυτά τα έργα. Οι επαγγελματίες να αναγνωρίσουν τους, τις χώρες όπου είναι προσβάσιμες οι ταινίε και να ξεκινήσει ο προβληματισμός για τη δυνατότητα διαδικτυακής πρόσβασης και στις χώρες που οι ταινίε είναι διαθέσιμες και μπορούν να γίνουν αντικείμενα εκμετάλλευσης και ε, στις χώρες όπου δεν είναι διαθέσιμες. Ενδεχομένως μπορούν να εξεταστούν δράσεις χρηματοδότησης της μεταγλώτησης, για παράδειγμα, των ταινιών. Σκοπός είναι να έχουμε ένα διαδικτυακό εργαλείο που θα χρησιμοποιούν οι ίδιοι οι πολίτες και θα μπορούν διαδικτυακά να έχουν πρόσβαση στην ταινία που αναζητούν. Δηλαδή να παραπέμπονται οι χρήσει εντό των υφιστάμενων υπηρεσιών video on demand στη νόμιμη οδό να κατεβάσουν την ταινία που τους ενδιαφέρει και στους νόμιμους παρόχους ε, τέτοιου είδους περιεχομένου. Ε, έχουμε και την πρωτοβουλία το ψηφιακό, η ψηφιακή εποχή και ο πολιτισμός είναι μια πρωτοβουλία που συντηρίζω. Θέλουμε να συνδέσουμε το ψηφιακό κομμάτι με την κουλτούρα και τον πολιτισμό, έτσι ώστε τα θετικά ωφέλη της κουλτούρας και του πολιτισμού στην οικονομία και στην κοινωνία να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο λόγω της ψηφιακής εποχής, λόγω του ψηφιακού χαρακτηριστικού. Η ψηφιακή αγορά δεν είναι λόγος απεσιοδοξίας, είναι πηγή ενότητας, ευημερία και αισιοδοξία. Αυτή η στρατηγική θα στραφεί γύρω από έξι βασικούς πυλώνες που έχουν να κάνουν με την διευρυμένη και πιο δημοκρατική πρόσβαση στην κουλτούρα και στο πολιτισμό μέσα από δράσεις που έχουν σκοπό να διευρύνουν το κοινό, τα ακροατήρια, δράσεις που έχουν να κάνουν επίσης με την ε, προώθηση των ταλέντων, με την αξιοποίηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, με την ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση. Και όταν έρθει η στιγμή να τα συζητήσουμε αυτά, θα επανέλθω με περισσότερες λεπτομέρειες, εάν το επιθυμείτε βεβαίως. Άλλο σημαντικό θέμα, και το είπατε και εσείς κυρία Πρόεδρε, τα fake news, οι ψευδείς ειδήσει. Κοιτάξτε, οι αξιόπιστες ειδήσει βρίσκονται στον πυρήνα κάθε δημοκρατική κοινωνία. Ωστόσο, όλο και περισσότερο ανακριβείς πληροφορίε διαδίδονται μέσω ψηφιακών σε όλο τον κόσμο. Μετά από ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που απαιτεί δράση να αναλυφθούν ε, στο θέμα της πληροφόρησης, εμείς εργαζόμαστε για να βρούμε αντισταθμιστικά μέτρα αποτελεσματικά, αρχές λειτουργικές αυτορύθμισης για τους βασικούς παραγόντες της αγοράς, και θα παρουσιάσουμε ανακοίνωση τον Απρίλιο στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Έχουμε διαβουλευτεί με τα εμπλεκόμενα μέρη, με τα κράτη-μέλη, με τις ομάδες εμπειρογνωμόνων για την εκπαίδευση και για τα μίντια. Έχουμε δημόσια διαβούλευση ανοιχτή που ολοκληρώνεται στις 23 Φεβρουαρίου. Δημιουργήθηκε ομάδα εμπειρογνωμόνων που αυτή τη στιγμή οριστικοποιούν την έκθεσή τους και ε, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τη σύνθεση ε, των πορισμάτων όλων αυτών των εργασιών. Όμως με ανησυχεί και με προβληματίζει ιδιαίτερα ο αρνητικός αντίκτυπος των ψευδών ειδήσεων στις, ε, και η αρνητική επιρροή τους στις ευρωπαϊκές αξίες και στα θεμελιώδη δικαιώματα. Πρέπει η δημόσια αρχή, τα κράτη, να είναι σε επαγρύπνηση για να υπάρχει ένα περιβάλλον επικοινωνιακό το οποίο θα είναι καθαρό και δεν θα δίνει χώρο για τέτοιου είδου ψευδείς ειδήσει. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές όταν μιλούμε για ψευδείς ειδήσει. Και η κόκκινη γραμμή είναι η ελευθερία έκφρασης και το δικαίωμα πρόσβασης στην πληροφορία. Όμως, σε αυτό το πλαίσιο ε, πρέπει να υπάρχει και χώρος για την ανάληψη ευθύνης. Πρέπει να έχουμε το θάρρος και την πολιτική βούληση, να έχουμε κοινή προσέγγιση. Και αν δεν το πράξουμε αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ε, θα ε, ε, υπάρξει ο κίνδυνος να υπάρξουν και άλλες γραμμές κατακαιρματισμού και να υπάρξουν άλλες πρωτοβουλίες που θα εμφανιστούν σε εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο κρατών, ενώ το ξέρουμε πολύ καλά ότι οι ψευδείς ειδήσει δεν γνωρίζουν σύνορα και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να δουλέψουμε όλοι από κοινού. Σταματώ κάπου εδώ για να τεθώ στη διάθεσή σας για ερωτήσεις και διευκρινήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε, για το πολύ φιλόδοξο, θα έλεγα, πρόγραμμα εργασίας που έχετε καταρτήσει. Περνάμε στη συζήτηση. Ξεκινούμε με τους ε, συντονιστές. Σίλβια Κώστα, δύο λεπτά. Ε, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί επίτροπε. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία για αυτή τη συνάντηση και είχαμε και μία συνάντηση στην ε, Μικτή Επιτροπή για τους ε, ανηλίκους, ε, προστασία ανηλίκων, ημέρα ασφαλούς διαδικτύου. Ίσως θα μπορούσατε να σταθείτε και σε αυτό. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συνάντηση και οι συγκεκριμένε προτάσεις που είχε η Επιτροπή να καταθέσει για το θέμα της προστασίας από το cyberbullying, το κυβερνό έγκλημα, το κυβερνό εκφοβισμό και βέβαια γενικότερα την ασφάλεια των νέων. Είχαμε ειδική ημερίδα τον Οκτώβριο με συγκεκριμένε ε, προτάσεις. Βλέπουμε ότι προχωρά, προχωρεί καλά η προσπάθεια αυτή και η Βουλγαρική Προεδρία φαίνεται να ε, ξεκολουθεί στο στόχο αυτό με προσήλωση. Είναι πολύ σημαντικό και να δώσουμε τα εργαλεία ε, και στους νέους αλλά και σε όποιον έχει την ευθύνη για την προστασία της αξιοπρέπειας του ανθρώπου για την καταπολέμηση του παρανομού περιεχομένου και στις κοινωνικές πλατφόρμες ε, και σε όλο το υλικό που είναι στο διαδίκτυο. Θα ήθελα να αντιληφθώ καλύτερα σε σχέση με το πρόγραμμα δράσης για την ψηφιακή ε, μόρφωση, εκπαίδευση. Σε σχέση με την ε, σύσταση και θα μας πει η κυρία Κρυμπάτσκα που είναι η αρμόδια εισηγήτρια πώς προβλέπετε την προϋπόθεση αυτή, ε, την πρόταση αυτή και ως προϋπόθεση για την κοινωνική πρόοδο, τι προτάσεις θα ενσωματωθούν, τι πόροι μπορεί να προβλεφθούν. Για το Ταμείο Επενδύσεων, το Ταμείο Juncker, δεν προβλέπει τίποτε για τη μόρφωση, αν και κάνατε λόγο και για τις πλατφόρμες ε, e-learning ε, ηλεκτρονικής ε, εκμάθησης για τους διδάσκοντες, αλλά και για τη διευκόλυνση του ψηφιακού εξοπλισμού, του, του εξοπλισμού σε ηλεκτρονικό υλικό των σχολείων. Επίσης, θεωρώ ότι πρέπει να προχωρήσει αυτό γρήγορα και θα ήθελα να καταλάβω καλύτερα ποια είναι συγκεκριμένα η πρόταση για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα δίνει νόμιμα, θα επιτρέπει νόμιμα πρόσβαση στο υλικό σε ταινίε που έχουμε στο, στην Ευρώπη. Ναι, πρόεδρε, τελειώνω. τελειώνω. Για το ψηφιακό μέλλον. Αυτή η νέα στρατηγική για το ευρωπαϊκό έτος. Μα δεν είμαστε και τόσοι. Ίσως να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο καθένας να μιλήσει. Η πρόεδρος, ναι, όχι, δεν είμαστε και πολλοί, αλλά όπως είπα το πρωί, τα ίδια δικαιώματα για όλους. Αν περισσέψει χρόνος θα ξαναδώσουμε δυνατότητα. Νομίζω ότι αυτό είναι πιο δίκαιο. Η Επίτροπος παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κώστα. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Απάντω ευθύς αμέσως στην πρώτη για την προστασία των ανηλίκων. Ένας χρήστης μεταξύ των τριών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο αυτή τη στιγμή είναι νέος Άρα οι νέοι έρχονται πολύ γρήγορα σε επαφή και με τη θετική πλευρά του διαδικτύου, λογικό είναι να συμπεράνουμε ότι μπορεί να έρθουν πολύ γρήγορα σε επαφή και με τη σκοτεινή πλευρά του διαδικτύου. Και γι' αυτό στις 6 Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο ξεκινήσαμε μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία πληροφόρησης ε, Safer Internet for the EU, ασφαλέστερο διαδικτύο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνει το επόμενο έτος ένα έτος εκπαίδευσης στα ε, μέσα επικοινωνίας, έτος εκπαίδευσης προστασίας από τις κυβερνοεπιθέσεις και αυτή η εκστρατεία θέλει να θέσει στη διάθεση των πιο νέων εργαλεία που θα τους επιτρέψει να καταλάβουν πώς λειτουργεί το διαδίκτυο, σε ποιο θα απευθυνθούν όταν εκφοβίζονται, όταν παρενοχλούνται, όταν βλέπουν αρνητικές επιδράσεις και επιπτώσεις. Το σημαντικό είναι ότι αυτή η εκστρατεία πρέπει να γίνει μαζί με τους γονείς και με τους διδάσκοντες. Μόνο εάν κινητοποιηθούμε όλοι μαζί θα μπορέσουμε να ε, φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Έχουμε τα κέντρα για ασφαλέστερο διαδίκτυο που θα υπάρχουν σε όλα τα κράτη-μέλη που θα προβλέπουν δράσεις που θα είναι πολύ δραστήρια και ενεργητικά και θα προσπαθούν να διευρύνουν και να απευθύνονται σε όσο τον πιο ευρύ κοινό για να διαδώσουν απλές χειρονομίες. Πώς μπορεί κανείς να προστατεύσει τον κωδικό του, πώς μπορεί να μην πέσει θύμα του phishing, του ηλεκτρονικού ψαρέματος. Ε, ε, είναι απλά μέτρα που πρέπει να διαδοθούν περισσότερο και βασίζομαι σε εσάς. Ε, αυτό το κάλεσμα, αυτή την έκκληση, έκκληση και έχουμε και σημαντικούς πρέσβεις. Θέλουμε και εσείς το ίδιο να γίνετε. Ε, πρέσβεις και αγγελιοφόροι του μηνύματος ε, που κομίζει αυτή η εκστρατεία. Μόνο αν δουλέψουμε όλοι μαζί θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεύτερο, το σχέδιο δράσης για την εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή. Είναι πολύ θαρρυντικό το το ότι μπαίνει ένα τέλος σε αυτή τη δουλειά την μεμονωμένη. Πρέπει να δουλέψουμε μαζί στα μεταεκπαιδευτικά συστήματα. Είπαμε ξεκάθαρα ότι θέλουμε από τη μία μεριά η θέση των νέων γυναικών, των κοριτσιών να είναι ενισχυμένη, να έχουμε περισσότερες εκπαιδεύσεις και καταρτήσεις που οργανώνονται για τους εκπαιδευτικούς και τους διδάσκοντες. Πολύ συχνά λέγεται ότι οι νέοι δεν έχουν απαραίτητα τις ε, ψηφιακές διεξιότητες που χρειάζονται. Συχνά και οι εκπαιδευτικοί δεν τις έχουν. Μόνο το 25% των Ευρωπαίων εκπαιδευτικών έχουν δεξιότητες που να μπορούν να μεταδώσουν στους μαθητές τους και εμείς δουλεύουμε με τα Υπουργεία για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Εξτρατεία πληροφόρησης, πρόγραμμα selfie πολύ συγκεκριμένο. Δίνουμε τη δυνατότητα στα σχολεία να αυτοαξιολογηθούν σε ποιο επίπεδο βρίσκονται από την πλευρά της σύνθεσης με την ψηφιακή εποχή και ποιες είναι οι ε, ανάγκες τους. Σε μια πρώτη φάση 650 σχολεία συμμετείχαν στο πρόγραμμα Selfie και ε, στο δεύτερο εξάμεινο του 2018 θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση του προγράμματος. Είναι πολύ ενθαρρυντικό που μπορούμε να συνεργαστούμε με τα Υπουργεία Παιδείας των χωρών για να δούμε πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά τα μέτρα και πώς θα έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Χέλια Τρίπελ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Τους τελευταίους μήνες είχαμε πολλές ευκαιρίες να συζητήσουμε τα θέματα αυτά και στην τελική ανάλυση το ερώτημα που μας απασχολεί είναι πώς θα διαχειριστούμε αυτήν την ψηφιακή ε, επανάσταση. Σε όλους μας αρέσει το ότι έχουμε ε, πρόσβαση σε όλο αυτό το περιεχόμενο, ταινίες, σειρές κτλ. Από την άλλη μεριά έχουμε όμως τις ψευδείς ειδήσει, την παραπληροφόρηση ε, και για τους κινηματογραφιστές και, τον, και τους δημοσιογράφους του μέλλοντος είναι προφανές ότι χρειαζόμαστε ευφυείς ευφυή νομοθετήματα για να διέπεται το, το καθεστώς και το πλαίσιο. Ε, Μπορεί να μην άκουσα σωστά, αλλά θέλω να σας θέσω το εξή ερώτημα. Ε, ανακοινώσατε πριν από κάποιες εβδομάδες ε, ε, αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα. Θα ήθελα να μου πείτε ε, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σε σχέση με αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Κυρία Τρούπελ, σας ευχαριστώ για την πολύ επικοδομητική συνεργασία, γιατί συνεχώς δεχόμαστε ιδέες, προτάσεις, υποδείξεις και έτσι καταφέρνουμε να μιλούμε με μία και ενιαία φωνή και αυτό χρειάζονται οι πολίτες. Έρχομαι αμέσω στο ερώτημά σα, γιατί το ανέφερε και η κυρία Κώστα για το ευρωπαϊκό ρεπερτόριο, τον ευρωπαϊκό κατάλογο ευρωπαϊκών ταινιών. Ε, είναι δύο οι στόχοι μας να αυξήσουμε την ορατότητα των ευρωπαϊκών ταινιών, να γίνουν πιο ορατές στον κόσμο, γιατί είμαστε υπερήφανοι για την παραγωγή μας, να γίνουν πιο ορατές λοιπόν έτσι ώστε και οι νέοι μπορούν, να μπορέσουν να μάθουν ότι υπάρχουν τέτοιες ταινίε και άρα να τους δημιουργηθεί ανάγκη να τις δουν. Σε αυτό το ρεπερτόριο, σε αυτό το κατάλογο, όπως... Ε, ε, το έχουμε φανταστεί, ε, θα πρέπει να υπάρξουν δύο στάδια. Σε μία πρώτη φάση ε, θα εμπλέξουμε μόνο τους επαγγελματίες. Μία πλατφόρμα B2B, business to business, από επιχειρηματίες σε επιχειρηματίες. Δηλαδή να μπορούν οι επαγγελματίες του κλάδου να δουν ποιο ατενία είναι διαθέσιμη σε ποιο κράτος μέλος. Υπάρχει ήδη αυτή η ιδέα. Στο Βερολίνο οργάνωσα την πρώτη συζήτηση στρογγυλή τραπέζη. Δύο άλλε ιδέε είναι αυτή τη στιγμή ε, υπό επεξεργασία. Πρέπει να δουλέψουμε το branding, το κομμάτι της μάρκας, του σήματο και να έχουμε και μια πολιτική για τα editorial. Ε, δηλαδή στήριξη από την αρχισυνταξία για να, μπορούμε, να, μπορεί να υπάρχει επιθυμία να ειδωθούν αυτές οι ταινίε. Ένα δεύτερο κομμάτι που έχουμε προβλέψει, η δεύτερη φάση θα είναι πολύ πιο μακροχρόνια. Είναι να πάμε προς μια πλατφόρμα B2C, από business to consumer δηλαδή. Ε, δηλαδή να έχει ο Ευρωπαίος πολίτης ένα εργαλείο, να μπαίνει σε αυτή την πλατφόρμα και να μάθει πού μπορεί να δει νόμιμα τη συγκεκριμένη ταινία. Σε ποια επικράτεια θα είναι σε άμεση μετάδοση ζωντανή ή θα είναι σε λήψη ε, κατέβασμα ε, με βίντεο on demand. Επομένως, Πολύ γρήγορα μπορεί να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση που αφορά μόνο τους επαγγελματίες του κλάδου. Θέλουμε αυτό να το εγκαινιάσουμε τον Οκτώβριο του 2018 και να ξεκινήσει η λειτουργία την επόμενη χρονιά. Όμως, Τη δεύτερη φάση θα χρειαστεί πολύ περισσότερους χρόνους για να δούμε τις ιδιαιτερότητες και τα επιμέρους συμφέροντα. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Προχωρούμε. Μετά τους συντονιστές, τους λοιπούς συναδέλφους. Κύριος Φίσας, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για το απατητικό αυτό πρόγραμμα. Δεν περίμενα και τίποτα λιγότερα βέβαια, γιατί σας γνωρίζω. Τα εξή έχω να υπογραμμίσω. Καταρχάς, ψηφιακό περιεχόμενο για τους ηλικιωμένου. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό βεβαίως και για τους νέους που είναι στο σχολείο, του που έχουν τελειώσει το σχολείο. Υπάρχουν και ηλικιωμένοι οι οποίοι είναι αναλφάβητοι. Επομένως, τι μπορούμε να κάνουμε για αυτούς. Ε, λαμβάνουν ε, όλο και περισσότερο επίσημα έγγραφα με ψηφιακή μορφή. Έχετε κάποια λύση να προτείνετε. Και δεύτερον, για να ολοκληρώσω, ξέρω ότι είναι νωρί να συζητούμε για fake news, αλλά μπορείτε να μα δώσετε κάποιε ιδέε για το πώ θα μπορούσαμε αυτό το καρκίνωμα ε, που μα μαστίζει να το αντιμετωπίσουμε από το ψηφιακό περιεχόμενο. Παρακαλώ, κυρία Καμπριέλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φίσας για τις πολύ εύστοχες αυτές ερωτήσεις. Για την πρώτη, που είναι πολύ δύσκολη βέβαια, πρέπει να ξέρουμε πότε χρειάζεται να γίνει κάτι περισσότερο από ό,τι έχουμε προβλέψει. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε θαυματουργές λύσεις. Όταν μιλούμε για τους ηλικιωμένους πρέπει πάντα να στακόμαστε στο ότι υπάρχουν διάφορες κατηγορίες. Αυτοί που έχουν ε, την ε, επιθυμία να ακολουθήσουν μια επιμόρφωση στο ψηφιακό περιεχόμενο και εκείνοι που δεν έχουν τέτοια επιθυμία. Μέχρι τώρα βέβαια δεν έχουμε κάνει τίποτα. Έχουμε μια δομή που επιτρέπει στους ηλικιωμένου να αποκτήσουν ε, την ψηφιακή επιμόρφωση, το Upskilling Pathways, είναι αυτό το πρόγραμμα με την Επιτροπή Τίσεντ έχουμε αναπτύξει ε, για εκείνους που θέλουν να συνεχίσουν ε, να αποκτούν προσθέτες δεξιότητες στο ψηφιακό περιεχόμενο. Από την άλλη θα πρέπει να συστήσουμε και άλλες λύσεις. Μία από αυτές είναι στα Digital Innovation Hubs στους ε, κόμβους ψηφιακής σε ένα πρόγραμμα για, τα πέντε, για πέντε χρόνια γιατί που τρέχει ήδη το δεύτερο του έτος, έχει άλλα τρία και προβλέπει 900 εκατομμύρια ευρώ μας επιτρέπει να εξασφαλίσουμε έναν κόμβο ψηφιακής καινοτομία σε κάθε περιφέρεια. Αυτό ε, λοιπόν ενσωματώνει και την πρότασή μου για ένα τμήμα επιμόρφωση των κάθε από αυτού του κόμβου. Εάν μπορέσουμε να το αναπτύξουμε σε επίπεδο περιφέρεια, όχι μακριά από το σπίτι του καθενό, γιατί ξέρουμε ότι για του ηλικιωμένου οι αποστάσει, η κινητικότητα δεν έχουν την ίδια έννοια με αυτό που μπορεί να εννοεί κάποιο νέο. Αυτό είναι μια λύση λοιπόν, αλλά βεβαίω πρέπει να συνεχίσουμε να αναζητούμε περισσότερε λύσει. Και τότε ναι, ίσως και τα κράτη-μέλη να μην δείξουν ε, τέτοια διάθεση να διαφυλάξουν ζηλότυπα τι αρμοδιότητέ του και να επιτρέψουν να αναπτυχθεί η δραστηριότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάτι ακόμη που θέλω να τονίσω ότι μας έχει επιτρέψει αυτή τη δράση η Συμμαχία για την ψηφιακή απασχόληση και τις δεξιότητες 3,5 εκατομμύρια ε, επιμορφώσεων, επιμορφωτικών προγραμμάτων. βεβαίω με περισσότερη αστίαση στους νέου μα έχει επιτρέψει αυτή η συμμαχία, αλλά ταυτόχρονα βλέπω ότι όλο και περισσότεροι δίνουν ε, την διάσταση των πιο ευάλωτων και των ηλικιωμένων. Όχι μόνο στου νέου δηλαδή να δίνουμε έμφαση, γιατί αυτή τη στιγμή ο ψηφιακός αναλφαβητισμός ε, συνιστά και κίνδυνο για αποκλεισμό, για δυναμία συνεργασίας, συμμετοχή στην κοινωνία κτλ για τα fake news και θα ήθελα αμέσω να κάνω τη διαφοροποίηση μεταξύ των fake news και του παράνομου περιεχομένου που επίση αναφέρθηκε. Εμείς για το παράνομο περιεχόμενο έχουμε μια σαφή, ένα σαφή ορισμό στο ευρωπαϊκό δίκαιο που είναι η, το λαθρεμπόριο, η παιδική πορνογραφία, η ρητορική του μίσους, όλα αυτά. Τώρα για τα fake news, για τις ψευδείς ειδήσει έχουμε ανάγκη για ορισμό. Έχουμε θεσπίσει μια σειρά από ομάδες και των οποίων μία ομάδα εργασίας επεξεργάζεται τον ορισμό και θα σας πω ότι εκεί πέρα ακριβώς είναι και οι πιο ζωντανές ε, συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα. Έχουμε τρεις ομάδες συντακτικέ με τους ειδικού ε, για το θέμα της νομοθεσίας που ακόμη δεν έχει προχωρήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να κοιτάξουμε τι εννοούμε ως fake news. Fake news δεν είναι ούτε τα ειρωνικά σχόλια, ούτε οι σχολιασμοί. Εδώ έχουμε να κάνουμε περισσότερο με την προσπάθεια να παραπλανηθεί ο πολίτης μέσω διαφημιστικών ε, αλλά και άλλων πολιτικών μηνυμάτων. Αυτή τη στιγμή δουλεύει, όπως είπα, η ομάδα εργασίας, επεξεργάζεται τις προτάσεις για ένα ε, ορισμό στα fake news. Τέσσερα είναι τα σημεία κλειδιά που θα πρέπει να μας καθοδηγήσουν. Αφενός, περιεκτικότητα. Πρέπει όλοι να κάνουμε τη δουλειά μας. Ευθύνη έχουν και οι κοινωνικές, τα κοινωνικά δίκτυα, οι πλατφόρμες, ε, τα μέσα, οι υπηρεσίες για τους νέους, η κοινωνία των πολιτών, τα θεσμικά όργανα. Όλοι έχουν δουλειά να κάνουν στην αντιμετώπιση των fake news. Δεύτερον, η διαφάνεια θα πρέπει να γνωρίζουμε περισσότερα για τους μηχανισμούς που αξιοποιούνται για την διάδοση των ψευδών ειδήσεων, οικονομικές ροές, εισόδημα το οποίο προέρχεται από την ε, διασπορά αυτών των ψευδών ειδήσεων, ευαισθητοποίηση του πολίτη επίσης με τα και ε, δυνατότητες που θα του προσφέρουμε με εργαλεία κατάλληλα. Αλλά το θέμα είναι δεν θα αποφασίζει κανείς για κάποιον άλλον. Θα πρέπει αυτή η ελευθερία να διαφυλακθεί. Αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να ενισχύσουμε το fact-checking, την επαλήθευση των ειδήσεων, των γεγονότων. Και τέλει, η ποικιλία, η ποικιλομορφία. Δεν μπορούμε να καταργήσουμε, δεν μπορούμε να απαλείψουμε τις ψευδείς ειδήσει. Γιατί όμως να μην δώσουμε περισσότερη έμφαση σε ένα ποιοτικό περιεχόμενο, το οποίο κάποια στιγμή θα ε, αποδιαρθρώσει τον χώρο τον οποίο έχουν μπορέσει να καταλάβουν οι ψευδείς ειδήσει. Αυτή είναι η δουλειά εν εξελίξη. Μέσα Μαρτίου θα δημοσιευθεί η σχετική έκθεση. 27 ε, Φεβρουαρίου πάλι έχω μία δημόσια συζήτηση προβλέψη, για να μπορέσουν να λάβουν το λόγο όσοι δεν είχαν μέχρι τώρα την ευκαιρία να τοποθετηθούν. Πρέπει να συνεχιστεί αυτή η δουλειά, πιστεύω, να ακούγονται οι διαφορές απόψεις και να εισακούγονται για να μπορέσουμε να καταλήξουμε και ιδιαίτερα θέλω να επαναλάβω κάτι που είπα και στους ειδικού στην ομάδα των ειδικών. Θέλω κάτι το καινούριο και κάτι το συγκεκριμένο. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Λιμπάτσικα, ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα αυτή. Όχι, η διερμηνία είναι εντάξει, μπορούμε να συνεχίσουμε. Entschuldigung, Martina, ich kann nicht... Όχι, Ματίνα, όταν κάποιο θέλει να λάβει το λόγο ω συντονιστή, πρέπει να με έχει ενημερώσει εγκαίρω, έτσι. Κριστίνα, εσύ. Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε. Τρία ζητήματα θέλω να γύρω και επιτρέψτε μου να επανέλθω στο ζήτημα της ε, απουσίας της έλλειψης ψηφιακών δεξιοτήτων σε παιδό δασκάλων, διδασκόντων. Πολλές φορές οι μαθητές ξέρουν περισσότερα για τη χρήση του ψηφιακού περιεχομένου από ότι οι δάσκαλοι τους. Στους διδάσκοντες όμως σε πανεπιστημιακό επίπεδο θα πρέπει να ενισχυθεί και αυτό μέσα από τις, από τις σχολές για να ενισχυθεί να ενισχυθούν οι ψηφιακές δεξιότητες των διδασκόντων του εκπαιδευτικού προσωπικού. Επίσης, κύριε Επίτροπε, στη χώρα μου εγώ οργανώνω ε, μαθήματα για τους ηλικιωμένους συμπολίτε μου για το ψηφιακό περιεχόμενο και πρέπει να σας πω ότι έχω τέτοια ζήτηση που δεν είμαι στη θέση να ικανοποιήσω όλες τις αιτήσει. Βεβαίως, μέσα από οργανώσεις, μέσα από ε, ενώσεις προσώπων συμμετέχουν οι ηλικιωμένοι, ενώσεις προσώπων και οργανώσεις που θα μπορούσαν, εάν εξασφαλίσουν τη σχετική χρηματοδότηση από τις τοπικές κυβερνήσεις, να βοηθήσουν σε αυτό το έργο της επιμόρφωσης. Πώς μπορούμε εντωμεταξύ να εξασφαλίσουμε την αξιολόγηση της ποιότητας, τρίτη ερώτηση, της εκπαίδευσης και τέταρτο, Θεωρείτε ότι πρέπει οι τεχνικές ε, λύσεις που προσφέρονται να είναι και προσαρμοσμένες στην ηλικία του χρήστη. Η πρόεδρο. ευχαριστώ πολύ. Αν θέλετε και εσείς κάπως σύντομα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λιμπάτσκα. Ναι, για τις ψηφιακές ε, δεξιότητες των διδασκόντων στηρίζω κάθε ιδέα που θα επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς να είναι καλύτερα ενημερωμένοι, να διαθέτουν ένα δίκτυο, γιατί αυτό είναι κάτι που αφορά και τους ενήλικες. Σε τοπικό επίπεδο μπορεί να υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες. Έχει έρθει η ώρα, χάρη στις νέες τεχνολογίες, να υπάρξει δίκτυο να συνδέονται καλύτερα οι μεν με τους δε, να υπάρχουν διαδικτυακές τοποθεσίες, εργαλεία εκπαιδευτικά διαδικτυακά, εργαλεία εκπαιδευτικής κατάρτισης διαδικτυακής. Θέλω να στηρίξω όλες αυτές τις πρωτοβουλίες. Τώρα, για μια ποιοτική εκπαίδευση. Δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα, δεν είναι δικό μου χαρτοφυλάκιο η εκπαίδευση παραμένει στην εθνική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Όμως, χάρη στη ψηφιακή εποχή, μπορούμε να δημιουργήσουμε περισσότερες συνέργειες και γι' αυτό θα στηρίξουν πρωτοβουλίες. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα. Να μια πολύ ωραία πρωτοβουλία που επιτρέπει σε ένα εκατομμύριο ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη για τρεις εβδομάδες τον Οκτώβριο μήνα να δουν θέματα κώδικα και προγραμματισμού, να καταλάβουν ότι μπορούμε να είμαστε όχι μόνο χρήστες περιεχομένου, αλλά και δημιουργοί περιεχομένου ψηφιακού. Το ίδιο και για την εβδομάδα επαγγελματικής κατάρτισης. Φέτος, τον Νοέμβριο, για δεύτερη συνεχή χρονιά, οργανώθηκε αυτή η εβδομάδα και χαιρετίζω τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, γιατί η ποιοτική εκπαίδευση για μένα είναι ποιοτική όταν συνδέεται ακριβώς με αυτό στο οποίο στοχεύει στην αγορά εργασίας. Γνωρίζουμε σήμερα ότι έχουμε ανάγκη νέους που να είναι εκπαιδευμένοι και τα προσόντα τους να αντιστοιχούν σε αυτό που ζητάει η αγορά εργασίας. Έχουμε αυτή τη στιγμή 350.000 ειδικού σε θέματα τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών. Το 2020 αυτή θα είναι πάνω από 500.000. Ο κόσμος των πανεπιστημίων και ο κόσμος των επιχειρήσεων πρέπει να συνεργαστούν περισσότερο. Και εγώ θα συμβάλλω προς αυτή την κατεύθυνση, στο βαθμό που μου αναλογεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε η κυρία Μίχελ. Ευχαριστώ και συγγνώμη. Θεώρησα δεδομένο ότι θα κάνουμε έναν κύκλο τοποθετήσεων για όλες τις πολιτικές ομάδες στην αρχή. Γι' αυτό, συγγνώμη, μπερδεύτηκα ίσως, ε, δεν ήθελα να διακόψω τη ροή της συζήτησης. Κυρία Επίτροπε, σας συγχαίρω ε, για την ιδέα που παρουσιάσατε στο, στην Περλινάλε. Ως Βερολινέζα βεβαίω ενημερώθηκα σχετικά με αυτήν την ευρωπαϊκή online πλατφόρμα ταινιών. Εμένα θα με ενδιέφερε ποιος, κατά πόσο θα είναι δημόσιος ή εμπορικός ο χαρακτήρας αυτού του project. Πώς θέλετε επίσης να πείσετε την, τον, ε, την ευρωπαϊκή κινηματογραφική βιομηχανία που έχει τις ανησυχίες της όσον αφορά την, ε, τις, ε, τα, ζητήματα των, των δικαιωμάτων στις διάφορες επικράτειες. Επίσης, για τα αρχεία, της βιβλιοθήκες, τα, τα μουσεία που βρίσκονται ε, σε μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με την ψηφιοποίηση του υλικού τους. Ε, έχετε συγκεκριμένες προτάσεις, σκοπεύετε να προχωρήσετε σε κάποιον συγκεκριμένο διάλογο ως προς αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Πίτροπος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις αυτές για το Ευρωπαϊκό Κατάλογο Ρεπερτόριο Ευρωπαϊκών Ταινιών. Δεν έχουμε φτάσει στην εμπορική φάση. Πόρο απέχουμε. Το σημαντικό είναι να έχουμε ένα χώρο ενιαίο, μοναδικό, γιατί τώρα υπάρχουν ένα σωρό πλατφόρμες video on demand, παρόλο που υπάρχουν καλές εμπειρίες και καλά διδάγματα. Σκοπός είναι να υπάρχει ένας ενιαίος χώρος όπου αυτό γιατί η πολιτιστική κληρονομιά, όλα αυτά τα προϊόντα πολιτιστικής κληρονομιάς να μπορούν να αντιπροσωπεύονται εκεί και να μπορούμε να βλέπουμε ποια ευρωπαϊκή ταινία διατίθεται και πού. Τέτοιου είδους ε, κατάλογος, ρεπερτόριο υπάρχει σε ορισμένα κρατημέλη και λειτουργεί πολύ καλά. Θα πρότεινα λοιπόν το ίδιο να πράξουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά για την πρώτη φάση. Τώρα για τη δεύτερη φάση. Είμαι πολύ ανοιχτή στη συζήτηση. Δεν θέλω να έρθω και να επιβάλλω τις ιδέες μου. Θέλω για τη δεύτερη φάση να μάθω ακριβώς τι πιστεύει ο καθένα. Και βεβαίως υπάρχουν συγγραφικά δικαιώματα, συμβάσει και συμβόλαια που υπογράφονται. Και εγώ θέλω να ε, σεβαστούμε ε, όλα αυτά. Στην Περλινάλε είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση στρογγυλής τραπέζης. Θα έχουμε ανανεώσει το ραντεβού μα για δύο μήνε αργότερα, όπου θα είναι πολύ πιο τεχνική η συζήτηση. Στο Φεστιβάλ των Κατών θα οργανώσουμε και μια άλλη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης και ελπίζουμε τον Οκτώβριο να μπορέσουμε να ε, παρουσιάσουμε την πρώτη μακέτα, να το πω έτσι, το πρώτο πρωτότυπο ε, αυτού του έργου. Τώρα για τα συγγραφικά δικαιώματα, τα δικαιώματα του δημιουργού ε, για θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, ε, το, η μπάλα βρίσκεται από την πλευρά του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ την Επιτροπή Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εσείς τη δουλειά σας την έχετε κάνει. Περιμένουμε να ψηφιστεί το τελικό κείμενο στα τέλη Μαρτίου ή στον τον Απρίλιο για να περάσουμε και στα σημαντικά για να μην χαθεί η φιλοδοξία της πρότασης. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει. Ευχαριστούμε. Κύριε Στογεύσκη. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας πω ότι όταν παρουσιάσω την έκθεσή μου ε, για, την, ε, για τα οικονομικά και άλλα εμπόδια που εμποδίζουν την πρόσβαση στον πολιτισμό, θα ήθελα να σας καλέσω να παραστείτε, κυρία Επίτροπε, για να ακούσετε τα ευρήματά μας. Ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα για ε, το τι έχει να, για ό,τι έχει να κάνει με τη συμμετοχή σε προϊόντα πολιτισμού στο διαδίκτυο. Και εσείς το είπατε ότι δεν ξέρουμε πού διατίθενται διαδικτυακά ευρωπαϊκές ταινίε και πού δεν διατίθενται. Θα ήθελα να σας καλέσω να διευρύνετε την έρευνα της ε, Ευρωστάτ, της Eurostat έτσι ώστε οι πολιτικές μας να χαράσσονται καλύτερα σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόσβαση στον πολιτισμό. Κατά τη διάρκεια της Πλωνικής Προεδρίας, εγώ ήμουν υπουργό Πολιτισμού και συνειδητοποίησα τότε πόσες πολλές ευρωπαϊκές ταινίε δεν είναι προσβάσιμες, δεν είναι διαθέσιμες, διότι υπάρχουν προβλήματα με το copyright, με τα πνευματικά δικαιώματα και θα ήθελα να διευρυθούν αυτές οι προτάσεις και έτσι να μην μπλοκάρονται ε, τα ε, προϊόντα ευρωπαϊκού πολιτισμού λόγω αυτών των επιχειρηματικών και εμπορικών συγκρούσεων. Ευχαριστώ. Η, πρόεδρο, η Επίτροπος, σας ευχαριστώ και εγώ. Σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία που έχετε αναλάβει. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ακριβώς ε, σαφή εικόνα για το ποια είναι τα εμπόδια της πρόσβασης στον πολιτισμό, οικονομικά ή άλλα, και βεβαίω δέχομαι την πρόσκλησή σας. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέκαθεν είναι συνομιλητής πρώτης γραμμής για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι κάτι το οποίο προσυπογράφω 100% και πρέπει να δούμε ποια είναι τα μέτρα τα ιδανικά. Να έχουμε πιλωτικά προγράμματα, να υιοθετήσουμε άλλου είδου μέτρα για να προωθήσουμε ακριβώς αυτές τις ε, επιδιώξεις οι οποίες με βρίσκουν απολύτως σύμφωνοι. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριος Νίκοφ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γκαβριέλ, 40% του ευρωπαϊκού πληθυσμού δεν διαθέτει ψηφιακές δεξιότητες. Επαρκείς τουλάχιστον. 20% μάλιστα δεν έχει καθόλου ψηφιακές δεξιότητες. Η Βουλγαρία βρίσκεται στην ε, πρώτη τελευταία θέση. Ε, ένα πολύ μικρό μέρος του πληθυσμού μόλις της Βουλγαρίας έχει ψηφιακέ δεξιότητε. Και αυτό αποτελεί φραγμό για την πρόσβαση και στον πολιτισμό. Εμείς εδώ χαράσουμε στρατηγικές, τις υλοποιούμε, όμως δεν λαμβάνουμε υπόψη πόσο μεγάλη απόσταση τελικά υπάρχει ανάμεσα στις στρατηγικές αυτές και, τον, και τους πολίτες λόγω της έλλειψης ψηφιακών δεξιοτήτων. Υπάρχουν προσπάθειες ε, διάδοσης ε, των ψηφιακών δεξιοτήτων σε εθνικό επίπεδο και μάλιστα είχαν καταρριφθεί σχετικά σχέδια ως τα μέσα του 2017. Δεύτερο θέμα. Αναφερθήκατε στην ψηφιακή εκπαίδευση. Προβλέπονται συγκεκριμένα μέτρα για τις ε, χώρες στις οποίες υπάρχει ε, όπου ο πληθυσμό τέλο πάντων είναι ε, διασπαρμένο σε όλη την επικράτεια. Πράγματι, λέει η Επιτροπό, τα αριθμητικά αυτά στοιχεία είναι ανησυχητικά και έχετε απόλυτο δίκιο που μα επιστάτε την προσοχή στο γεγονό αυτό και γι' αυτό δίνουμε έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες, στα ψηφιακά προσόντα. Μπορεί να έχουμε καταπληκτικά οικονομικά εργαλεία, χρηματοδοτικές στρατηγικές και ό,τι να είναι. Αν δεν αναβαθμίσουμε όμως τα ψηφιακά προσόντα των πολιτών μας, δεν θα δρέψουμε ποτέ τα ωφέλη της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή. Ξέρουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν εθνικές στρατηγικές το θέμα όμως δεν είναι να έχει κανείς ε, μια στρατηγική, δεν είναι μόνο αυτό το θέμα, αλλά πώς εφαρμόζεται και ποια πρόοδο σημειώνεται. Προσπαθούμε να δείξουμε την προσθεθέμενη αξία που έχει η δική μας συνεισφορά στις εθνικές στρατηγικές. Μπορώ να σας δώσω το παράδειγμα της εβδομάδας για την Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Κατάρτιση και άλλα παραδείγματα για ένα σωρό πρωτοβουλίε που δείχνουν πόσο σημαντικά είναι τα ψηφιακά προσόντα και δεξιότητες. Θα ήθελα όμως να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι τα κράτη-μέλη επιμένουν στο τη διατήρηση των αρμοδιοτήτων τους και θέλουν να εργαστούν σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, οι νέες τεχνολογίες προχωρούν, εξελίσσονται και ίσως πρέπει να αλλάξουμε την προσέγγισή μας. Ε, θέσατε το ερώτημα για τους διδάσκοντες και καθηγητές στις περιοχές που υπάρχει πολύ αραιή κατανομή του πληθυσμού. Θα έλεγα ότι όταν υιοθετούμε προγράμματα και μέτρα σε ε, κοινοτικό επίπεδο, πρέπει πρώτα να υπάρξει πρόσβαση στο διαδίκτυο σε αυτές τις περιφέρειες, τις αραιοκατοικημένες για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στο οτιδήποτε. Ας δώσουμε πρώτα πρόσβαση στο διαδίκτυο για να μπορούμε να μιλάμε μετά. 76% των νοικοκυριών στις αστικές περιοχές έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ενώ στην Ήπεθρο και στις αεροκατοικημένες περιοχές πρόσβαση στο διαδίκτυο έχουν λιγότερο από το 40% των νοικοκυριών. Αυτό πρέπει να είναι το σημείο κίνησής μας. Και αυτή είναι η βασική συνιστόσα του σχεδίου μας και η βασική πρόκληση είναι να εφαρμοστεί στην πράξη. Να υλοποιηθεί δηλαδή. Υπ' αυτή την έννοια θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και τους πόρους που χρειάζεται να κατανεμηθούν στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Φλάνακαν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είμαι μέλος Επιτροπής και γι' αυτό ευχαριστώ που μου επιτρέπετε να λάβω το λόγο. Νομίζω ότι οι, πρόεδρος, οι πρόεδροι των άλλων επιτροπών στις οποίες συμμετέχω έχουν πολλά να μάθουν από εσά. Για την ομάδα αυτή των εμπειρογνωμόνων, κυρία Γκάμπριελ, για τα fake news, για τις ψευδείς ειδήσει, μιλήσατε για διαφάνεια, μιλήσατε για αξιοπιστία, καλή επικοινωνία, περι... επικοινωνίας υγιές. Όταν ε, οι Ιρλανδοί από εκπρόσωπο αυτής της ομάδας υψηλού επίπεδου για τα fake news έμαθαν ότι υπάρχει αυτή η ομάδα, άρχισαν αμέσως να μου γράφουν ε, τι πρόκειται εγώ να κάνω για να αντιμετωπίσω αυτό το φαινόμενο. Και ξέρετε ότι αισθάνθηκαν, ε, ανατρίχιασαν όπως και εγώ άλλωστε, γιατί ξέρουν ποιος είναι αυτός, από ποια εφημερίδα προέρχεται, από εφημερίδα ακριβώς που έχει απολύσει δημοσιογράφους επειδή έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Και γι' αυτό το λόγο σας έστειλε επιστολή 16 Ιανουαρίου, πριν από ένα μήνα. Μιλάτε για περιβάλλον ε, καλό περιβάλλον επικοινωνία. Γιατί δεν μου απαντήσατε. 25 Ιανουαρίου σας στέλνω email. Πάλι δεν έχω λάβει απάντηση. Εγώ αυτό που ζητώ είναι για μένα και τον εν λόγω δημοσιογράφο να έχουμε την ευκαιρία να κάτσουμε μαζί σας και να εξηγήσουμε γιατί ήταν τόσο κακή η ιδέα να επιλέξετε τον Steven Ray από την Independent News Media ή Media. Μιλάτε για πολυμορφία, αλλά πολυμορφία δεν υπάρχει. Ναι, ναι, σταμάτω πρόεδρε, ευχαριστώ. Νομίζω ότι έχει περάσει το μήνυμα επαρκώς. Κυρία Γκαμπριέλα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Φλάναγκαν. Μια απόφαση, μια απάντηση απεστάλλει εξ ονόματος της Γενικής Διεύθυνσης. Την είδα εγώ. Και στην απάντηση αυτή λεγόταν αυτό που και εγώ θα σας είχα πει και προσωπικά και τώρα σας το λέω που σας ε, κοιτώ ενωπία, Δεν γίνονται επιλογές με προσωπικούς όρους. Θα αντιλάβετε την επιστολή, ναι. Πάντως αυτό που λέμε στην, στην επιστολή είναι ότι η επιλογή γίνεται με τη βάση κάποιων ανεξάρτητων κριτηρίων. Πραγματογνωμοσύνη υπήρξε, γεωγραφική ισορροπία ε, επίσης, όπως και ε, ισότιμη κατανομή μεταξύ των φύλων. 350 υποψηφιότητε, λάβαμε σε ένα μήνα. Οι εμπειρογνώμονε που επιλέξαμε είναι συνολικά 39 παραμένω στη διαθεσή σας για να συναντηθούμε, αν θέλετε πολύ σύντομα να κλείσουμε ένα ραντεβού για να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάλινοφ. Δεν θα χάσω χρόνο στις ε, ευρωφροσύνες. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Τρεις ερωτήσεις. Περισσότερο μια σύσταση μάλλον ή μια πρόταση για πολιτική. Ξέρετε, φαντάζομαι ότι ο τομέας ε, της, ε, πληροφ... της κοινωνίας πληροφορίας έχει θεσπίσει ένα δίκτυο πολύ αποτελεσματικό για, τα, ε, για τις ψηφιακές δεξιότητες για τους νέους. Μπορούμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε το δυναμικό αυτό μέχρι ότου αναπτυχθούν τα αντίστοιχα συστήματα των κρατών μελών, τα εκπαιδευτικά. Είναι τόσο καλό εστιασμένο και ίσως και να αξιοποιηθεί πολύ σύντομα σε όρους ιδιωτικής ε, λειτουργίας. Νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα λοιπόν. Το δέχεστε να το ενσωματώσουμε. Ε, δεύτερη ερώτηση, προστασία των ανελίκων, που θα συστήσουμε ειδικότερα αύριο. Πολλές όμως οικογένειες και παιδιά ιδιαίτερα μεγαλώνουν χωρίς πατέρα και μητέρα που ζουν στο εξωτερικό, τα έχουν εγκαταλείψει, τα έχουν αφήσει μάλλον να μεγαλώνουν με τους παππούδες. Πρέπει και οι παππούδες και οι γιαγιάδες να μάθουν πώς να χειρίζονται το διαδίκτυο και πώς να προστατεύουν τα παιδιά από τους κινδύνους του διαδικτύου. Είναι πολλή η δουλειά που έχουμε να κάνουμε ακόμα. Και τρίτη ερώτηση. Για τα fake news, ψευδείς ειδήσει και απαντήστε σε όποια θέλετε και σε όποιον θέλετε. Θα υπάρξουν ευρωεκλογέ το 2019. Ας επικεντρωθούμε στον αγώνα κατά των ψευδών ειδήσεων, κυρίω σε σχέση με τις ευρωεκλογέ του 2019. Ας μην δαπανίσουμε πόρους τόσο στις μακροπρόθεσμες στρατηγικές. Α τα αφήσουμε για την προσεχή ε, επιτροπή. Ξέρω ότι εσείς δεν μπορείτε αυτό να το πείτε δημοσία, εγώ όμως μπορώ να το υποδείξω. Ας επικεντρωθούμε λοιπόν σε αυτή τη διάδοση ψευδών ειδήσεων που θα επιδιώξει την ε, διάβρωση του αποτελέσματος των ευρωεκλογών. Γιατί αν τα καταφέρουμε τότε θα έχουμε και τα καλύτερα αποτελέσματα από τις ευρωεκλογέ στην ιστορία του αν είμαστε επιτυχείς βέβαια σε αυτό. Η κυρία Γκάμπριελ, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαλινόφ. Και οι τρεις ερωτήσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές. Πρώτον, Πράγματι θα ήταν καλύτερο να έχουμε ευρύτερη συνεργασία. Και αυτό ήδη συμβαίνει σε ορισμένα κράτη-μέλη, διότι υπάρχουν εθνικοί συνασπισμοί, εθνικές συμμαχίες για ψηφιακές θέσεις απασχόλησης. Η δική μας συμμαχία απαρτίζεται από 19 εθνικές συμμαχίες. Θα ήταν καλό για κάθε χώρα μέλος να έχει μια εθνική συμμαχία. Στις αιτήσεις συναντήσεις ή τον Ιούνιο κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής για την ψηφιακή εποχή στη Βολγαρία είναι το κατάλληλο πλαίσιο για να συζητηθεί αυτή η ιδέα. Και ενδεχομένως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και μια ξεχωριστή συνεδρία για το θέμα αυτό. Τώρα για τα παιδιά των οποίων οι γονείς εργάζονται στο εξωτερικό. Δεν έχουμε ασχοληθεί με αυτό το θέμα μέχρι σήμερα, αλλά είναι πολύ σημαντικό σε ορισμένες ε, χώρες μέλη. Είμαστε ανοιχτοί ε, ε, σε όλες τις, ιδέες, τις νέες ιδέες. Τώρα, ψευδείς ειδήσει και επόμενες ευρωεκλογές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μία από τις διαστάσεις που πραγματικά θα ενσωματώσουμε και είναι ένα θέμα που θα αντιμετωπιστεί και από την ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επίπεδου. Αυτό το μήνυμα προσπαθώ να περάσω και στους εμπειρογνώμονες. Έχουμε μακροπρόθεσμα μέτρα και έχουμε ένα κάποιο επίπεδο αλφαβητισμού στα ΜΜΕ. Ο αλφαβητισμός, ο μηντιακός θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο ε, την επόμενη δεκαετία. Χρειαζόμαστε όμως και βραχυπρόθεσμα μέτρα. Και για αυτά τα βραχυπρόθεσμα μέτρα, ο ορίζοντα μέχρι τι επόμενε ευρωεκλογέ θα είναι προτεραιότητα και η έκθεση θα είναι δημόσια και θα λάβουμε υπόψη όλε τι γνωμοδοτήσει, όλε τι απόψει πριν από τη δημοσίευση τη ανακοίνωσή μα που προγραμματίζεται για τον Απρίλιο. Περιμένω δύο λεπτάκια γιατί ξέρω ότι στα γερμανικά με θα τελειώσει η πρόταση από τη διερμηνία. χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα. Κυρία Ward, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να σας ρωτήσω πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε την περιέργεια, την πολιτιστική κυρίως περιέργεια για όλους αυτούς που είναι σε διαδικασίες μάθησης και κυρίως ε, δεδομένου ότι προάγονται χάρη σε αλγορίθμους ε, πολιτιστικά περιεχόμενα τα οποία είναι μόνο ε, τα τρέχοντα, μόνο τα mainstream. Υπάρχει δυνατότητα για μια στρατηγική για την ψηφιακή επιμόρφωση αλλά και την επιμόρφωση σε σχέση με τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό νομίζω εντάσσεται σε όσα συζητούμε σήμερα. Και επίσης θέλω να προτείνω Η επιμόρφωση σχέση με τις δυνατότητες για απασχόληση νομίζω θα μας ε, απασχολήσει στο μέλλον. Ε, θα έχουμε πολύ χρόνο στη, στα χέρια μας στο μέλλον ε, χάρη στην τεχνολογία αυτή της πληροφορίας και δεν θα ξέρουμε τι θα τον κάνουμε. Πολλοί δεν έχουν λοιπόν δυνατότητες να αναζητήσουν κάποια δημιουργική απασχόληση και θα πρέπει να τους ενισχύσουμε. Επίσης, STEM και όχι STEAM. Το A στα αρχικά αυτά σημαίνει arts, τέχνες. Μην μιλάμε μόνο για μαθηματικά, μην μιλάμε μόνο για τεχνολογία. Να μιλούμε και για τέχνες και δημιουργικότητα. Κάτι ακόμη, σήμερα ήταν κάποιος από το δικό σας επιτελείο στο πρόγευμα της IF και έμαθα από ό,τι είπε δηλαδή ότι ενδιαφέρεστε ιδιαίτερα για τα προγράμματα που βρίσκονται στη βάση, στις τοπικές κοινωνίες. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Ως προς την πρώτη ερώτηση για το πώς θα ενισχύσουμε το ενδιαφέρον. Πιστεύω ότι είμαστε αρκετά φιλόδοξοι, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε φιλόδοξοι γιατί έχουμε κάποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες και κάποιες άλλες που δεν είναι νομοθετικές. Έχουμε την οδηγία SMA. Και μέρος της διαπραγμάτευσης είχε να κάνει με το ποσοστό των ευρωπαϊκών έργων που υποχρεούνται οι πλατφόρμες να κυκλοφορήσουν και να διαθέσουν χώρο για αυτά. Είναι μια νέα πρόταση αυτή και υπάρχει και νομοθετική πρόταση που θα μπορέσει να το κάνει αυτό πραγματικότητα. Αυτό από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά ε, δεν μπορούμε στους νέους να επιβάλλουμε αλλαγή συμπεριφοράς με τον νόμο, επειδή έχουμε θετήσει συγκεκριμένη νομοθεσία. Μιλούμε για εκπαίδευση, για αγωγή, να μάθουν να εκτιμούν το περιεχόμενο. Και αυτό είναι ανάγκη να ξεκινήσουμε να το κάνουμε από την πολύ νεαρή ηλικία. Ίσως να έχουμε πρέσβεις προσωπικότητες που οι νέοι γνωρίζουν. Άλλο είναι ε, κάτι που βγαίνει από το στόμα ενός ανθρώπου που οι νέοι ε, θαυμάζουν δεν έχει, έχει πολύ μεγαλύτερη ισχύ αυτό το μήνυμα από το μήνυμα που βγαίνει από έναν εκπαιδευτικό ή καποιο γονέα μόνο. Ούτε αυτά είναι βέβαια μελιτέα. Από εκεί και πέρα πρέπει να δείξουμε ποια θέση έχει ο χώρος της, ε, του πολιτισμού. Η βιομηχανία της δημιουργίας πολιτιστικών έργων είναι ο τρίτος κλάδος στην ευρωπαϊκή οικονομία. Ένα από τα success stories, ιστορίες επιτυχίες στην Ευρώπη είναι το animation το ευρωπαϊκό, οι ταινίε τέτοιου είδους. Νέοι μπορούν να απασχοληθούν χάρη στο λογισμικό, χάρη στις νέες τεχνολογίες. Ε, είμαστε πρωτοπόροι και μπορούν να βρουν θέση απασχόλησης η οποία θα είναι ενδιαφέρουσα και η οποία θα έχει και καλή αμοιβή. Ε, είναι ένας πολύ σημαντικός κλάδος της ευρωπαϊκής οικονομίας. Πρόκειται για μία από τις βασικές βιομηχανίες και σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε για τον αλφαβητισμό, τον ψηφιακό και τη δυνατότητα απασχόλησης. Δεν υπάρχει μία μαγική συνταγή, ε, ένα μαγικό ραβδάκι, αλλά χάρη στη ψηφιακή εποχή μπορούμε όλοι να συνδυαστούμε και να συνδυάσουμε τα διαφορετικά επίπεδα για να τα κάνουμε όλα αυτά πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σοφρίν. Ευχαριστώ. Θέλω να ρωτήσω την Επίτροπο για αυτό το ζήτημα των fake news. Είπατε ότι δεν υπάρχει ορισμός. Συμφωνείτε μαζί μου ότι θα πρέπει αυτός ο ορισμός να είναι σφιχτός, στενός ε, και να αφορά πράγματα, ισχυρισμούς οι οποίοι πραγματικά μπορούν να διαψευστούν και όταν πρόκειται για σκόπιμη προσπάθεια να παραπληροφορήσει κανείς, γιατί κάποιες φορές πολιτικοί επιλεκτικά ε, επιλέγουν ενδεχομένως κάποια επιχειρήματα για να τονίσουν την δική τους θέση. Ο κύριος Ντράγκη, για παράδειγμα, θα μπορούσε να πει ότι η Ευρωζώνη είναι μια ιστορία επιτυχίας γιατί κοιτάξτε τι έγινε τους τελευταίους 18 μήνες με την ανάπτυξη εγώ από την άλλη μεριά θα μπορούσα να πω το αντίθετο ότι η Ευρωζώνη είναι μια αποτυχία λαμβάνοντας υπόψη όλη την ιστορία της τα τελευταία δέκα χρόνια. Κανείς από, από τους δυο μας όμως δεν θα διέδιδε ψευδείς ειδήσει, όποια άποψη και αν ε, εξέφραζε. Και μετά τις αμερικανικές εκλογές υπήρχαν όντως κάποιες ιστοσελίδες οι οποίες ε, στο Twitter για παράδειγμα έλεγαν ότι ο Ντόναλτ Τραμπ για παράδειγμα πήρε τις περισσότερες ψήφους. Αυτό είναι πράγματι fake news, είναι ψευδής είδηση διότι δεν είχε λάβει τις περισσότερες ε, ψήφους. Ωστόσο θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι η εμπιστοσύνη ε, στις δημόσιες αρχές είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και αυτό που είπατε ε, μια μονάδα δηλαδή που θα εξασφαλίζει την επαλήθευση των ειδήσεων ενδεχομένως θα μπορούσε να, να γίνει αντικείμενο κατάχρησης ε, και να χρησιμοποιηθεί για μια φιλοενωσιακή ε, προπαγάνδα. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι ένα στόχο τον οποίο μπορούμε να τον εξυπηρετήσουμε ή θέλουμε να τον εξυπηρετήσουμε όλοι μας. Oui, la question est oui. Η απάντηση είναι ναι πρέπει να προτείνουμε έναν ορισμό που θα αντέχει σε οποιαδήποτε δοκιμασία. Δεν μπορούμε να έχουμε έναν ορισμό μεταβλητής γεωμετρίας. Και γι' αυτό το είπα εξ αρχής. Ψευδείς ειδήσει δεν είναι η γνώμη, η άποψη, ούτε η ηρωνία, ούτε η αίσθηση. Στον ορισμό πρέπει να ορίσουμε κριτήρια ε, που θα μας βρίσκουν ομόφωνα σύμφωνους και το υπογραμμίζω. Δεν θα έχουμε Υπουργείο Αλήθειας, ούτε Υπουργείο Λογοκρισίας. Δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοια πράγματα. Και γι' αυτό σήμερα θέλουμε να διατηρήσουμε τις θεμελιώδεις μας ελευθερίες, την ελευθερία του εκφράζεστε και την ελευθερία της πρόσβασης στην πληροφόρηση, αλλά να επιθεωρήσουμε, να εποπτεύσουμε αυτή τη φανταστική ικανότητα των ηλεκτρονικών πλατφόρμων να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης και να έχουν start-up και επιχειρήσεις που θα ανθίσουν, θα ανοίξουν τα φτερά τους στη συνέχεια. Είναι πολύ λεπτή αυτή η ισορροπία. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Στον ορισμό πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Ευχαριστούμε πολύ. Προτού περάσουμε σε ένα δεύτερο γύρο τοποθετήσεων, θέλω να κάνω εγώ ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει τεθεί ακόμη. Η Κομισιόν δυστυχώς δεν κατάφερε στην Συμφωνητή χρονικη χρονική έντε 11-2017 δηλαδή, να υποβάλει μια ενδιάμεση ε, αξιολόγηση του προγράμματος Creative Viewer και το λέω μεταξύ μας ότι κανονικά κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο η Κομισιόν να μην τηρεί τέτοιες ε, προθεσμίες που έχουμε συμφωνήσει. Εν πάση περιπτώσει, ε, βρισκόμαστε και στο στάδιο που σκεφτόμαστε ένα νέο πρόγραμμα. Η Κομισιόν, εξ όσων γνωρίζω, ήδη εργάζεται επ' αυτού και κυκλοφορούν ήδη διάφορες φήμες σχετικά με ένα πιθανό ε, μελλοντικό πρόγραμμα Creative Viewer και την πιθανότητα να υπάρξει μια ένα σπάσιμο μεταξύ του, του, του, του προγράμματος για τα μέσα και του προγράμματος για τον πολιτισμό. Εσείς είπατε ότι ε, θα θέλατε να ενισχύσετε αυτές τις δύο διαστάσεις, και είπατε και στο Βερολίνο, σας ακούσαμε, πόσο σημαντικό είναι για εσάς ε, το πρόγραμμα για τα, για τα οπτικοακουστικά μέσα και πόσο σημαντικό είναι και για την ε, κινηματογραφική βιομηχανία. Μπορείτε μήπως σήμερα να μας δώσετε ε, κάποιες σκέψεις ε, για το ποιο θα μπορούσε να είναι το μέλλον ε, για τα media. Θα παραμείνει συγχωνευμένο με το Creative Viewer, θα αποτελέσει αυτόνομο πρόγραμμα στο μέλλον. Για μας αυτό που είναι σημαντικό είναι η αναγνωρισιμότητα και η ορατότητα του πολιστικού προγράμματος, που δεν είναι στην αρμοδιότητά σας, αλλά του προγράμματος για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα χαρακτηρίζεται από ένα ευρωπαϊκό σήμα θα έχει έναν ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Να διατηρηθεί δηλαδή αυτή η πτυχή και να μην χαθεί μέσα σε μια ευρύτερη σούπα που θα τα περιλαμβάνει όλα. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες πρώτες σας σκέψεις από αυτού. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και... Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να προβλέψουμε το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Δεν έχουμε αρκετά στοιχεία για να κάνουμε προβλέψεις αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι τι υπερασπιζόμαστε εμείς. Ε, το πρόγραμμα Media είναι μία από τις πιο θαυμάσιες ιστορίες επιτυχίας. 2,4 δις ευρώ έχουμε αφιερώσει σε 26 χρόνια. 2.000 προγράμματα χρηματοδοτούμε κάθε χρόνο. Είναι απαραίτητο να διατηρηθεί. Είναι εμβληματική επιτυχία. Για μένα λοιπόν η απάντηση είναι όχι. Δεν θα υπερασπιστώ θέση που θα αραιώσει το πρόγραμμα, θα το υπονομεύσει. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό για το πρόγραμμα. Κανείς δεν μπορεί να προδικάσει αν αυτό θα γίνει. Αλλά ξέρουμε ότι υπάρχει άλλος προϋπολογισμός μεταξύ 2014 και 2020. Είναι Δηλαδή 2014-2020 είχαμε στραγάλια για χρήματα ουσιαστικά, ελάχιστα και παρόλα αυτά χρηματοδοτήσαμε σπουδαία έργα. Πρέπει να προβληματιστούμε για την περίοδο 2018-2020 και πρέπει να αναθεωρήσουμε ορισμένες δράσεις. Έχουμε 14 ε, σχήματα με 20 διαφορετικές δράσεις. Ίσως πρέπει να τα αναθεωρήσουμε αυτά, να έχουμε λιγότερο σε στοιχεία και αριθμούς και περισσότερο σε ε, προοπτικές και σε αντίκτυπο, σε επίδραση. Είμαστε ανοιχτοί στη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μπορέσουμε να το υπερασπιστούμε και στις διαπραγματεύσεις για το επόμενο πολιτεύσιο δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ. Όσον αφορά την ενίσχυση αυτού του προγράμματος, ε, θα έχετε σίγουρα στο πλευρό σας εμάς, την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, και για τον νέο προσανατολισμό του ε, προγράμματος βεβαίως θα ήταν πολύ χρήσιμο να γίνει αυτή η ενδιάμεση αξιολόγηση για να δούμε ποια κατεύθυνση πρέπει να χαράξουμε, τι θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε, τι θα μπορούσαμε να αφήσουμε πίσω. Γι' αυτό και θα ήταν ε, πολύ χρήσιμο αν ολοκληρώνεται αυτή την ενδιάμεση αξιολόγηση σύντομα. αλλά 12 λεπτά. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στη Χέλγα Τρούπελ που ξαναζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ Πέτρα. Θέλω να ε, αναφερθώ σε δύο συγκρούσεις στόχων. Δεν είναι η πρώτη φορά που το συζητούμε άλλωστε. Αφενός είναι αλήθεια ότι οι ψηφιδές ειδήσει δεν είναι νέο φαινόμενο. Υπήρχε πάντοτε στην ιστορία της ανθρωπότητας. Όμως με το ίντερνετ η διάδοση, η κλίμακα διάδοσης αυτών των ψευδών ειδήσεων είναι τελείως διαφορετική και προφανώς χρειαζόμαστε ορισμό. Αλλά ας μην ξεχνάμε αυτό που είπε ο Τραμπ για τα, για, τις για τα εναλλακτικά στοιχεία, τα εναλλακτικά γεγονότα. Έχουμε λοιπόν κάποιες ε, περιπτώσεις όπου ε, ρομπότ, bots ε, από τη Ρωσία για παράδειγμα, προσπαθούν να επηρεάσουν την ευρωπαϊκή, τη δυτική κοινή γνώμη. Δεν πρέπει λοιπόν να είμαστε αφελεί. Προφανώ και είναι ορθό ότι αν θέλουμε να έχουμε ευφυή νομοθεσία, δεν μπορούμε να παραβιάσουμε την ελευθερία του τύπου. Και εδώ πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Αλλά το να είναι κανεί προσεκτικό δεν σημαίνει να μην αναλαμβάνει καμία δράση. Πρέπει να υπάρχει έξυπνη νομοθεσία, όχι υπερβολική νομοθεσία, ε, ούτε όμως μπορεί κανείς να κάνει ό,τι θέλει στο τοπίο των media, γιατί αυτό σημαίνει ότι τα bot θα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν μέσω του ίντερνετ. Δεύτερον, για το copyright και ε, για τον κινηματογράφο και αυτήν την ψηφιακή δημόσια πλατφόρμα. Γιατί η συνάδελφος Μίχηλ είπε ότι υπάρχει ε, υπερβολική προσήλωση του, της βιομηχανίας στις, στις άδειες χρήσης και στην εδαφικότητα. Προφανώς, αν θέλουμε να υπάρχει ευρωπαϊκή βιομηχανία κινηματογράφου, θα πρέπει να υπάρχει διασυνοριακή τρόπος να έχει κανείς πρόσβαση σε αυτές τις ευρωπαϊκές ταινίες, διότι διαφορετικά πρόκειται για εκμετάλλευση των δημιουργών. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Αν θέλουμε διασυνοριακή πρόσβαση θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι δημιουργοί θα πληρώνονται. Και εδώ δεν υπάρχει καμία αντίφαση, αλλά το να λέμε ε, εδώ και 8 χρόνια ε, τα ίδια και τα ίδια, ε, δεν πείθει πια. Πρέπει να βρούμε νέους τρόπους ε, χρηματοδότησης προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τους στόχους. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκάβριελ. Ευχαριστώ κυρία Τρουπελ για τα fake news. Συμφωνώ μαζί σας. Γι' αυτό ξεκινήσαμε και αυτή τη δουλειά. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να παρατηρούμε αμέτωχοι τόσα συμβαίνουν. Από την άλλη, σας το είπα και από την αρχή, δεν έχουμε φτάσει σε επίπεδο να χαράξουμε νομοθεσία, γιατί για να νομοθετήσουμε πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε να ρυθμίσουμε. Πρέπει δηλαδή να αναγνωρίσουμε καλύτερα τις διαστάσεις του προβλήματος και γι' αυτό προτείνω στην ομάδα και γι' αυτό περιοριζόμαστε στην ανακοίνωση το του 2018, όχι νομοθεσία δηλαδή. Ας καταλάβουμε πρώτα ποιο είναι το πρόβλημα, ας εντοπίσουμε μηχανισμούς, δράσεις πρώτα απ' όλα και μετά ας δούμε ποια συνέχεια θα δώσουμε. Για το γεωγραφικό προσδορισμό, ναι, συμμεριζόμαστε τους στόχους. Πρέπει ο δημιουργός, ο πνευματικός και ο ερμηνευτής να έχουν την αμοιβή που ε, είναι η σωστή. Είναι θέμα δικαιοσύνη. Αλλά για το κάψατ θέλω να αναφέρω κάτι το οποίο πολύ συχνά έχει παρερμηνευθεί. Δεν παρεμποδίζουμε την δυνατότητα σύναψης συμβάσεων Θέλουμε μόνο να δώσουμε τη δυνατότητα σε ορισμένου να κάνουν αυτή την επιλογή. Όπως είπα χθε, έγινε ο πρώτος τριμερής διάλογος, έγινε μια καλή συζήτηση σε θετικό κλίμα και αν όντω χρειάζεται να διευκρινιστούν κάποια ζητήματα, μέσα από τον τριμερή διάλογο αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί. Ταυτόχρονα σήμερα Α σκεφτούμε πώ θέλουμε να αναπτυχθεί αυτή η ενιαία ψηφιακή αγορά μια σειρά πολιτών, όπως οι παραδείγματοι αυτοί που ανήκουν σε μειονοτικές γλώσσες, να μην κινδυνεύουν όταν ανοίγουν τη τηλεόραση ή τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή να αντιμετωπίσουν μια μαύρη οθόνη. Αυτοί είναι που δεν καταλαβαίνουν τι χρησιμότητα φέρνει αυτή η ενιαία ψηφιακή αγορά. Είναι δύσκολη περίπτωση, ναι, το ομολογώ, αλλά πρέπει να διατηρήσουμε υψηλέ τις φιλοδοξίες μας και ταυτόχρονα να περιοριστούμε στο ουσιώδες και πολύ χρόνο δεν έχουμε γιατί είναι κρίσιμη σημασία το 2018. Στο τέλος του χρόνου δηλαδή θέλουμε να έχουμε ολοκληρώσει το σύνολο των προτάσεων που είναι επιτάπητο. 44 πρωτοβουλίες, 25 νομοθετικές, 11 μόνο έχουν ολοκληρωθεί. Επομένως, αν θέλουμε πράγματι να δείξουμε στον πολίτη ότι μεριμνούμε για την κυβερνοασφάλεια, της ε, ε, δυνατότητες για την ευρωπαϊκή βιομηχανία να έχει την πρωτοκαθεδρία για το ψηφιακό περιεχόμενο και την επιμόρφωση πρέπει να ξεκινήσουμε και να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Δεν ε, διαφωνούμε εμεί στην Επιτροπή μα. Δεν λέμε είτε το ένα είτε το άλλο, αλλά θέλουμε και τα δύο να τα προωθήσουμε και την προστασία του πνευματικού δημιουργού που θα πρέπει να έχει μια κατάλληλη, μια σωστή και προσήκουσα αμοιβή, αλλά ταυτόχρονα και τη δυνατότητα για πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο στους, για του πολίτε. Ε, το μόνο που μένει να βρούμε ποιο είναι ο σωστότερο δρόμο. και εκεί βέβαια είναι και μεγάλε δυσκολίε. Ακόμη ένα άνθρωπος έχει στήσει το λόγο. Κύριε Φλάνναγκαν, πάρα πολύ στο. Ευχαριστώ. Και μια και μου απαντήσατε ότι μου έχετε στείλει επιστολή, ε, από την ώρα που μου απαντήσατε μάλλον, απέστειλα εγώ μήνυμα στην, στο γραφείο μου και τους ρώτησα λάβατε τίποτα και μου λένε όχι, καθόμαστε πάνω στην, ε, μπροστά στην οθόνη, χτυπάμε συνέχεια το κουμπί για να δούμε αν έφτασε κάτι. Εάν λοιπόν μου ε, αποστήλατε απάντηση, γιατί δεν μου απαντήσατε στο δεύτερο mail που σας λέω, μα δεν μου έχετε απαντήσει. Και επίσης πώς μπορούμε να ορίσουμε αυτή τη συνάντηση μεταξύ ημών, εμού και του συναδέλφου, του δημοσιογράφου, γιατί είμαι βέβαιο ότι θα πέστε από την καρέκλα σα όταν ακούσετε τι έχουμε να σα πούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό ο άνθρωπο να είναι ικανό να αντιμετωπίσει το θέμα των fake news. Μην ξεχνάμε ότι η διάδοση ψευδών ειδήσεων μάλιστα έχει ξεκινήσει από το γραπτό τύπο και όχι από τον ηλεκτρονικό. Η πρόεδρο, ευχαριστώ. Νομίζω ότι έφτασε το μήνυμα. Έχει προφανώς αποσταλεί η επιστολή, δεν τη λάβατε απλώς εσείς κύριε Φλάναγκαν. Κυρία Γκαμπριέλη, είμαι βέβαια ότι θα με ρημνήσετε, θα μιλήσετε με το επιτελείο σας ώστε να ξανασταλεί η επιστολή και βεβαίως διμερώς να βρείτε με το ε, προσωπικό σας τη δυνατότητα για μια συνάντηση όπως τη ζήτησε ο συνάδελφος. Καλώς, έτσι ολοκληρώνουμε αυτό το κομμάτι στην ημερήσια μας διάταξη. ευχαριστώ θερμά για την πολύ καλή διάθεση για συνεργασία, για συνομιλία, για τη δεξιοδική συζήτηση. Ξέρω ότι είναι πολύ πιο κουραστικό αυτό το πινκ-πονγκ που κάνουμε, γιατί καλείστε να δώσετε απαντήσει σε πολύ περισσότερα ερωτήματα, αλλά από την άλλη καλό είναι να έχουμε λεπτομερέστερες απαντήσεις αντί ένα πακέτο απαντήσεων μέσα στις οποίες χάνουμε και την ε, εστίαση. Αυτά λοιπόν δεν είναι βέβαια τελευταία σας ε, επίσκεψη. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τις πολλές και καλές ερωτήσεις και την ε, πολύ καλή συζήτηση που είχαμε σήμερα. Σας εύχομαι καλή ημέρα, καλό απόγευμα. Και τώρα ένα σύντομο διάλειμμα, πέντε λεπτάκια. Για να συνεχίσουμε με την ακρόαση για την πρόσβαση στο πολιτιστικό περιεχόμενο. Λοιπόν, συνάδελφοι, ας συνεχίσουμε. Έχουμε την υπόλοιπη συνεδρίασή μας που θα αφιερωθεί στο θέμα της πρόσβασης στο πολιτιστικό περιεχόμενο. Ξεκινάμε με ακρόαση και αμέσως μετά θα γίνει ανταλλαγή απόψεων για το σχέδιο έκθεσης με το αντίστοιχο θέμα Είναι η πρώτη φορά που η Επιτροπή μας ε, αποφάσισε να συντάξει ε, έκθεση πρωτοβουλίας. Ο κ. Στογεύσκη είναι ο εισηγητής μας και φαντάζομαι ότι βεβαίως θα συμμετάσχει ενεργά στη συζήτηση. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η άποψη, η άποψη των εμπειρογνωμόνων που έχουμε προσκαλέσει ως προς το ποια, ποια είναι τα εμπόδια, ποια είναι η φραγμή που έχετε εντοπίσει που βρίσκονται, αλλά και πώς μπορούν να ξεπεραστούν οι φραγμοί αυτοί. Μιλήσαμε μόλις και με την Επίτροπο. Είχαμε πολύ καλή εμπειρία με αυτή τη διαδικασία ping-pong. Ε, αποδεικνύεται πάντοτε ότι εξασφαλίζει τη ζωηράδα της συζήτησης και την αποτελεσματικότητά της. Θα πρότεινα λοιπόν να το ξανακάνουμε έτσι. Δηλαδή, θα δώσουμε το λόγο για 10 λεπτά σε κάθε έναν από τους προσκεκλημένους μας ώστε να τοποθετηθεί για το θέμα αυτό. Στη συνέχεια θα γίνει μια δεκάλεπτη ε, διαδικασία έρωτα απαντήσεων. Γρήγορες απαντήσεις όσο γίνεται, ε, γρήγορες ερωτήσεις, γρήγορες απαντήσεις όσο γίνεται. Okay, five. Πέντε, πέντε, εντάξει. Πέντε λοιπόν, 5 λεπτά η παρουσίαση από τους εμπειρογνώμονες και μετά 10 λεπτά ερωταπαντήσεις και θα δούμε πώς θα πάει. Καταρχάς να σας παρουσιάσω τους προσκεκλημένους μας. Έχουμε τον Πέρα Αλμέδα που είναι ε, επιστήμον, πολιτικός επιστήμον στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης και συντονιστή της Φουντατσιό Καταλούνια Ευρώπα. Jill Κάζινς που είναι ευθύνουσα σύμβουλος της, ε, του Europeana Foundation, Φρέντερικ Μεσέουφ, που είναι επικεφαλής σύμβουλος στο Σάντρ Μποζάρ, τον Ντίκ Μολνάρ, που είναι φοροτεχνικός στο All Arts Tax Advisors και ερευνητής του Πανεπιστημίου Εράσμου του Ρότερνταμ. Είχαμε προσκαλέσει και έναν πέμπτο προσκεκλημένο, τον Όλαφ Τσίμερμαν, διευθυντή του Πολιστικού Συμβουλίου της Γερμανίας. Ωστόσο, δυστυχώς ε, έχει αρρωστήσει, τον έπιασε η γρήπη. Δεν μπόρεσε λοιπόν να παραστεί σήμερα εδώ ζητήσει γνώμη, αλλά νομίζω ότι οι τέσσερις ε, που κατάφεραν να έρθουν θα μας εξασφαλίσουν μια πολύ γόνιμη και ζωηρή συζήτηση. Ξεκινούμε λοιπόν με τον κύριο Αλμέδα και στη συνέχεια οι υπόλοιποι προσκεκλημένοι μας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ για την ε, πρόσκληση που μου απευθύνατε να συμμετάσχω σε αυτή την ακρόαση. την ακρόαση αυτή για, τη, για τα δομικά και οικονομικά εμπόδια στις πρόσβαση στον στο πολιτισμό. Σκοπός μου είναι να παρουσιάσω μια έκθεση που κάναμε με τους συναδέλφους από το Ίδρυμα για την Καταλωνία και την Ευρώπη το 2016 που δείχνει πώς εξελίχθηκαν οι δημόσιες δαπάνες για το πολιτισμό μεταξύ 2007 και 2015. Έχουμε ενημερώσει με νέα στοιχεία την έκθεση αυτή από τη στιγμή που έχουν παρεμβληθεί σχεδόν δύο χρόνια από τότε που δημοσιεύθηκε και θα ήθελα να αναλύσω και να αξιολογήσω τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης που ξέσπασε το 2007-2008 και τον αντίκτυπο των πολιτικών λιτότητας στις δημόσιες δαπάνες για τον πολιτισμό στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος λοιπόν και υπόθεση εργασίας της μελέτης αυτής ήταν να δούμε και να επιβεβαιώσουμε το κατά πόσο η οικονομική κρίση και οι πολιτικές λιτότητες επηρέασαν επηρέασαν ή όχι και με ποιο τρόπο τις πολιτιστικές πολιτικές και τους προϋπολογισμούς για την κουλτούρα και τον πολιτισμό στις διάφορες χώρες και πώς επηρέασαν την πρόσβαση στα προϊόντα πολιτισμού που είχαν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Και εδώ τα αποτελέσματα και τα πορίσματα επιβεβαίωσαν την υπόθεση εργασίας, ότι δηλαδή η οικονομική κρίση είχε ως αποτέλεσμα την υποχώρηση της δημόσιας υποστήριξης στον πολιτισμό και θελήσαμε να δούμε ποιοι είναι οι, νέοι μηχανισμοί και νέα εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να ενισχύσουμε τη σύγκληση των πολιτιστικών πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρώτη έκπληξη δεν υπάρχουν ενημερωμένες μελέτες για τις δημόσιες δαπάνες σε θέματα πολιτισμού στην Ευρώπη. Και οι μελέτες που είχε κάνει το Συμβούλιο της Ευρώπης σε μορφή compendium εγκαταλείφθηκαν το 2011. Δράτομαι λοιπόν της ευκαιρίας της σημερινή μου παρουσίας εδώ για να σας πω ότι είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε πόσα ξοδεύουν οι κυβερνήσεις για τον πολιτισμό στην Ευρώπη. Ε, η μελέτη δική μας είναι μία από τις ελάχιστες που υπάρχουν με ενημερωμένα στοιχεία, επικαιροποιημένα. Να δούμε όμως και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήσαμε. Χωρίσαμε τις ευρωπαϊκές χώρες σε τέσσερις μεγάλες γεωγραφικές ομάδες, νότος, κέντρος, ε, ανα... νότος, κέντρο, ανατολή και βοράς. Θεωρήσαμε ότι οι χώρες αυτές είχαν συμπεριφορές αρκετές παρε, αρκετά όμοιες και παρεμφερείς και η μελέτη ήρθε και το επιβεβαίωσε αυτό και συγκρίναμε με τα στοιχεία της Eurostat. Και αυτή είναι η πρώτη γραφική παράσταση που θέλουμε να σας δείξουμε. Αυτό επιβεβαιώνει ότι οι δημόσιες δαπάνες στο πολιτισμό στα 28 κράτη-μέλη μειώθηκαν κατά 3% από το 2007 ως το 2015 με πραγματικούς αριθμούς και το βάρος του πολιτισμού τον ε, κρατικό προϋπολογισμό από το 1,14 πήγε στο 1,01 ε, μέσα σε λίγα χρόνια. 113 ευρώ ανακάτοικο δημόσιες δαπάνες για τον πολιτισμό 6 ευρώ λιγότερα από ό,τι το 2007. Τι βλέπουμε σε αυτό το γράφημα. Έχουμε δύο μεγάλα μπλοκ χωρών. Οι χώρες του Βορρά και του κέντρου της Ευρώπης, της κεντρικής Ευρώπης, ε, διατηρούν και έχουν αυξήσει κιόλα τις δημόσιες δαπάνες στο θέμα του πολιτισμού κατά τα χρόνια κρίσης για να αντισταθμίσουν τις αντικυκλικές πολιτικές στην οικονομική τους ε, κατάσταση. Και υπήρξε τεράστια υποχώρηση, αντιθέτως, τεράστια μείωση 30% μειώθηκαν οι δημόσιες δαπάνες για τον πολιτισμό κατά κεφαλήν στις χώρες του Νότου και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης είχαμε μία ελάχιστη σύγκληση. Ε, για παράδειγμα, το 2007 στη Δανία 247 ευρώ ανά άτομο δαπανόταν για θέματα πολιτισμού το έτος, το 2015 271 ευρώ ανά άτομο, ενώ στην Ελλάδα από 128 ευρώ ανά άτομο οι δημόσιες δαπάνες στον πολιτισμό το 2015 υπήρξε μείωση στα 15 ευρώ ανά άτομο δημόσιες δαπάνες για θέματα πολιτισμού. Αλλά έχουμε και άλλα νούμερα 36% μείωση στην Ισπανία δημόσιες δαπάνες σε θέματα πολιτισμού. Ε, πολλής λόγος μπορεί να γίνει. Μιλούμε για μια ε, πολιτιστική φούσκα. Τα χρόνια των παχαιών αγελάδων έγιναν τεράστιες επενδύσεις σε θέματα πολιτισμού και στα χρόνια ισχνών αγελάδων η ε, η κουλτούρα και ο πολιτισμός ήταν η τελευταία προτεραιότητα, ο πιο αδύναμος κρίκος στο κράτος πρόνοιας. Και εδώ βλέπουμε το σχετισμό μεταξύ του ΑΕΠ, του κατακεφαλήν ΑΕΠ και των πολιτιστικών δαπανών, των κατακεφαλήν δαπανών. Το 2007 δύο μεγάλες ομάδες που πλησίαζαν μεταξύ τους τα στοιχεία και συγκριτικά το 2015 αυτές οι δύο μεγάλες ομάδες έχουν ακόμα μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους. Μεγάλη ροχμή, μεγάλο χάσμα και αυτό προϋποθέτει και δείχνει ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν πρόσβαση στον πολιτισμό μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό ενώ πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες απομακρύνονται από το στόχο της σύγκλησης. Και έχουμε αυτούς τις δύο πολύ διαφορετικές ομάδες. Τώρα, τρίτη εικόνα που θα θέλω να τονίσω και στο γύρο των ερωτήσεων μπορώ να μπω και σε λεπτομέρειες αν θέλετε και να τα αναλύσω περισσότερο. Οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, κάτι που μας εκπλήσει και αξίζει να το αναλύσει κανείς περισσότερο με περισσότερες λεπτομέρειες ότι το ποσοστό επενδύσεων στον προϋπολογισμό, στον κρατικό προϋπολογισμό είναι πολύ ανώτερο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό Μεσοόρο Ίσως αυτό οφείλεται στην παράδοση, στην πολιτική κουλτούρα, στην μετάβαση από το κομμουνιστικό σύστημα στο δημοκρατικό φιλελεύθερο σύστημα. Είναι κληρονομιά του παρελθόντος, είναι ανάγκη να ε, επιβεβαιώσουν την ε, ε, πολιτιστική τους ταυτότητα. Σε κάθε περίπτωση υπερέχει σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και συγκριτικά με τις χώρες του Νότου, οι οποίες υπολείπονται πάρα πολύ και υστερούν σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Μεσόωρο. Μιλούμε πάντοτε για το ποσοστό των δημοσίων δαπανών του προϋπολογισμού που απευθύνεται και προορίζεται για τον πολιτισμό. Βεβαίως το ποσοστό ε, που αφαιρώνεται στην υγεία ή στην εκπαίδευση έχει μειωθεί πολύ περισσότερο. Και ε, κάτι το σημαντικό και ολοκληρώνω για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας είναι το εξής. Δημόσιες δαπάνες της κεντρικής κυβέρνησης μειώθηκαν σε αυτή την περίοδο 2007 με 2015 και μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα στις, εθνικές, στις τοπικές αυτοδιοικήσεις. Είναι παραδειγματική περίπτωση της Ελλάδας όπου οι Δήμοι η τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση πριν από την κρίση οι δαπάνες για τον πολιτισμό ανήλθε στο 3% του του τοπικού προϋπολογισμού και μετά από το 2015 οι δαπάνες ήταν πάνω του 50% του δημοτικού πλέον προϋπολογισμού. Δηλαδή βλέπετε ότι το κράτος εκχωρεί πλήρως αυτή την αρμοδιότητα στους Δήμους. Και αυτό συμβαίνει σχεδόν παντού στην Ευρώπη. Τεράστια υποχώρηση των δημοσίων δαπανών στον προϋπολογισμό, τεράστια υποχώρηση και των δαπανών των οικογενειακών, ε, από τον οικογενειακό προπολογισμό ε, βέβαια, ο πολιτιστικός τομέας ε, μπόρεσε να βγει ενισχυμένος γιατί ε, κάποια μέρη του οικογενειακού προϋπολογισμού ανέλαβαν αυτή την ευθύνη. Τέλος, να έχουμε υπόψη μας τις δαπάνες που ανέλαβαν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στο σύνολό τους. Η Ευρώπη που δημιουργεί, το Ταμείο Συνοχής, όλα Αυτά είναι το 0,63% του ευρωπαϊκού ποροϋπολογισμού. 0,63%. Μιλούμε για 1,87 ευρώ ανά έτος, ανά πολίτη για θέματα πολιτισμού. Και πώς κατανέμονται όλα αυτά με άνισο τρόπο μέσα από το Ταμείο Συνοχής. Άρα εποφελούνται οι χώρες του Νότου και της Κεντρικής Ευρώπης, όμως για, το, για την Ευρώπη που δημιουργεί επωφελούνται κυρίως οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και του Βορρά χάρη στις επενδύσεις που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Αυτά είναι τα βασικά ε, πορίσματα και συμπεράσματα. Εάν θέλετε ευχαρίστω να μπούμε στις επιμέρους λεπτομέρειες όλων αυτών των θεμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι είναι η πρώτη μελέτη στην Ευρώπη για το πόσα χρήματα δαπανώνται από το Δημόσιο Κορβανά για τον πολιτισμό. Είναι λοιπόν πολύ ενδιαφέροντα και για, για μας αυτά τα πορίσματα. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να δώσω τον ε, λόγο πρώτα στον ε, εισηγητή μας, τον κύριο Στογεύσκη, για ένα-δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Όσον αφορά τις δαπάνες στην Ευρώπη, εγώ κάποτε ήμουν υπουργό πολιτισμού στην Πολωνία και θυμάμαι ότι οι δαπάνες μας ήταν ε, πολύ υψηλές. Και τα πράγματα είναι όπως ακριβώς τα παρουσιάζεται υπάρχει μειούμενη δαπάνη ε, σε χώρες όπως η Ιταλία, κάτι που συνδέεται και με το γεγονός ότι ε, πολύ συχνά αλλάζουν οι υπουργοί πολιτισμού. Όταν πήγα στην Ισπανία, ε, συνάντησα, κάθε φορά που πήγαινα στην Ισπανία ή στην Τσεχία ή στην Ιταλία, γνώριζα και άλλον υπουργό πολιτισμού. Ωστόσο, νομίζω ότι κάνατε ένα μεθοδολογικό σφάλμα που κατηγοροποιήσατε αυτές τις δύο χώρες, αυτές τις δύο κατηγορίες. Το 2015 η κατάσταση στη Γερμανία και στις κάτω χώρες ήταν πολύ διαφορετική. Οι κάτω χώρες ε, περιέκοψαν δραματικά τις δαπάνες στον πολιτισμό, ενώ η Γερμανία δεν το έκανε. Επίσης, ε, για τις ε, επιστροφές θυμηθείτε και μην ξεχνάτε ότι η κυβέρνησή μας ήταν εκείνη που θέλησε να αντλήσει χρήματα από τα διευθυντικά ταμεία για τον πολιτισμό μόνο. Εννιά ε, κράτη ήθελαν να υπάρχει τέτοια κατανομή ε, κονδυλίων για τον πολιτισμό ε, από τα διευθυντικά ταμεία. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονταν και η Πολωνία, 22% και μετά ήταν η Γερμανία και η Ιταλία, ενώ κάποιες χώρες βρίσκονται πραγματικά σε ένα απόλυτα ελάχιστο επίπεδο όσον αφορά τις επενδύσεις. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε την ε, κατανομή των ε, επενδύσεων σε κάθε χώρα ξεχωριστά. Γιατί υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί που διέπουν τις επενδύσεις στον πολιτισμό στα διάφορα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, στην Ισπανία ένα εισιτήριο για ένα κορίντα αποτελεί δαπάνη για ε, τον πολιτισμό. Ε, στις κάτω χώρες ε, ένα, μια κάρτα κάμπα επίσης είναι πολιτισμός. Τα λεφτά που δαπανάς για στυλό στη Γαλλία αποτελούν δαπάνη για τον πολιτισμό, αλλά όχι σε άλλες χώρες, δεν ισχύει σε άλλες χώρες αυτό. Οπότε πρέπει να ξεπεράσουμε αυτόν τον, ε, αυτό το εμπόδιο, το καταλαβαίνω, αλλά πρέπει, με κάποιο τρόπο να ενοποιήσετε τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείτε, την επιστημονική. Ευχαριστώ. Κύριε Αλμέδα, θέλετε να απαντήσετε στον κύριο Στογεύσκη. Ναι. Ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας. Η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε είναι ε, η εξής. Προσπαθήσαμε να δούμε τις διεθνείς δαπάνες για τον πολιτισμό με βάση τα διεθνή πρότυπα για τις πολιτιστικές υπηρεσίες έτσι όπως καθορίζονται από την Eurostat και το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών. Για παράδειγμα, αποκλείονται οι τηλεοράσει, στα κανάλια, τα ραδιόφωνα, το οπτικοακουστικό τομέα και περιλαμβάνονται τομεί που είναι συγκρίσιμοι και απαρεμφερεί και ομόλογοι μεταξύ των διαφορετικών χωρών. Ε, χρησιμοποίησαμε στοιχεία από την Ευρωστάτ και τα αποπληθωρικοποιήσαμε για να μπορέσουμε να κάνουμε τη σωστή συγκρίση ε, μεταξύ των διαφόρων χωρών και να είμαστε συνεπείς και συνεκτικοί στην ανάλυση αναχώρα και ανά περίοδο, δηλαδή σε βάθος χρόνου, να υπάρχει συνέπεια. Έχουμε όλα τα στοιχεία και μπορούμε να σας τα στείλουμε και άλλωστε τα πρακτικά ε, τα, ε, ε, μια περίληψη έχω αφήσει στην είσοδο της αίθουσας της έκθεσης αυτής και μπορείτε να τα διαβάσετε, να τη διαβάσετε αν σας ενδιαφέρει. Ευχαριστώ. Άλλες ερωτήσεις. Όχι από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή. Α, κύριε Στογεύση και εσείς παρακαλώ και θα ξαναπατήσετε. Ναι, Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να προσθέσω κάτι ακόμα. προδιαγραφές Ηνωμένων Εθνών και ε, Ευρωπαϊκής Ένωση είναι διαφορετικέ. Μπορεί να συμφωνούν σε κάποιες ε, βασικές ε, ιδέες και αρχές, αλλά η Eurostat έχει μπορέσει να ενοποιήσει τις αρχές για τις δαπάνες για το πολιτισμό το 2010 ενώ η δική σας η μελέτη πιάνει τα 2007-2015 ως έτη φαντάζομαι ότι είναι πολύ δύσκολο το έργο στο οποίο αποδεθήκατε και τα καταφέρατε μια χαρά συγχαρητήρια. Ja, vielen herzlichen Dank. Ναι, σας ευχαριστούμε πολύ για τους επένους Βεβαίως οι μελέτες μας ξεκινάνε από το 2007, το ένα έτος πριν από την έλευση της κρίσης και έχουμε αξιοποιήσει μόνο τα στοιχεία τα οποία είναι διαθέσιμα στη Eurostat και που έχουν εξελιχθεί. Κάποια στιγμή συνειδητοποίησαμε ότι η ίδια η Eurostat διόρθωσε, τροποποίησε κάποια από τα δικά της στοιχεία και επικαιροποιήσαμε την μελέτη αναλόγω. Το σαφές είναι ότι έχουν υπάρξει αλλαγές έκτοτε. Επομένως, αυτή τη στιγμή τα στοιχεία φτάνουν μέχρι το 2015 και ελπίζουμε ότι το 2016 τα στοιχεία για το 2016 θα τα συμπληρώσουμε τους επόμενους μήνες. Σας ευχαριστώ. Θα μένετε λίγο περισσότερο φαντάζομαι αν τυχόν ε, λίγο αργότερα προκύψουν και άλλα ερωτηματικά για σας. Επιφυλασσόμεθα. Και περνώ στον επόμενο. Στην επόμενη ομιλήτρια, την κυρία Cousins. Τα δικαιώματα των ε, παραγωγών ως εμπόδιο. Και σας δίνω το λόγο. Κυρία Cousins. Ευχαριστώ και καλησπέρα. Η διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κληρονομιάς έχει τα τελευταία χρόνια με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής από την Ευρωπαϊκή Ένωση πάρει νέα ορμή. Έχουμε να κάνουμε με την ενθάρρυνση του πολιτιστικού περιεχομένου της πολιτιστικής κληρονομιάς και το πλαίσιο της Ευρωπαίανα έχει αντιγραφεί και ε, τύχει απομίμηση σε όλο τον κόσμο, διευκολύνει την πρόσβαση ε, την ανταλλαγή ένα ισότιμο πεδίο επικοινωνία στα 28 κράτη-μέλη. ευρωπαία να καταγράφεται ως ένα από τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως το καταγράφει και η Σύνοδος του και το 2017. Ωστόσο, πρέπει να δούμε τι είδους πολιστική κληρονομιά είναι διαθέσιμη πέραν των σύνορων και στο διαδίκτυο. Υπάρχουν ακόμη φραγμοί, λοιπόν. Ο γεωγραφικός περιορισμός ε, των δικαιωμάτων του παραγωγού και οικονομική υποστήριξη και διατήρηση, προστασία του οικοσυστήματος Ευρωπαίνα. Θα ήθελα να αναφερθώ, γιατί είναι γνωστά βέβαια τα θέματα του copyright σε οικονομικά προβλήματα, παρά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2016 δεν έχουμε καμία βεβαίωση ότι η Ευρωπαίνα και η διασυνοριακή πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονομιά θα έχει επαρκή χρηματοδότηση. Χρειάστηκε χρήμα για να στηθεί το δίκτυο να ενοποιηθούν ε, τις της Ευρώπης για να εισφέρουν το, η πολιτιστική κληρονομιά, αλλά η διατήρηση αυτής της αλυσίδας ε, προμήθειας πολιτιστικής κληρονομιάς διαβρώνεται, κινδυνεύει, μειώνονται τα χρήματα χρόνο με το χρόνο και υπάρχει και συμβασμό σε σχέση με το... και διαπιστώνουμε ότι πρέπει να συμβαστούμε με την ιδέα ότι διαρκώς θα πρέπει να μειώνεται αυτή η χρηματοδότηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν μπορεί, πιστεύουμε, να αναλάβει δράση για να αποτρέψει τις αποτυχίες αυτές, αλλά δεν έχει τους κατάλληλους μηχανισμούς. Εάν λοιπόν θεωρούμε ότι η πολιτική κληρονομιά υπογραμμίζει και την έννοια του ανήκειν, την κοινωνική συνοχή, την καινοτομία και την εκπαίδευση στην Ευρώπη και είναι μηχανισμός για την ισότητα, τότε χρειάζεται και ισότιμη χρηματοδότηση μέσα στο πλαίσιο της έρευνας και της ανάπτυξης και της επιστήμης. Ε, χρειάζεται μια αφύπνιση λοιπόν, να είναι γνωστό ότι υπάρχει διαθέσιμο όλο αυτό το πολιτιστικό περιεχόμενο. Πρέπει να είμαστε σε θέση να χρησιμοποιούμε υλικό από διαχρονικά αρχεία εφημερίδων και μέτρα που μπορούν να ενισχύσουν την ε, αηφορία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μπορεί να δυσκολεύουν ε, τα θέματα του copyright και του να υψώνουν φραγμού στην ενιαία αγορά της πολιτιστικής κληρονομιάς. Πιστεύουμε. Θέλετε να μιλάτε λίγο πιο γρήγορα για να σας προλαβαίνουμε. Ναι, με συγχωρείτε επειδή εγώ τα αγγλικά τα έχω μητρική γλώσσα και αυτό μιλάω γρήγορα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι τα όργανα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς έχουν ρόλο θέματοφύλακα και σαφώς καθήκον για την παροχή του αποτελέσματος. Πρέπει να αναγνωριστεί ο τρόπος με τον οποίο όλοι μας θέλουμε να Έχουμε πρόσβαση και δυνατότητα κατανάλωσης πολιτιστικού περιεχομένου στο σχολείο, στο μάθημα, στα μέσα, στην ε, χρήση, ακόμα και την ανάπτυξη μιας εφαρμογής ηλεκτρονικής για την αναζήτηση πολιτιστικών ε, μνημείων, Φερρυπίν, για έναν επισκέπτη πόλης. Πρέπει λοιπόν ε, να βρούμε λύσεις με συμβεσμό μεταξύ των δικαιούχων, μεταξύ των θεματοφυλάκων και ημών Επομένως δεν υπάρχει αμφιβολία ως προς την ανάγκη για συμβιβασμό. Έχουμε αρκετή επιτυχία στις διάφορες αγορές. Με αδελφοποίησης 300 ε, διδασκόντων από 20 χώρες, 22 χώρες. Ε, ε, το πρόβλημα δεν είναι ότι η κυρία μιλάει γρήγορα. Το πρόβλημα είναι ότι διαβάζει ένα κείμενο το οποίο δεν έχει δώσει στους διερμηνείς και ως εκ τούτου δεν ξέρει ακριβώς πώς να τονίσει τις προτάσεις της. Οι διερμηνείς παρόλα αυτά συνεχίζουν την προσπάθεια. Θέλουν λοιπόν υλικό από τον 20ο αιώνα και εδώ βλέπουμε μια γελιογραφία την οποία ίσως να έχετε δει και εσείς. Χρειάζεται οπτικό-ακουστικό υλικό, Υπάρχουν πολλές ταινίες τεκμηρίωσης που θα μπορούσαν να διατηθούν αν δεν έπρεπε να περάσουμε από τη διαδικασία αδειοδότησης για κάθε δικαιούχο. Μπορεί να είναι χρήσιμο και για την ιστορία το ίδιο αυτό υλικό. Υλικό που καλύπτεται ακόμη από τα δικαιώματα του παραγωγού, χωρίς όμως να είναι διαθέσιμο στο εμπόριο. Πρέπει να είναι δυνατόν λοιπόν αυτό το υλικό το οποίο δεν υπάρχει στο εμπόριο να το χρησιμοποιούν οι αρμόδιοι φορείς και άρα το πλαίσιο για την προστασία των πνευματικών δημιουργών πρέπει να τροποποιηθεί. Είναι τεράστιο το έργο της εξασφάλισης αδειών για τον κάθε παραγωγό προκειμένου να μπει το υλικό στο διαδίκτυο είναι μια μαύρη τρύπα και όπως είπα είναι μεγάλος όγκος του υλικού που δεν διατίθεται στο εμπόριο αλλά ανήκει ε, η άδεια σε κάποιες εταιρείες διαχείρισης. Μπορεί κάποιες λύσεις που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να, δίνουν, ε, να αποδεσμεύουν ορισμένο περιεχόμενο αλλά όχι όλο Πρέπει λοιπόν όπου δεν υπάρχει αδειοδότηση ε, να μπορούν να ε, αξιοποιούν μια παρέκκληση οι αρχές δυνάμει της νομοθεσίας. Επίσης η εναρμόνιση της εξαίρεσης προκειμένου να διαφυλαχθεί και αυτό πρέπει να είναι υποχρεωτικό. Ωστόσο η πρόταση της Επιτροπής δεν δίνει σαφή εικόνα για το αν η ψηφιοποίηση καλύπτεται από αυτή την παρέκκληση και αν αυτό συμβεί, αν όντω δεν υπάρχει δηλαδή αυτή η παρέκκληση, τότε μόνο περισσότερη αμφιβολία και ασάφεια θα επικρατήσει σε σχέση με την ενσωμάτωση σε ψηφιακό περιεχόμενο. Τρίτον, το υλικό που ανήκει σε, σε αναλογική μορφή στο δημόσιο χώρο πρέπει να παραμένει στο δημόσιο χώρο και για το ψηφιακό περιεχόμενο. Βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι προσπαθούν να αποκτήσουν ε, αποκλειστικά δικαιώματα για την μεταφορά στο ψηφιακό περιεχόμενο υλικού, όπως σε παραδείγματι πίνακες του 17ου αιώνα που μπαίνουν σε αποκλειστικά δικαιώματα ορισμένων ε, φορέων ε, προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσης δεν πρέπει να περιορίζεται η δυνατότητα για ανείχνευση, για data mining δηλαδή του υλικού. Το copyright, για να καταλήξω, είχε σαν στόχο να εμποδίσει την χρήση του υλικού και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αυτά και ευχαριστώ. ε, οι συνάδελφοι διερμηνείς μας είπαν από την καμπίνα τους ότι είχατε ξεπεράσει την ταχύτητα του ήχου κατά 4 5 φορές. Ε, τέλος πάντων, όπως μπορέσαν τα καταφέρανε, ο κύριος Τρογεύης και έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ένα ερώτημα και ένα σχόλιο. Ερώτημα. Όσον αφορά την απόφαση του Κοινοβουλίου. Πριν από 8-9 χρόνια, όταν το copyright παρατάθηκε στα 70 χρόνια. Κάποιοι μάλιστα θεωρούσαν ότι πρέπει να διατηρηθούν τα 50, άλλοι λέγανε 60, 90 χρόνια. Τέλος πάντων στα 70 το οριστικοποιήσαμε. Τότε φαινόταν ότι θα υπάρξουν ωφέλη από αυτή την απόφαση, τα οποία όμως δεν εμφανίστηκαν ποτέ. Οι επιχειρήσεις ήταν αυτές που ωφελήθηκαν, οι επιχειρήσεις διανομής πολιτικών αγαθών. Αναρωτιέμαι λοιπόν ποια είναι η δική σας θέση σχετικά με αυτήν την παράταση των πνευματικών δικαιωμάτων, τη ισχύω των πνευματικών δικαιωμάτων. Πιστεύετε ότι πρέπει να επιμείνουμε, ε, να μην παραταθούν έτσι περαιτέρω ε, τα πνευματικά δικαιώματα. Όσον αφορά την πολιτιστική κληρονομιά, το βασικό μας μέλημα είναι αυτή τη στιγμή να ε, επιλύσουμε διαμάχες ε, απεικόνησης ε, εκθεμάτων ή μνημείων. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο όγκος, για παράδειγμα, επίσης ευρωπαϊκών ταινιών λόγω περιορισμών πνευματικών δικαιωμάτων. Το ίδιο αφορά και φωτογραφίες ή από την Ισπανία, για παράδειγμα, ή συγγραφέα από την, ε, ε, Βρετανία και εκδότη από τη Γερμανία. Είναι δύσκολα αυτά να, να, να μπορεί κανείς να, να παράγει ένα ευρωπαϊκό πολιτιστικό αγαθό όταν υπάρχουν τόσοι περιορισμοί όσον αφορά ε, το copyright. Κυρία Κόλλινς, για το πρώτο ερώτημα πιστεύω πραγματικά ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου οι παραγωγοί θα αμείβονται. Διότι αν δεν αμείβονται δεν θα παράγουν και πολιτιστικό ε, προϊόν στο μέλλον. Χρειάζεται να μπορούν να ζήσουν. Νομίζω ότι 70 χρόνια είναι πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ειδικά στον σημερινό, στο σύγχρονο κόσμο. Ε, ζούμε σε μια εποχή όπου οι οι εξελίξεις τρέχουν με ραγδαίους ρυθμούς. Σε 70 χρόνια μου φαίνονται πάρα πολλά. Δεν έχω ακριβώς πολύ... Δεν ξέρω πώς, ποιο, ποιο, ποια ακριβώς θα μπορούσε να είναι η λύση. Δεν έχω συγκεκριμένη άποψη. Θέλω όμως να εξασφαλιστεί αυτή η, η αρχή ότι τα... τα ε, αγωθ αγαθά θα μπορούν να είναι προσβάσιμα στον κόσμο. Υπάρχει δυνατότητα ψηφιοποίησης και αυτό που ε, υπάρχει πραγματικά τεράστιο χάσμα ε, ως προς την πρόσβαση σε πολιτιστικά αγαθά του 20ου αιώνα. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να δουν φωτογραφίες ή τέλο πάντων άλλο υλικό από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από τη δεκαετία του 60. Αυτό το υλικό πρέπει να γίνει προσβάσιμο. Για το δεύτερο ερώτημα. Είναι πρόβλημα βεβαίω να προσανατολιστεί και να πλοηγηθεί κανείς ε, σε όλα, αυτά τα δικαιώματα. Νομίζω ότι ε, δεν, νομίζω ότι το κάθε αρχείο ή ο κάθε παραγωγός ε, δεν θέλει να διατίθεται το περιεχόμενό του. Προφανώς και θέλει. Και χρειάζονται συγκεκριμένα πλαίσια. Πολλές φορές όμως η, η εικόνα που βρίσκεται μέσα σε μια ε, ταινία θα πρέπει να έχει λάβει άδεια προκειμένου να μπορεί να διατεθεί η ταινία αυτή σε μια άλλη επικράτεια. Ε, ο μηχανισμός που αναφέρατε είναι ε, θετικός, ωστόσο δεν είναι πανευρωπαϊκός. Άρα το πρόβλημα είναι δομικό, είναι διαρθρωτικό και πρέπει να βρούμε μια λύση για το πώς θα το ξεπεράσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Χέλγα Τρούπελ. Ευχαριστώ Πέτρα. Ευχαριστώ την Ζιλ Κάζινς. ξέρετε ότι υποστηρίζω την Ευρωπαϊάν, εδώ και πολλά χρόνια πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ένα τέτοιο οργανισμό και να μην ε, τα αφήνουμε όλα στην Google και σε άλλες μεγάλες εταιρείες. Θέλω όμως να σας θέσω ένα ερώτημα σχετικά με το copyright ως φραγμό ε, στην πρόσβαση. Άμα το δείτε από την σκοπιά της διανομής είναι αλήθεια. Αλλά πρέπει να δούμε και την πλευρά της παραγωγής. Το είπατε και εσείς. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα παράγεται νέο περιεχόμενο και ότι θα αμείβονται όλοι οι παραγωγοί, οι δημιουργοί, διότι διαφορετικά δεν θα έχουμε περιεχόμενο σε λίγα χρόνια. Αυτή είναι η βασική αντίφαση ε, που υπάρχει και είπατε βεβαίως ότι δεν, είστε, ε, δεν αντιτάσσεστε στην, ε, στο να αμείβονται οι δημιουργοί, Ωστόσο πρέπει να εξασφαλίζεται και η πρόσβαση ε, των ε, πολιτικών κέντρων, ιδρυμάτων. Και είπατε να πληρώσουν οι προπολογισμοί. Δεν είναι ότι δεν το συμμερίζομαι αυτό. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα στους προϋπολογισμούς. Ε, ούτε για το Ευρωπαίνα, ούτε για άλλα πολιτιστικά ιδρύματα υπάρχουν επαρκή χρήματα στους προπολογισμού. Άρα, αυτό που κρατώ από αυτά που είπατε είναι ότι θα πρέπει να υπάρξουν ε, ευφυείς, αποτελεσματικές λύσεις, οι οποίες όμως για μένα ε, πρέπει να λαμβάνουν ιδιαίτερο υπόψη τους παραγωγούς. Εμείς ε, επιμένουμε πάντοτε να... η κοκακόλα να πληρώνει τους εργάτες της. Ε, το ίδιο πρέπει να αμείβονται και οι δημιουργοί. Θέλουμε να υπάρχει πρόσβαση, αλλά η πρόσβαση αυτή δεν μπορεί να είναι δωρεάν για όλους και πρέπει να βρούμε ε, τρόπο να, να ξεπεράσουμε αυτό, αυτή την αντίφαση. Το ίδιο ισχύει και για το geo-blocking, για το γεωγραφικά αποκλεισμό. Δεν είναι δυνατόν να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια πανευρωπαϊκή πρόσβαση στι ευρωπαϊκές ταινίε και τελικά αντί για αυτό να κατα... καταλήξουμε να σκοτώσουμε την ευρωπαϊκή βιομηχανία κινηματογράφου. Φυσικά, ε, οι Ευρωπαίοι παραγωγοί δεν θέλουν να μην διανέμεται το προϊόν τους, θέλουν να διανέμεται, αλλά θέλουν και να αμείβονται με δίκιο τρόπο. Ευχαριστώ. Κυρία Κάζινς, έχετε το λόγο, παρακαλώ. συμφωνώ με αυτό που είπατε και σχετίζεται και με το προηγούμενο ερώτημα. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα αμείβονται με δίκαιο τρόπο οι δημιουργοί. Το copyright δημιουργήθηκε μεταξύ άλλων και για αυτόν τον σκοπό όχι για να ε, το επεκτείνουμε πέραν των 70 ετών, ούτε για να δημιουργήσει εμπόδια, ώστε να μην μπορεί κανείς να, να χρησιμοποιήσει ένα περιεχόμενο ή ένα πολιτιστικό αγαθό, εφημερίδες, ε, φωτογραφίες κτλ. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός δημιουργίας του. Άρα πρέπει με κάποιο τρόπο να βρεθεί ένας συμβιβασμός και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να είναι τέτοιο συμβιβασμό. Και επίση πιστεύω ότι τα ε, Ιδρύματα Πολιτιστικής Κληρονομιάς παρέχουν αυτό το υλικό Ακριβώς γιατί ε, είναι απαραίτητο για την εκπαίδευση, για τις δημιουργικές βιομηχανίες. Ε, υπάρχει τεράστια ζήτηση η οποία δεν μπορεί να καλύπτεται γιατί, γιατί τη χρειάζονται σε συγκεκριμένο επίπεδο ποιότητας ή μπορεί να χρειάζεται να, να, να είναι απαραίτητο ένα συγκεκριμένο υλικό, μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδου. Άρα χρειάζεται να ψηφιοποιηθεί όλο αυτό το υλικό ε, και αυτό απαιτεί χρήματα. Και Ωστόσο, Νομίζω ότι ευθύνονται τα πολιτικά ιδρύματα και για το γεγονός ότι ε, καταχρώνται αυτά τα, τα το, το, τη δημόσια σφαίρα. Ε, για το γεγονός ότι υπάρχουν αγαθά τα οποία θα έπρεπε να βρίσκονται στη δημόσια σφαίρα, να είναι κοινή ε, κτήση όλων των ανθρώπων και ταυτόχρονα αυτά τα ιδρύματα είναι εκείνα που θέτουν ε, φράγμους. Ευχαριστώ. Και εγώ ένα ερώτημα να θέσω, λέει η Πρόεδρος. Είπατε ότι πολλές φορές το θέμα δεν είναι αν μπορεί κανείς να πληρώσει τα δικαιώματα, αλλά και ότι είναι δύσκολο και δαπανηρό να προσδιοριστεί ποιος τελικά ε, δικαιούται τα χρήματα από τη χρήση ενός πολιτικού αγαθού. Είπατε ότι αυτό το Extended Collective Licensing System ε, που υπάρχει στη Σκανδιναβία ε, και που λειτουργεί εκεί καλά θα μπορούσε να είναι μια λύση ή τέλο πάντων που μπορεί να έχει οδηγήσει ε, στην ικανοποίηση όλων των πλευρών. Θα, μπορούσατε, θα μπορούσε κατά τη γνώμη σας ένα τέτοιο σύστημα να εφαρμοστεί σε ολόκληρη την Ευρώπη και αν ναι θα μπορούσε μέσω αυτού του συστήματος να απλουστευτεί τουλάχιστον το καθεστώς ε, γύρω από τα δικαιώματα. Κοιτάξτε, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, το copyright, δεν είναι αρμοδιότητά μου. Νομίζω ότι το Extensive Collective Licensing, οι επεκταταμένες αδειοδοτήσεις οι συλλογικέ είναι καλό πράγμα, αλλά πρέπει να έχει πρακτικές εταιρείε που να λειτουργούν σωστά. Ε, και ε, σε όλες τις χώρες δεν φαίνονται να είναι ε, αξιόπιστες. Άρα αυτό δεν δουλεύει ούτε για τους δημιουργούς, ούτε για αυτούς που προσπαθούν να εισπράξουν τα δικαιώματα που, του, που δικαιούνται. Χρειάζεται χρόνος για να δημιουργηθεί αυτός ο μηχανισμός. Είναι καλό μοντέλο, καλό, είναι να εξαπλωθεί, αλλά η επιτυχία του εξαρτάται από πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες. Ναι, πριν από λίγο καιρό είχαμε προσπαθήσει να διαρευνήσουμε το θέμα των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων Πρέπει να κοιτάξουμε βέβαια τι απήχηση είχε και τις προσέφερε. Αν παραμένουν τα προβλήματα ως προς τις ε, ε, υπηρεσίες διαχείρισης. Η κυρία Κώστα. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και ενημερωτική τοποθέτησή Σα Η Ευρωπαϊκή ε, κάνει πολύ καλή δουλειά για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Παραμένει για μένα το θέμα της προσβασιμότητας και της ανταμοιβή βεβαίω ε, τη δημιουργική δουλειά, αλλά και τη επιστημονική πάντα. Δεν μιλούμε μόνο για δημιουργική καλλιτεχνική δουλειά. Θέλω επίση να αναφερθώ στην ε, μεταρρύθμιση και τις προτάσεις που έχει υποστήριξει και δική μας η Επιτροπή για εξαιρέσεις που αφορούν ε, αντίγραφα όταν υποκείμενο είναι ένα ε, ένας φορέας πολιτιστικός, βιβλιοθήκες κτλ, ακόμη και ψηφιακά, σε αντιπαράθεση με τους εμπορικούς, με την εμπορική εκμετάλλευση. Εκεί βλέπετε εσείς κάποια διαφορά σε σχέση με τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορεί να αποτελέσει δηλαδή αυτό ένα βήμα. Και η μεταρρύθμιση που έγινε σε σχέση με την προσβασιμότητα σε ε, ορφανά, όπως τα λέμε, έργα εκείνα των οποίων είναι δύσκολο να ανεβρεθεί ο δικαιούχος και για τα οποία μία οδηγία επιτρέπει μία πρόσβαση. Σας ικανοποιεί? σε σχέση με, αυτό με αυτή τη δυνατότητα, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή, αλλά για οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή, ε, να χρησιμοποιεί κατά τρόπο παράνομο το περιεχόμενο αυτό επίσης είναι κάτι που με απασχολεί. Δηλαδή κάποιος που να μπορεί να, κάνει, να, να, ξουπίσει υλικό που εσείς διαθέτετε για, λόγους, για σκοπούς παράνομους. Απάντηση. Ναι, προχωρούμε προς την ορθή κατεύθυνση πιστεύω μένα. Εάν όμως δεν πραγματοποιηθεί το επιπλέον βήμα, δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα της παρέκκλησης ως εναλλακτική αν ε, δεν δίνονται λύσεις ε, από τις άλλες προτάσεις γιατί όλα καλά είναι επέκταση ε, του συστήματος της αδειοδότησης κτλ. Αλλά ταυτόχρονα θέλουμε και μια εναλλακτική για τις χώρες οι οποίες δεν έχουν συλλογικές, συλλογική διαχείριση αδειών ή για όσα έργα δεν καλύπτονται από αυτά. είναι πολύ συχνά, ιδιαίτερα στο εφήμερο πολιτιστικό υλικό, φανταστείτε μια κάρτα ποστάλ, μια φωτογραφία που έχει βγάλει κάπως, όπου δεν είναι δυνατόν να ανεβρεθεί ο δικαιούχος. Τώρα για τις άλλες ερωτήσεις σας τις ξέχασα. Ναι, δύο ερωτήσεις είχα ακόμα. Αν συμφωνείτε με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας που επιτρέπει την παρέκκληση, μια νέα δυνατότητα για παρέκκληση λοιπόν, και δεύτερον, όρφανα έργα που ήδη έχουν εγκριθεί ως δυνατότητα για δημοσίευση έργων που εντός εισαγωγικών ονομάζονται ορφανά. Αυτή είναι η καινοτομία. Τι έχετε να πείτε. Κοιτάξτε για τα ορφανά έργα. Το θέμα που έχουμε στην οδηγία αυτή είναι ότι πρώτον καλύπτει πολύ περιορισμένο όγκο υλικού, αριθμό έργων. Δεν είναι τόσο πολλά τα έργα. Είναι πάρα πολύ μικρός όγκος, όπως σας δείχνω, και άρα χρειαζόμαστε να χρειάζεται να καλυφθεί όλο το υλικό και όχι μόνο τα ορφανά έργα. Η Πρόεδρος ευχαριστώ και βέβαια τα έργα τα οποία πια δεν είναι στο εμπόριο δεν καλύπτονται από την νομοθεσία για τα ορφανά. Ο κύριος έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μια ερώτηση γιατί ήταν πολύ εύστοχη αυτή της κυρίας Τρούιπελ και θα ήθελα να επανέλθω για τη μελέτη, αν μου επιτρέπετε. Για τον κύριο Αλμέντα. Να τα πω στα ισπανικά τώρα. Για αυτή τη μελέτη είχα λίγο χρόνο και εγώ είχα λίγο χρόνο να τη δω μας δίνει υποδείξεις και προτάσεις. Δεν θέλω να μιλήσω για τις υποδείξεις και προτάσεις για τις δημόσιες δαπάνες. Έχετε προβλέψεις όμως για το μέλλον. Κάποιες εκφράσεις που συνάδαν με αυτά που έχει πει ο κύριος Γιούνκερ. Το βλέ... Τις βλέπουμε. Έχετε κάποια κόκκινη γραμμή θα υπάρξει πρόβλημα στο μέλλον αν δεν τα καταφέρουμε όλα. Ή υπάρχουν άλλα στοιχεία που δείχνουν άλλες κόκκινες γραμμές για εσάς. Τι θα συμβεί στο μέλλον δηλαδή αν δεν τα καταφέρουμε αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για να δούμε αν θα τα καταφέρετε μέσα σε δύο λεπτά. Κοιτάξτε, το να εμφανίζεται κανείς σε μια επιτροπή του και ο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει να κάνει με τον πολιτισμό ε, και σημαίνει ότι πρέπει να πει ξεκάθαρα και να παραδεχθεί ότι είναι δραματικό το γεγονός ότι η Ευρώπη είναι δύο ταχυτήτων σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στο προ... στον πολιτισμό. Πού ε, είναι η πρόσβαση η κουλτούρα, ο πολιτισμό πρέπει να είναι στρατηγικός άξονας του ευρωπαϊκού προπολογισμού. και αυτή τη στιγμή δεν έχει αυτή τη θέση. Αυτό είναι κάτι το δραματικό και πρέπει να το τονίσουμε ξανά και ξανά. Για κάθε ευρώ που επενδύεται στον πολιτισμό είναι τεράστια η επιστροφή στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αυτής της χώρας που το επενδύει και στο σύνολο της Ευρώπης. Και υπάρχουν ένα σωρό μελέτες που το αποδεικνύουν αυτό. Η συνεισφορά του πολιτισμού στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ υπολογίζεται και είναι της τάξης του 4-4,5%. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει ότι θα είναι βασικός στρατηγικός άξονας η καινοτομία, η κοινωνία της γνώσης, από τη στιγμή που τα αποφασίζει αυτά, η κουλτούρα, ο πολιτισμός είναι θεμελιώδη ζητήματα. Αυτή τη στιγμή συνειδητοποιούμε ότι στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό η κουλτούρα, ο πολιτισμός είναι κάτι το περιθωριακό, το ελληματικό αν θέλετε, το παραμελημένο. Αισιόδοξη ερμηνεία είναι να πούμε ότι υπάρχει τεράστιο περιθώριο βελτιώσεων. 0,70% είναι το βάρος του προϋπολογισμού για τα θεσμικά όργανα π.χ. Να, να προσδιορίσουμε λοιπόν να φτάσει στο 1% ή να το ξεπεράσει αν 0,70% είναι αυτό που αφιερώνεται στον πολιτισμό. Εάν τώρα με απόλυτους αριθμούς αυξηθεί ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, τότε θα πρέπει να υπάρχει αυτονομία και η κουλτούρα και ο πολιτισμός να, να αντιστοιχηθούν με το 3 ή 4% ε, του ε, προϋπολογισμού. Υπάρχει τεράστιο περιθώριο βελτίωσης, να δημιουργηθούν νέα εργαλεία, νέες πολιτικές, να ενοποιηθεί ο φόρος προστιθέμενης αξίας, να υπάρξει η ιδέα της ε, των μεκίνων και των χορηγών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πολιτιστικών δηλαδή, με τους πολιτιστικούς μεκίνες. Ε, μας εκπλήσει πολύ αυτή η μελέτη, κάτι το οποίο είναι βασικό για το μέλλον, για την ταυτότητα του προγράμματος πολιτισμού είναι κάτι που είναι παραμελημένο και δεν, το, δεν του δίνει καμία ε, σημασία η Ευρώπη. Όταν έχουμε πραγματικά ευρωπαϊκό πολιτισμό, έχουμε πολίτες με κριτική σκέψη, με δυνατότητες ε, ε δημιουργίας, παραγωγής, έχουμε μια πιο δημοκρατική κοινωνία. Εάν ε, αυτό δεν γίνει, τότε το ευρωπαϊκό όραμα θα κινδυνεύσει και θα συγκλονιστεί έτσι όπως έχει συμβεί και τα τελευταία χρόνια και το βλέπουμε όλοι. Ευχαριστώ. Καλώς, ευχαριστώ πολύ και περνούμε στον επόμενο ειδικό τον κύριο Μούσου από τον Ποζάχ. Ένα κέντρο πολιτισμού, θα πω, το οποίο κάνει μεγάλες προσπάθειες και συμμετέχει σε πολλά project για τη διευκόλυνση και της πρόσβασης στο πολιτιστικό περιεχόμενο και όντως εξασφαλίζει αυτή την ε, πρόσβαση για πολλούς πολίτες. Έχετε το λόγο. Χαίρετε και καλησπέρα. Δουλεύω για το Μποζάρ, το κέντρο τεχνών στις Βρυξέλλες, θα το έχετε ακούσει ίσως. Και δεν ήξερα όταν μου ζητήθηκε να έρθω αν θα πρέπει να μιλήσω για το οικονομικό μοντέλο, για το πώς προσεγγίζουμε το κοινό μας. Διαφορετικά πράγματα, αλλά θα προσπαθήσω να τα κάνω και τα δύο. Ας μιλήσω λοιπόν πρώτα για το μοντέλο μας. Ευρωπαϊκό σπίτι της κουλτούρας, του πολιτισμού, όπως θέλουμε, ένα υβριδικό δηλαδή μοντέλο, αλλά να μιλήσω και για τις τέχνες, κυρίως τις οπτικές, γιατί θα μπορούσα να μιλήσω και για αρχιτεκτονική και για μουσική, αλλά και τις ε, ε τέχνες θέλω να ε, αναφέρω ιδιαίτερα και τι θα μπορούσε να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το Μποζάρ. Θα το έχετε δει, ίσως θα το έχετε επισκεφθεί, δεν είναι και μακριά από εδώ. Ένα χαρακτηριστικό κτίριο του Βικτόρ Ορτά σε αρτεκό τέχνη του μεγάλου Βέλγου ε, αρχιτέκτονα είναι πολιτιστικό project από το 2002 κέντρο των καλών τεχνών ομοσπονδιακό με ένα κομμάτι του κύβεσματος που αξιοποιούμε μόνο εμείς και το όλο το, το οποίο το εκμισθώνουμε για διάφορες εκδηλώσεις. Ξέρετε ότι συνεργαζόμαστε παραδείγματι με προεδρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συνόδους, κορυφής, για συνομιλία και επαφές με νέους, με ομογενείς, με πρόσφυγες. Πολλά είναι λοιπόν τα σύμβολα τα οποία μεταφέρουμε ως μήνυμα για την Ευρώπη, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει πάντα στα κέντρα τέχνης στην Ευρώπη, γιατί δεν είναι και τόσο κοντά στα θεσμικά όργανα όσο εμείς. Κάποια στοιχεία, πολύ σύντομα, ένα εκατομμύριο επισκέπτες, ένας μέσος όρος ε, αντίστοιχα πόλεων με, με αντίστοιχο πληθυσμό, Έχουμε 250 εργαζομένους και θέλω αυτό να το τονίσω. Γιατί έχουμε τεχνικού ήχου, έχουμε σκηνογράφους, άλλο τεχνικό προσωπικό που εμπλέκεται στις δραστηριότητες μας και αυτό έχει τεράστια και οικονομική σημασία. Κάποια στοιχεία, κάποιες εικόνες για τις υποδομές μας, ίσως δεν είναι τόσο ευκρινείς. Έχουμε αίθουσες ε, κινηματογραφικών προβολών, συναυλιών και ο Βικτόρ Ορτά εδώ, ο αρχιτέκτονας που έχτισε το, στη δεκαετία του 20 το κτίριο. Υβριδικό λοιπόν οικονομικό μοντέλο, ιδιωτικός και δημόσιο τομέα, διαφορετικά εισόδηματα, με τις πωλήσει, ε, η έσοδα καλύτερα με τις πωλήσει των ε, εισιτηρίων, την υποστήριξη από το κοινό, ε, δωρεές μεμονωμένες, χορηγίες από επιχειρήσεις, ιδρύματα και το καθεξής. 50% από το εισόδημα μας είναι από την υποστήριξη την κρατική. Ιδιαίτερα στις υποδομές μας πάει αυτό. Σημασία μεγάλη δίνουμε και στις συμπαραγωγές, 5 εκατομμύρια το χρόνο αποκομίζουμε από συμπαραγωγές με Ευρωπαίους και διεθνούς εταίρους, και επίσης έχουμε ως έξοδο την ε, συντήρηση του κτηρίου. Μια τεράστια επένδυση τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δέκα χρόνια για να προστατέψουμε αυτό το συντηρητέο κτίριο. Είναι πολύ μεγάλες οι απαιτήσει για την ε, ε, συντήρησή του, ακόμα και για μια χώρα όπως το Βέλγιο. Βλέπετε εδώ λοιπόν μια γενική εικόνα του οικονομικού μας μοντέλου, 50% όπως είπα δημόσιοι πόροι, βελγική, τοπική και ευρωπαϊκή, πωλήσει ε, εισιτηρίων και θέλουμε περισσότερο να αξιοποιήσουμε ευκαιρίες για μια απαλλαγή φορολογική που μέχρι πριν από δύο χρόνια ίσχυε για τον κινηματογράφο, τώρα και για τις ε, τέχνες όπως ο χορός, η μουσική και τα λοιπά, performing acts, αλλά θέλουμε να επιδιώξουμε την επέκταση και σε κάθε άλλη μορφή τέχνες. Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση έχει μεγάλη σημασία, όχι μόνο ως προς τον όγκο, αλλά και για την υποστήριξη που μας δίνει σε εταιρικέ συνεργασίες διασυνοριακές. Ιδιαίτερα θέλω να σας δείξω αυτήν τη διαφάνεια για τον νέο ρόλο των τέχνης στον 21ο αιώνα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε και κοινωνικές προκλήσεις πλέον με τον μετανάστες, πρόσφυγες. Είναι κοινωνικός ο ρόλος που καλούμαστε να υπηρετήσουμε στην ενίσχυση της δημοκρατίας αλλά και στην αφύπνιση των πολιτών. Μπορούμε να πούμε ότι ίσως είμαστε από τα λίγα κέντρα που προσφέρουν ως κτίριο τη δυνατότητα για την οικοδόμηση κοινωνικού ιστού με τις επαφές και τις ε, πολυτομεακές πλατφόρμες ε, επαφής μεταξύ πολιτών, αρμόδιων για λήψη αποφάσεων, καλλιτεχνών, ε, πανεπιστημιακών δασκάλων. Και εδώ βέβαια έρχεται και ο εκπαιδευτικός ρόλος που έχουμε αναλάβει για συγκεκριμένα τμήματα πληθυσμού, αλλά και για ομογενείς Έχουμε δει παραδείγματι οι καλλιτέχνες ε, των διαφόρων εκπροσωπουμένων στην ε, Ευρώπη, στο Βέλγιο και τη Βρυξέλλες συγκεκριμένα ομογενών ε, ή αποδήμων καλύτερα καλλιτεχνών. Από την Αφρική ιδιαίτερα έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση στου καλλιτέχνε από την Αφρική. Νέα πρόκληση λοιπόν τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί γιατί πρέπει και αυτό το ρόλο να αναλάβουμε και να υπηρετήσουμε και νομίζω ότι μας συναρπάζει όλους. Ιδιαίτερα η γνώση η δημιουργία ευρύτερης ευφυΐας και λύσης. Προσφέρουμε δηλαδή τη δυνατότητα για ανάπτυξη ευφυΐας για το ευρύ κοινό και να προσφέρουμε λύσεις ε, για τις ε, προκλήσεις της εποχής. Αυτό νομίζω ότι είναι μια γενικότερη συζήτηση για το ρόλο της τέχνης στην ιστορία, αλλά είναι μια άλλη συζήτηση. Εδώ ήθελα να φέρω τα μαθήματα που έχουμε αναπτύξει. Όλα Φουρέλια Σον είναι ο παραγωγός των σχέσεων με το Βερολίνο, με το Ελσίνκι και με άλλες πόλεις συνεργαζόμαστε. Τώρα στις προκλήσεις έχουμε την εκρηκτική αύξηση των καλλιτεχνών, καλλιτεχνικών έργων, κινητικότητας. Έχουμε περί τα 30.000 και περισσότερα μουσεία στην Ευρώπη, αναδιόμινες ε, καλλιτεχνικές σκηνές, ευρωπαϊκά έργα που προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε. Ε, όλοι αυτοί οι νέοι καλλιτέχνες που βγαίνουν από τις ε, σχολές καλών τεχνών χωρίς πρόσβαση στο εγκαθιστική απροβολή της τέχνης πρέπει και αυτοί να υπηρετηθούν και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε μεταξύ άλλων. Ε, ανταγωνισμός ε, μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης. Το βλέπουμε και στο έργο Creative Europe. Έχει όλο και μεγαλύτερη σημασία και για μας. Είναι και θέμα ευθύνη να συνεργαζόμαστε με, με φορούς από τη Δυτική, την Ανατολική Ευρώπη, τα Βαλκάνια. Είναι θέμα δέσμευσης για μας και στράτευσης. Και βέβαια και ο διαγωνισμός ή ο ανταγωνισμός μεταξύ μικρών, μεγάλων, μουσείων, νεοαφιχθέντων, νεο, νέα, νέο μουσείο στο Παρίσι, συλλογές, ε, κάποια που δεν έχουν συλλογές, όπως και είπα, κυρίως οι οικαστικές. Για ένα-δύο οι οικαστικές τέχνες ε, παίρνουν ε, τραβούν το ενδιαφέρον μας στην υπόθεση αυτή. Και βέβαια, μικρές και μεσές αστικές περιοχές και περιοχές της υπαίθρου είναι ένα ιδιαίτερο σημείο εστίασης για τις δραστηριότητες μας και όχι μόνο επειδή είμαστε στις Βρυξέλλες. Τώρα, μια, ε, πρακτική, ένα πρακτικό θέμα που θα ήθελα να συζητήσουμε εδώ. Κρατικές εγγύησεις μπορούν να χρήσιμο δηλαδή για τη δουλειά σας κρατικές εγγυήσεις και για την ε, πολιτιστική κληρονομιά και για τις οικοστικές τέχνες. Προσωρινές εκθέσεις λοιπόν, οι οποίες μπορούν να κοστίσουν από 1 έως 3 εκατομμύρια. Το κόστος της εγγύησης έχει διωγγωθεί τα τελευταία 30 χρόνια. Μπορεί να φτάσει στο 20 40% του κόστους μιας έκθεσης. Πράγμα το οποίο πιέζει πολύ βέβαια τα μουσεία που δεν έχουν επαρκεί οικονομικού πόρου. Κρατικέ εγγυήσει κρίσιμε για τη μείωση του κόστου στο Ηνωμένο Βασίλειο τη Γαλλία, ενώ υπάρχουν 17 χώρες οι οποίες δεν προσφέρουν κρατικές εγγύσει. Αυτά είναι στοιχεία της ε, μελέτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2003 για το ζήτημα αυτό. Δεν έχω δει εντωμεταξύ κάποια πιο επικαιροποιημένη μελέτη. Εμείς στο Βέλγιο δεν ε, γνωρίζουμε κρατικές εγγύησεις για τις εκθέσεις. Μάλιστα πολλές από αυτές ε, απορρίπτονται ως εγγύησεις από τους από τις τράπεζες, από τους δανειοδότες και τίποτε δεν έχει παρουσιαστεί πρόβλημα. Είναι σπάνιο να χρειάζεται να καταπέσει η εγγύηση. Είναι μικρός ο κίνδυνος δηλαδή. Έτσι λοιπόν χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση, εναρμόνιση, εμπιστοσύνη, διάδοση του συστήματος των εγγύησεων, των κρατικών εγγύησεων, ε, είτε ως ευρωπαϊκό παιδό ή παγκόσμιο, είτε σε έκφραση υποστήριξης προς τα εθνικά προγράμματα εγγύσεων για την τέχνη. Στις προκλήσεις, πρόκληση για μας βεβαίως για τις σύγχρονες τέχνες, ε, γιατί έχουμε μείνει σε μια λογική του λευκού κύβου ως λογική για τη σύγχρονη τέχνη. Πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο, να προσελκύσουμε περισσότερο το κοινό μας να προσφέρουμε περισσότερη κοινωνική καινοτομία, ε, ανοιχτό πνεύμα για σχεδιασμό, για δημιουργία, για φαντασία. Να, εδώ ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα την επόμενη εβδομάδα. Αφροπόλιταν το φεστιβάλ μας. Σας καλούμε να είσαστε όλοι παρόντες. Πρόκειται για τέχνη από την Αφρική. Και συνεχίσω σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ειδικέ ανάγκες ε, για τις οικαστικές τέχνες που ίσως δεν αναφέρονται ρητά ως προτεραιότητα στο πρόγραμμα Creative Europe μας ξαφνιάζει αυτό βεβαίως, έχει πολύ μεγάλη σημασία ε, μειωμένη είναι η παρουσία των σχεδίων για οικαστικές τέχνες στο Creative Europe και συγκεκριμένα το που διεκδικούμε κάθε πέντε χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μακροπρόθεσμος στόχος πρέπει να παραμείνει, το, τον υποστηρίζουμε, συμφώνουμε μαζί σας, η... ο πολιτισμός στην Ευρώπη και οι εξωτερικές σχέσεις, νέα προτεραιότητα, ε, δυνατότητα για ε, υποψηφιότητες από, μη, από χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, μικροί και μεγαλύτεροι φορείς ή παράγοντες στην τέχνη, ε, οικονομική αλληλεγγύη, υποστήριξη, ισορροπίες μεταξύ Βορρά, ε, Νότου, Ανατολής, Δύσης και ένα ευρωπαϊκό σύστημα κρατικών εγγύσεων για τις Εικαστικές τέχνες. Και βέβαια η διασύνδεση με τα άλλα προγράμματα, τα ΕΦΚΟ, Horizon και ούτω καθεξής. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επισκόπηση που μας δώσατε σχετικά με το έργο του Μποζάρ και ποιες θεωρείτε ότι θα προκλήσεις για το, για το, για το μέλλον. Το λόγο στον κύριο Στρογεύσκη. Ευχαριστώ πολύ. Με μεγάλη ικανοποίηση. Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησα τα λεγόμενά σας όταν ήμουν υπουργό πολιτισμού στην Πολωνία και εγώ είχα θέσει αυτό το θέμα της ασφάλισης και των ασφαλίσεων, υπάρχει ανισορροπία. Υπάρχουν χώρες που εγγυώνται την ασφάλιση και άλλες χώρες που δεν το εγγυώνται σε τέτοιου είδους καταστάσεις και σε τέτοιου είδους ανταλλαγές μεταξύ μουσείων. Και είναι δύσκολο αυτό. Ξέρω τον Μποζάρ πολύ καλά, ε, το έχω επισκεφθεί επανειλημμένος. Κατά τη διάρκεια της πολωνικής προεδρίας Είχαμε διάφορες ε, δραστηριότητες και θυμάμαι μια περιγραφή που ήταν εξαιρετικά δύσκολο να κάνει κανείς αποδεκτή. Στις οπτικές τέχνες, στις οικαστικές τέχνες έχουμε ε, όλο και μεγαλύτερο κενό μεταξύ αυτών που είναι καλοί σε αυτές και αυτών που δεν είναι καθόλου καλοί. Όσοι είναι καλοί γίνονται καλύτεροι και όσοι δεν έχουν επαφή απομακρύνονται ε, όλο και περισσότερο από αυτού του είδους την οικαστική και καλλιτεχνική έκφραση. Το Μποζάρ ήθελε να προσφέρει πρωτοποριακά εκπαιδευτικά προγράμματα σε νέους και σε παιδιά, πειραματικά. Το καταφέρατε αυτό, ε, καταφέρατε να ενισχύσετε την προσφορά την εκπαιδευτική, να υπάρχει καλύτερη πρόσβαση και συμμετοχή στα έργα πολιτισμού. Ευχαριστώ. Μπορώ να μιλήσω γαλλικά. Κοιτάξτε, είτε μεγάλη η πρόκληση εδώ και πάρα πολλά χρόνια και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε αυτή. Εξαρτάται από το κοινό για το οποίο μιλούμε. Υπάρχουν ακροατήρια πολύ πιο ενεργητικά, πολύ πιο δραστήρια. Υπάρχουν άλλα μέλη του κοινού που περνούν μπροστά από το κτίριο και δεν ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια προσπαθούμε να βγούμε εκτός των τυχών, να δουλέψουμε μέσα της τάξης. Έχουμε ε, την εβδομάδα της μουσικής της Βρυξέλλης, εκεί οργανώνουμε συναυλίες. Θέλουμε να διευκολύνουμε την πρόσβαση και να φτάσουμε ε, σε ένα κροατήριο που από μόνο του δεν θα ερχόταν και δεν θα πατούσε το πόδι του μέσα στο Μποζάχ. Επίσης μεγάλο, μεγάλη πρόκληση για τα σύγχρονα κέντρα ε, τα ευρωπαϊκά τέχνης είναι να κατοχυρωθούν θεσμικά, να το κάνουν αυτό και δηλαδή να συμμετέχει περισσότερο το κοινό, να θεσμοθετηθεί αυτή η συμμετοχή, να συμμετέχει όχι μόνο στις ε, εκθέσεις, αλλά να υπάρχει μια τακτική πρόσβαση, μια ροή, πρόσβαση σε άτομα επίσης μειωμένης κινητικότητας, και ελπίζουμε με ορίζοντα το 2020 να έχουμε καλά νέα για τον ορίζοντα 2020 για το πρόγραμμα αυτό και θα πρέπει εκ των προτέρων να ερευνήσουμε περισσότερο ε, σε ποιο κρατήριο θέλουμε να απευθυνθούμε για να καθορίσουμε μετά τον προγραμματισμό μας. Δεν είναι εύκολο το εγχείρημα. Ο επιμελητής μιας έκθεσης συχνά θέτει στον εαυτό του το ερώτημα του ακροτηρίου και του κοινού στο οποίο απευθύνονται και κυρίως οι εικαστικές τέχνες. Ευχαριστώ. Η κυρία Κώστα παρακαλώ πολύ ενδιαφέρον. Γνωρίζω τον Μποζάρ, εκτιμώ ιδιαίτερα αυτά που κάνατε. Κάνατε μια πρόταση που θα ήθελα να επαναφέρω και βεβαίως υποστηρίζουμε το 1% για, το, για τη δημιουργική Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό. Στο ευρωπαϊκό επίπεδο ε, θα ήθελα να σταθώ την ε, ασφάλιση που θα μπορούσαμε να ορίσουμε ευρωπαϊκή, δηλαδή ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης, κινητικότητα των έργων τέχνης, ε, ε, διευκόλυνση των ε, καλλιτεχνών κτλ. Και το άλλο είναι αυτό των εγγυήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη δανειοδότηση. Είπατε, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι μπορεί να υπάρχει ένα ταμείο εγγύσεων αυτή τη στιγμή. Βέβαια δεν λαμβάνει υπόψη αυτόν τον τομέα της ε, τέχνης. Και υπάρχουν επίσης ιδιωτικά ταμεία πέραν ιδρυμάτων και άλλων που προσφέρουν διευκολύνσεις ε, οικονομικού χαρακτήρα. Δεν ξέρω ε, αν υπάρχει στο Βέλιο. Υπάρχει στην Ιταλία όμως εδώ και δύο χρόνια το Art Bonus, ένα μέσον που έχει φέρει 200 εκατομμύρια ευρώ τους τελευταίους μήνες και έτσι επιτρέπει σε ιδιώτες να επενδύσουν σε πολιτιστική κληρονομιά, θέατρα, γκαλερί, πινακοθήκες κτλ. Και να εξασφαλίσουν ταυτόχρονα και μια ε, έκπτωση φόρου. Μήπως αυτό ήταν μια λύση για να προσελκύσετε κονδύλια. Απάντηση. Κοιτάξτε, δεν είμαι ειδικό στο θέμα αυτό για τα φορολογικά, αλλά έχουμε εδώ το tax shelter, το φορολογικό καταφύγιο. Υπήρχε για το κινηματογράφο και τώρα έχει διευρυνθεί να περιλάβει και τις ε, ε, performing arts και ελπίζουμε να πάμε ακόμα, ακόμα πιο μακριά, ε, να προχωρήσουμε περισσότερο. τώρα η εγγύηση ευρωπαϊκή θα ήταν όνειρο για μας. Ε, ανακάλυψα τη μελέτη του 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 15 χρόνια έχουν περάσει. Το, η Δημιουργική Ευρώπη είναι άλλο πρόγραμμα που μπορεί να μας ενισχύσει. Θα το διερευνήσουμε για την επόμενη προγραμματική μας περίοδο. Ευχαριστούμε πολύ. Να προχωρήσουμε λοιπόν και να πάμε στον επόμενο εμπειρογνώμονά μας που ακριβώς θα ασχοληθεί με αυτά τα φορολογικά θέματα, φορολογικά εμπόδια και όλα αυτά που σχετίζονται με αυτόν τον ε, τομέα που ενδέχεται δηλαδή να αποτελούν ε, εμπόδια στην πρόσβαση στο πολιτικό ε, περιεχόμενο. Κύριε Μολυνά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα μιλήσω για φορολογικά καταφύγια. Σας ευχαριστώ καταρχάς ε, για την πρόσκληση. Θα μιλήσω για φορολογικά προβλήματα και ε, στη συνέχεια για καλλιτέχνες που κάνουν performance, όχι καστικούς, δηλαδή. Έχω και μια παρουσίαση μαζί μου. Και εκτός από την την ε, παρουσίασή μου έχω αποστείλει και ένα σημείωμα που, και ένα άρθρο που σας έχω αποστείλει και που έχω δημοσιεύσει. Ποιο είναι το πρόβλημα λοιπόν για το οποίο θα σας μιλήσω. Υπάρχει στη διεθνή φορολογία υπάρχει ένας ειδικό κανόνας για τους ε, performing artists και Ε, οι αυτοαπασχολούμενοι καλλιτέχνες εμπίπτουν στο άρθρο 7 του μοντέλου του ΟΣΑ ε, και το άρθρο 7 λέει ότι πληρώνεις μόνο φόρο στην πατρίδα σου εκτός αν έχεις τη μόνιμη έδρα σου σε άλλη χώρα και εκεί πληρώνεις επί των κερδών ε, το φόρο σου. Όταν είσαι υπάλληλο, υπάγεσαι στο άρθρο 15 των Διεθνών Συνδικών που αναφέρουν ότι ο υπάλληλο πληρώνει φόρους στη χώρα όπου διαμένει εκτός αν, μεταφέρεται, αν πηγαίνει με τον εργοδότη του σε άλλη χώρα όπου και φορολογείται. Υπάρχουν πάρα πολλά που θα μπορούσα να πω για αυτές τις ε, γενικές αρχές αν και είναι αρκετά σαφείς και δεν δημιουργούν προβλήματα. Αλλά για αθλητές και καλλιτέχνες υπάρχει ειδικό κανόνας στο άρθρο 17 που αξιοποιούν περισσότερες χώρες στις διμερείς συμφωνίες τους και ο οποίος αναφέρει ότι οι καλλιτέχνες και αθλητές φορολογούνται εκεί όπου δραστηριοποιούνται ανεξάρτητα από το αν είναι αυτοαπασχολούμενοι ή ε, υπάλληλοι. Υπάρχει λοιπόν ένας ειδικό κανόνας για καλλιτέχνες και αθλητές. Το 1963 θεσπίστηκε αυτός ο κανόνας και η εντολόγηση τότε αφορούσε ε, πρακτικά χαρακτηριστικά των ε, επαγγελμάτων αυτών. Υπήρχε για παράδειγμα ένας μποξέρ ο οποίος ζούσε στο Μονακό και δεν ε, κατέβαλε ε, φόρους ε, ούτε εκεί ούτε στη χώρα από την οποία ε, καταγόταν. Αυτά βεβαίως το 1963 και το 1987 ο ΣΑ συνέταξε μια έκθεση για αυτές τις δύο κατηγορίες ε, όπου υπήρχε έλλειψη εμπιστοσύνης. Ανέφερε η έκθεση αυτή ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα μη συμμόρφωσης, δηλαδή αληθλητές και καλλιτέχνες δεν δηλώνουν τα εισοδήματά τους από το εξωτερικό, χρησιμοποιούν συστήματα φοροαποφυγής και ε, δεν είναι ιδιαίτερα ενημερωμένοι ε, γύρω από τα φορολογικά ζητήματα. Δεν ξέρω τι ακριβώ εννοούσαν, αλλά πάντως σε κάθε περίπτωση ε, εκπροσωπούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό πολυλογιστέ οι οποίοι του κάνουν τη δουλειά αυτά ω προ του διεθνεί κανόνε που αναφέρουν ότι οι καλλιτέχνε εκεί που δραστηριοποιούνται πρέπει να φορολογούνται και θα πρέπει να ε, δηλώνουν το εισόδημά του εκεί. Αυτά ως προς την φοροαποφυγή και τη μη συμμόρφωση. Αυτά είναι τα βασικά προβλήματα που υπάρχουν. Ωστόσο, στην πράξη, το, το μέτρο αυτό αποσκοπούσε στο να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα ονόματα. Όπως ο Chris Froome, ο Ποδηλάτης, ο Μαξ Verstopper, ο πρώην οδηγός Φόρμουλας 1 που μετέφερε την έδρα του στο Μονακό και που δεν αυτοί που δεν θέλουν να πληρώσουν φόρους πουθενά δηλαδή. Δεν αφορούσε το 90-95% των απλών καλλιτεχνών και αθλητών. Παρ' όλα αυτά ε, υπάγονται και εκείνοι στον ίδιο κανόνα γιατί δεν υπάρχουν εξαιρέσει. Υπάρχουν λοιπόν κάποια προβλήματα. Πρώτον, κατά πόσο μπορεί κανείς να... να πώς, κατά πόσο είναι... Ε, πόσο εκπίπτουν οι δαπάνες σε αυτές τις, ε, σε αυτές τις ε, δραστηριότητες ε, ας ε, πάρουμε μια, ένα παράδειγμα. Βλέπετε εδώ την, ε, τη μαέστρο Αριάν Ματιάκ. Έχει για παράδειγμα 20 δουλειές το χρόνο, φυσικά έχει δαπάνες, ζει, μένει στις κάτω χώρες αλλά πηγαίνει και σε άλλες χώρες και είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν πηγαίνει σε μια ορχήστρα στην Γαλλία. Η ορχήστρα αυτή δυσκολεύεται πάρα πολύ για, αυτές, για αυτές τις ε, μία-δύο-τρεις μέρες να ε, δηλώσει ως δαπάνες αυτά που έχει πληρώσει για την έλευση της Αριάν και η Γαλλία ε, φορολογεί σε, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό για την ίδια την καλλιτεχνική δραστηριότητα, για την εκδήλωση δηλαδή και όχι, για, και όχι βάσει των εσόδων. Έτσι λοιπόν καταλήξαμε σε τρία είναι, είναι πρόβλημα αυτό. Το επόμενο πρόβλημα είναι όταν έχει παρακρατηθεί ο φόρος στο εξωτερικό, πώς μπορείς να τον ξαναπιστωθείς, πώς θα πάρει την επιστροφή του φόρου. Γιατί όπω και η Αριάν Ματιάκ, είπα ότι έκανε 20 ε, συναυλίες το χρόνο, άρα πρέπει να πάρει 20 φορολογικές βεβαιώσεις σε 20 διαφορετικές γλώσσες ενδεχομένως από άλλες χώρες και εδώ βλέπετε το επόμενο θέμα Φιλαρμονική Ορχήστρα του Air, Rotterdam με 18 ε, ε, ε, μουσικούς που είναι απίστευτο, είναι, είναι αδύνατον να, να, να ζητήσεις επιστροφή φόρου γιατί μπορεί να πας στη Γερμανία αυτή η ορχήστρα για να γίνει μια παρακράτηση φόρου αλλά η οποία είναι πάρα πολύ μικρή και μετά επιστρέφει επιστρέφει στο Ρότερνταμ. Είναι, είναι, είναι αδύνατον πρακτικά να, να, να πάρει πίσω όλο αυτό το φόρο που έχει παρακρατηθεί σε διάφορε χώρε τι οποίε μπορεί να έχει κάνει κάποια εκδήλωση, να έχει δώσει κάποια συναυλία. Ακόμη όμω και αν τα ξεπεράσει όλα αυτά τα προβλήματα, ε, χρειάζεσαι φοροτεχνικό. Στην ε, Ολλανδία, εγώ δεν λέω ότι είμαι ο πιο ακριβώς ε, της αλλά κάτι πρέπει να πάρω κι εγώ, κάπω πρέπει να αμυφθώ και ε, μετά η Αριάν πρέπει να πάρει ένα φοροτεχνικό και στη Γαλλία και στις όλες χώρες και φυσικά και οι γαλλικές και οι ε, ολλανδικές, ολλανδικές φορολογικές αρχές επιβαρύνονται με κάποιο κόστος γιατί πρέπει να παρακρατηθεί ο φόρος, να, να ανταλλαχθούν κάποια έγγραφα, όλα αυτά δεν γίνονται αυτόματα, άρα μιλάμε για υψηλό διοικητικό κόστος όλης αυτής της διαδικασίας. Ιδίως αν συγκρίνεις τα έσοδα, τα φορολογικά, ε, με αυτά που έχουν τελικά αποτελέσει ε, τα έσοδα της, ε, της εκάστοτε εκδήλωσης. Όταν λοιπόν πηγαίνει σε άλλη χώρα, υπάρχει άλλος φορολογικός συντελεστής, άλλο φορολογικό σύστημα, άλλοι κανόνες για την επιστροφή ή την έκπτωση φόρου, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθείς μέσα σε αυτήν την παγίδα, μέσα σε αυτόν τον κικαιώνα κανόνων ε, όταν κανείς ε, δραστηριοποιείται καλλιτεχνικά στο εξωτερικό ή διασυνοριακά εν γέννη. Εδώ βλέπω, βλέπετε κι άλλο ένα παράδειγμα, το Within Temptation, ένα rock gothic ε, συγκρότημα, φαντάζομαι τους ξέρετε, εκπληκτική μουσική κάνουν και πηγαίνουν με το λεωφορείο τους, με το δικό τους εξοπλισμό, το, το φωτισμό τους, τον ήχο τους και με 12 τεχνικούς ε, έχουν και μάνατζερ και πράκτορες μαζί τους, ε, κάνουν 80% των δαπανών τους λοιπόν ε, καθώς βρίσκονται σε περιοδία και στη Γαλλία πρέπει να, πληρώσεις, να προπληρώσεις το 80% άρα έχεις μόνο 5% που σου μένουν από τον προϋπολογισμό για, για, για να πας να δώσεις μια συνευλία. Είναι προβλήματα αυτά. Ταυτόχρονα βεβαίως υπάρχουν και κάποιες λύσεις ε, η Ιρλανδία και η Δανία δεν εισπράττουν αυτόν τον καλλιτεχνικό φόρο εδώ και χρόνια. Λένε, ε, έχουν πει ότι δεν τον θέλουμε, δεν θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να τον εισπράττουμε. Ε, το ίδιο έκανε και η, Ολλανδία από το 2007 και έπειτα, αλλά μόνο αν ο καλλιτέχνης προέρχεται από χώρα με την οποία οι κάτω χώρες έχουν διμερή φορολογική συμφωνία. Όχι από το Μονακό, για παράδειγμα. Για πολλές χώρες, λέει ε, ε, η, η, Ολλανδία, ότι δεν θέλω το φόρο, αλλά για πολλές τον εισπράττει. Επίσης, άλλο παράδειγμα υπάρχει ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το ελάχιστο κατόφλι για τον κάθε καλλιτέχνη είναι 11.500 στερλίνες για τους Βρετανούς αλλά και για τους ξένους καλλιτέχνες. Ε, αυτά είναι τα χρήματα δηλαδή που δεν φορολογούνται εφόσον έχουν κερδιθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτές είναι, αυτά είναι παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών, καλές πρακτικές δηλαδή. Ε, ο αθλητικός κόσμος έχει αποφασίσει ότι δεν, το θέλει πια, δεν τη θέλει πια αυτή τη διαδικασία. Μετά τη, τους Ολυμπιακούς του Σίδνη, το, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή είπε στον Καναδά θα πάρετε τους τους ε, χειμερινούς ε, Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά δεν θα χρεώσετε το 15% του φόρου. Και το ίδιο ισχύει πλέον ε, και στο ποδόσφαιρο, χώρες δηλαδή που πηγαίνουν σε άλλη, ομάδες μάλλον που πηγαίνουν σε άλλη χώρα για να παίξουν έναν αγώνα, δεν επιβαρύνονται με αυτόν τον φόρο, την παρακράτηση του φόρου. Έχουμε λοιπόν έρθει σε επαφή με τον, τον ΟΣΑ για να, για να διαγράψει το άρθρο 17. Ε, Ο ΣΑ αποφάσισε να μην το κάνει, για λόγους που κατά τη γνώμη μου είναι εσφαλμένοι, μπορείτε να διαβάσετε και στο άρθρο που έχω γράψει. Υπάρχουν όμως κάποιες εξαιρέσεις κάποιοι, από κάποιους περιορισμούς. Για παράδειγμα, εξαιρούνται οι υπάλληλοι ε, της φιλαρμονικής ε, ε, του Ρότερνταμ, υπάρχουν κάποιες ελάχιστες, ελάχιστα κατόφλια, ε, όπως κάνουν ε, το, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Υπάρχει κάποιο όριο για επιδοτούμενες καλλιτεχνικές δραστηριότητες που ε, περιλαμβάνονται και σε διάφορες διμερείς συμφωνίες. Ποιες λοιπόν είναι οι λύσεις που θα πρότεινα εγώ. Πρώτον, μπορεί να ακολουθήσει κανείς την ε, Ολλανδία, την Ιρλανδία και την Δανία, αλλά εκεί μόνο για τους ανθρώπους ε, ε, που προέρχονται από χώρες με τις οποίες έχει φορολογική συμφωνία. Διαγραφή απαλληφή του άρθρου 17 ή χρήση των περιορισμών του ΩΣΑ. Και επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει έναν κώδικα δεοντολογίας για την παρακράτηση φόρου ε, στα δικαιώματα από πολιτιστικό περιεχόμενο και νομίζω ότι αυτός ο, ε, ο κώδικας θα πρέπει να αφορά και τους ε, καλλιτέχνες και τους αθλητές. Ένας κώδικας δεοντολογίας δηλαδή για την παρακράτηση φόρου. Η Κομισιόν επίσης έχει συστήσει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων η οποία κατέληξε και σε έκθεση ε, το Δεκέμβριο του 2015 σχετικά με την επίλυση προβλημάτων ε, διασυνοριακών προβλημάτων φορολογικού χαρακτήρα και εκεί υπάρχει ένα ειδικό κεφάλαιο, κεφάλαιο και για καλλιτέχνες και αθλητές και εκεί περιλαμβάνονται μια σειρά απολύσεις που θα μπορούσαν να προκριθούν και να εφαρμοστούν. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε. Αγγίξαμε τομείς που συνήθως δεν απασχολούν την Επιτροπή Πολιτισμού, φορολογικά, έκπτωση φόρου, παρακράτηση, αλλά βεβαίως πρέπει να πω ότι εγώ δεν γνώριζα ότι ήταν τέτοιε δυσκολίε που αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνε. Και βλέπουμε πιο ξεκάθαρα νομίζω, το βλέπουμε σας πιο ξεκάθαρα στον χώρο του αθλητισμού, αλλά και για τους ε, μεγάλους ε, καλλιτέχνες διαπιστώνεται ότι υπάρχει δυνατότητα πάντα να χρησιμοποιήσουν, να αξιοποιήσουν κάποια μαύρη τρύπα φορολογική. Και μετά επιβάλλονται ρυθμίσεις, ε, νομοθεσία η οποία πλήττει αυτούς που δεν έπρεπε να πλήξει. Βεβαίως και κανείς μας δεν δέχεται να υπάρχουν και καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν ε, πάρει έδρα στο Μονακό και δεν πληρώνουν φόρο αλλά εξίσου απαράδεκτο μου φαίνεται και να ε, πιέζονται τόσο πολύ από διάφορες πλευρές ε, μικρότερου ελληνικούς καλλιτέχνες. Ο Στοιεύσκη έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ για την παρουσίαση, ήταν ε, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Και θα ήθελα, Πρόεδρε, να ζητήσω να δώσουμε την ευκαιρία για μια συζήτηση για τα φορολογικά σε μια από τις ακροάσεις, από τις ε, συνεδριάσεις μας, μια ιδιαίτερη ακρόαση, γιατί είναι τόσο πολλά τα θέματα που θα πρέπει νομίζω να ασχοληθούμε μόνο με τα φορολογικά συστήματα, τα σχετικά με την τέχνη. Ευχαριστώ τον κύριο Μόλεναρ. Είχαμε μια συζήτηση νομίζω, μια εισαγωγή νομίζω στη συζήτηση από τον καθηγητή Ζικ Θέμελς την καθηγήτρια που συνεργάζεται μαζί σας, είχε έρθει για μια διάλεξη, διατύπωσε και προκλητικά ερωτήματα βέβαια, τα οποία θα επανέλθω. Καταρχάς, εάν μία νοσοκόμα πληρώνει φόρους, γιατί δεν θα πρέπει και ο καλλιτέχνης ή ο αθλητής να πληρώνει φόρους. Πρόκειται για διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Προνομιούχες. Και άλλη μια ερώτηση που διατυπώθηκε σε, εκείνο το, σχέδιο εκείνη τη διάλεξη και την επαναλαμβάνω. Καλύτερα να δοθεί η φοροαπαλλαγή, η φοροελάφρυνση ή να υποστηριχθεί μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, να ενισχυθεί ένας καλλιτέχνης δηλαδή. Αυτό το αναφέρω διότι οι περισσότεροι καλλιτέχνε είναι αυτοαπασχολούμενοι. 60% των καλλιτεχνών δεν έχουν ε, άλλη οικονομική δραστηριότητα και άρα δεν τους ε, προσφέρουν τίποτα οι φοροαπαλλαγές, δεν κερδίζουν τίποτα. Και άρα περνάμε σε ένα συναφές ζήτημα και σημαντικό. Είχα μία ορχήστρα σχηματίσει για δύο μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο με Τσέχους, Πολωνούς, Λευκορώσους και άλλους μουσικούς. Λόγω της διαφοράς στα φορολογικά καθεστώτα και του κόστους, άλλοι ε, κατέγραψαν υψηλά έσοδα, ενώ άλλοι χρειάστηκε να πληρώσουν και από την τσέπη τους για να παίξουν στην ορχήστρα αυτή. Ήταν τέτοιες οι διαφορές φορολογικές στην Ευρώπη. Για μένα κρίσιμη σημασία είναι όχι μόνο το τι κάνουν οι καλλιτέχνες, αλλά ταυτόχρονα και πάνω απ' όλα η υποστήριξη της ε, πολιτιστικής πληρονομιάς. Αλλού βλέπουμε ΦΠΑ 23% και αλλού ε, ευνοϊκότερη φορολογική μεταρρύθμιση ως κίνητρο, ε, μεταχείριση ως κίνητρο. Γι' αυτό λοιπόν, Πρόεδρε, προτείνω και επιμένω μια προσεχή μα συνεδρία να αφιερωθεί ειδικά στα θέματα τα φορολογικά στον πολιτισμό. Σα ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρο. Κυρία Σόιντρουβα. Αχ, με συγχωρείτε. Όχι, όχι. Είχα ξεχάσει ότι κάνουμε το σύστημα ping-pong τώρα. Για να ακούσουμε την απάντηση, κύριε Μόλεναρ. Ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Νομίζω ότι είναι καλή ιδέα να ε, συνεδριάσει η Επιτροπή για θέματα φορολογικά. Εγώ ασχολήθηκα με αυτό το ζήτημα μόνο σήμερα, αλλά κάποιες από τις παρατηρήσεις σας σχετίζονται με αυτό. Γνωρίζω την καθηγήτρια. Συνεργαζόμαστε στο Πανεπιστήμιο Εράσμους και πρόθεση της παρέμβασής μου σήμερα ήταν ακριβώς να μεταφέρω αυτό το μήνυμα. Θέλουμε μια δίκαιη φορολογία έτσι ώστε οι καλλιτέχνες να μην φορολογούνται χειρότερα και περισσότερο από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Στο παράδειγμα σας με την νοσηλεύτρια και τον καλλιτέχνη, στο θέμα που με απασχολεί, το performing arts που ο καλλιτέχνης που κάνει performing art και ε, δείχνει τη δουλειά του από τη μία χώρα στην άλλη φορολογείται χειρότερα από την νοσηλεύτρια. Υπάρχει ε, διπλή φορολογία ή υπερβολική φορολογία και πρέπει να αρθεί αυτό το εμπόδιο και το πρόβλημα να λυθεί. Ένα δεύτερο παράδειγμα με πολύ μικρό εισόδιο, με περίπτωση ατόμων με πολύ χαμηλά εισοδήματα που δεν ε, χρειάζονται ε, να πληρώσουν φόρο γιατί βρίσκονται εντός του αφορολόγητου ορίου, όμως αν πάνε στο εξωτερικό πρέπει το 50% των εσόδων να το πληρώσουν σαν φόρο στη Γαλλία ή το 20% τόσο στην Αυστρία. Αυτό είναι προβληματικό για αυτά τα άτομα, ότι δεν έχουν επιστροφή φόρου στο σπίτι τους, γιατί είναι στο φορολόγητο. Και είναι πολύ δύσκολο να υποβάλουν δηλώσεις ε, στη Γαλλία ή στην εκάστοτε χώρα για να απαλλαχθούν. Ε, ήδη δηλαδή πληρώνουν παρόλο που τα αιτήσια συνολικά εισοδήματά τους είναι πολύ χαμηλά. Και ε, αυτό συμβαίνει στα μέλη σε κάθε ορχήστρα και πολύ συχνά είναι και ο λόγος που δεν δέχονται να συμμετάσχουν. Ευχαριστούμε. Κυρία Σόιντροβα, προσπαθήστε σας παρακαλώ σε ένα λεπτό αν μπορείτε. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε να σας ε, ακούσουμε. Δεν έχω θέσει ερωτήματα, αλλά εδώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Είναι άλλο πράγμα η φορολογία και άλλο πράγμα το εισόδημα. Εμάς φυσικά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι καλλιτέχνες να έχουν εξασφαλισμένο εισόδημα. Βεβαίως η φορολογία θα συνεχίσει να αποτελεί εθνική αρμοδιότητα. Άρα δεν έχουμε εμείς αρμοδιότητα ευρωπαϊκή να ε, καταλήξουμε σε κάποια συγκεκριμένη σύσταση. Καλό είναι βεβαίως να ακολουθούνται τα καλά παραδείγματα που υπάρχουν. Όμως, ως προς τις φορολογικές ελαφρύνσεις, αναρωτιέμαι κατά πόσο είναι ηθικά σωστό όταν οι καλλιτέχνες χρησιμοποιούν δημόσιες υπηρεσίες που πληρώνονται, ε, χρηματοδοτούνται από τα χρήματα των ε, φορολογουμένων. Κάποιος πρέπει ε, για, όλους, για όλες αυτές τις υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης, υγειονομικές υπηρεσίες να καταβάλει το, το τίμημα. Φυσικά και θέλω οι δημιουργοί να έχουν τους θεατές τους, τους ακροατές κτλ. αλλά θα πρέπει και να φορολογούνται. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε, κύριε Μολινάρ. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Πρέπει όλες οι χώρες να έχουν φορολογικά έσοδα βεβαίως. Δεν το αφισβητώ αυτό ούτε υπερασπίζομαι τη θέση ότι θα πρέπει να έχουν ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς οι καλλιτέχνε. Όχι, να μην έχουν ευνοϊκό, να έχουν ίσο με τους υπόλοιπους πολίτες και όχι βαρύτερο και επαχθέστερο φορολογικό καθεστώς. Και να πω ξανά κάτι που έχω ήδη πει. Όταν οι χώρες μπουν σε συνθήκες μεταξύ τους και συνομολογήσουν ότι θα καταργήσουν αυτή την παρακράτηση φόρου, όταν πράγματι θα καταργήσουν το άρθρο 70, όντως θα απολέσουν τα εισοδήματα από τους ξένους καλλιτέχνες που έρχονται ε, στη χώρα τους, αλλά δεν θα χρειαστεί να δώσουν και φορολογική επιστροφή στους δικούς τους εγχώριους καλλιτέχνες που ε, κάνουν παραστάσεις στο εξωτερικό. Χάνει μια χώρα δηλαδή το έσοδο από αυτούς που την επισκέπτονται, αλλά δεν χρειάζεται να επιστρέψει ε, φόρο σε αυτούς που εργάζονται στο εξωτερικό. Και έτσι εξισώνεται η φορολογία. Είναι ίση, ισότιμη φορολογία με τους υπολείπους πολίτες. Ευχαριστώ. Η κυρία Ροντρίκες, για ένα λεπτό παρακαλώ. Δεν μπορώ να μιλήσω πορτογαλικά, μπορώ. Α, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τις ε, παρουσιάσεις σας. Δεν είμαι καθόλου βέβαιη ότι θα πρέπει ότι οι καλλιτέχνες με γίνονται αντικείμενο διαφορετικής μεταχείρισης. Ξέρετε, είμαι από μια χώρα που έχει υποφέρει από τη λιτότητα και η Ελλάδα το ίδιο στην Ευρώπη υπάρχουν εξόχως απόκεντρες περιοχές. Εγώ είμαι από τη Μαδέιρα και έχω, υπάρξει, έχω δουλέψει ως καθηγήτρια στη Βραζιλία. Για να πάει κανείς από τη Μαδέιρα στη Βραζιλία να δουλέψει, αυτό μου στήχει σε χι ευρώ για παράδειγμα. Χρειάστηκε να αξιοποιήσω το προσωπικό, να έχω εργαλεία. Ένα ταξίδι από τη Μαδέιρα στη Λισαβόνα στοιχίζει περίπου 500 ευρώ. Είναι πολύ πιο ακριβό από ότι να πάει κανείς από τη Λισαβόνα στις Βρυξέλλες. Και Μιλούμε για 8 εκατομμύρια άτομα, Ευρωπαίοι πολίτες, που ζουν στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες. Υπάρχει και το νησί της Ρενιού που είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν μέρη πολύ πιο απομακρυσμένα. Τονίζω λοιπόν το θέμα της κινητικότητας. Δεν λέω λοιπόν η φορολογία να είναι ανώτερη, αλλά έχουμε τρεις τρόπους φορολόγησης των καλλιτεχνών στην Πορτογαλία, όχι μόνο τους καλλιτέχνες, αλλά και όλων των υπολείπων. Στη Βραζιλία ήμουν καθηγήτρια Πορτογαλικών, αποσπασμένη και διορισμένη στη Βραζιλία. Και με φορολογούσαν και στη Βραζιλία και στην Πορτογαλία. Το ίδιο συμβαίνει και με τους καλλιτέχνες. Οι άνθρωποι που ζουν στις εξωγως απόκεντρες περιοχές έχουν κόστος πολύ ανώτερο ε, σε σχέση με τους άλλους και γι' αυτό αυτό το ίση φορολόγηση για όλους μου φαίνεται τελικά κάπως άδικο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μόλιναρ. Η ίση φορολόγηση επί των κερδών μετά τη της σύμφωνα με την οποία θα εκπέσουν οι δαπάνες. Δηλαδή πάει κανείς από τη Μαδέιρα στη Βραζιλία και έχει έξοδα, πρέπει να πάρει προσωπικό μαζί του, ε, την ομάδα του. Αυτό ήταν το πρώτο πρόβλημα που εξήγησα. Το να μπορούν να εκπέσουν οι δαπάνες είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ε, ο φορολογικός συντελεστής είναι δυσθεώρητος. Επομένως η φορολογία ή η φορολογία μετά την έκπτωση των δαπανών. Βεβαίως. Δώσατε και το παράδειγμα του ότι ήσασταν καθηγήτρια από την Πορτογαλία και διδάσκατε στην Βραζιλία. Αν πάτε από την Πορτογαλία στη Βραζιλία ως καθηγήτρια δασκάλα, θα πάτε για χι χρόνο, τρεις μήνες, έξι μήνες, ένα χρόνο. Στο άρθρο 15 λέει ότι η Βραζιλία έχει το δικαίωμα να φορολογήσει το εισόδημα και εσείς θα έχετε φοροαπαλλαγή ε, από την Πορτογαλία αντίστοιχη και άρα ε, είναι πολύ σαφές τι έχετε κερδίσει και τι έχετε βγάλει σε κάθε χώρα. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, αλλά είναι πιο εύκολο από ότι όταν μια πορτογαλική μπάντα, ας πούμε, πάει στη Βραζιλία να παίξει μουσική, πρέπει να εκπέσει τις δαπάνες, ε, κάνει δύο-τρεις συναυλίες και μετά πρέπει να τις επιστραφούν αυτά στην Πορτογαλία. Γιατί στη Τουρνέ έχει πάει και στη Μοζαβίκη, στην Αγκόλα, στις διάφορες χώρες της Ευρώπης και έχει πληρώσει φόρους όλες αυτές τις χώρες, ακόμα και στις χώρες που εμφανίστηκε για ένα μόνο βράδυ, σε μία μόνο αυλία. Έχει πληρώσει ένα σωρό φόρους σε ένα σωρό χώρες και είναι τεράστια διοικητικά έξοδα. Πολύ περισσότερα διοικητικά έξοδα από τη μία μετάβαση ενός πολίτη που είναι καθηγητής και πάει μόνο σε μία άλλη χώρα, στη Βραζιλία στην περίπτωσή σας. Εγώ νομίζω ότι αυτό απασχολούμενοι θα πρέπει να αφορολογούνται μόνο στη χώρα της απασχόλησής τους, όπου έχουν σταθερή απασχόληση, ε, γιατί και οι δικηγόροι και οι αρχιτέκτονες και όλοι όσοι είναι αυτά απασχολούμενοι πληρώνουν φόρο μόνο στη χώρα τους. Τρεις παρεμβάσεις ακόμη και κατά παρέκκληση από το συστήματος ε, ping-pong θα τις πάρουμε και τις τρεις μαζί. Πόκταν Βέτα. Ευχαριστώ. Το ερώτημά μου αφορά τον αθλητισμό. Γιατί ήμουνα... Και ο αθλητισμός είναι τμήμα του πολιτισμού. Γιατί ήμουνα στην μεταβατική φάση στη, στη χώρα μου αθλητής από το ερασιτεχνικό στο επαγγελματικό. Εγώ ε, ήμουν ε, μέλος ενός συλλόγου που είναι κάτι σαν εταιρεία. Στα, στη δεκαετία του 90 ε, η φορολογική μου δήλωση αποτελούσε δικαιολογητικό έγγραφο για να πάρω την, την άδεια σκήσεω επαγγέλματο. Δηλαδή όπου και αν ζούσα, Γερμανία, Ισπανία, έπρεπε να υποβάλω πάντοτε τα, τα χαρτιά μου, τι φορολογικέ μου δηλώσει προκειμένου να μπορώ να συνεχίσω να, ε, συνεχίσω να δουλεύω. Υπάρχουν πάντοτε αυτά τα, τα δικαιώματα εργοδοτών και εργαζομένων. Κάποιες, ε, κάποια αθλήματα δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμα ως επαγγελματικά στην Ευρώπη. Ε, ακούμε άλλες φορές ότι σε κάποια αθλήματα μπορεί να, να πάρεις και 200 εκατομμύρια ευρώ. Ε, και μετά η κοινωνία ε, θεωρεί δικαίως ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να, να, φορολογούνται, γιατί αλλιώς δημιουργείται μια, μια κοινωνική δυσαρέσκεια. Είπατε και για τη Δανία. Εγώ άκουσα ότι ε, ε οι συνάδελφοί μου Δανείοι που, που έπαιζαν στη Γερμανία, ε, όταν επέστρεφαν στη Δανία, στη Δανία ε, τα πρώτα χρόνια δεν δούλευαν, δεν πλήρωναν πάρα πολλά χρήματα. Έως ότου ε, άρχισε να εφαρμόζεται αυτό το σύστημα της Δανίας που περιγράψατε. Γιατί αυτό, και αυτό είναι σημαντικό, γιατί η συλλογή πραγματικά ενεργούν σε πολλές περιπτώσεις ως εργοδότες. Από αυτή την άποψη φυσικά θα πρέπει να φορολογούνται όλοι όσοι έχουν έσοδα. Σίλβια Κώστα, ένα λεπτό. Ξέρω ότι θα δυσκολευτείς πολύ, αλλά ελπίζω σε σένα. Ε, Μια διευκρίνηση μόνο. Υπάρχουν κάποια προβλήματα. Το ένα είναι η αναγνώριση του καθεστώτος του καλλιτέχνη που έχει ζητήσει κάποτε το κοινοβούλιο. Δηλαδή, το ιδιάζον χαρακτήρας του καλλιτέχνη που κυρίως για τους καλλιτέχνες του θεάματος έχει συντομότερη σταδιοδρομία αναγκαστικά, όχι βέβαια οι συγγραφής για την άλλη ιστορία. Όλο αυτό λοιπόν ε, μας οδηγεί στις εξής ε, υποθέσεις ή προσδοκίες να υπάρχει μια διευκόλυνση φορολογική σε εθνικό επίπεδο αν και εγώ πιστεύω ότι κάποιος κοινό παρονομαστής θα πρέπει να υπάρχει και το άλλο είναι αν κατάλαβα καλά ότι προτιμάτε αυτό με βέστο είπατε στο τέλος παρέμβασή σας πώς μπορούμε να ευνοήσουμε αυτό που θεωρούμε ότι το προτιμούμε και θεωρούμε ότι είναι προς το συμφέρον μας δηλαδή κινητικότητα των ε, καλλιτεχνών και ανάπτυξη μεταξύ τους συνεργασιών, χωρίς αυτό σημαίνει ότι επαλλάσσονται από το φόρο, χωρίς όμως ούτε να τους επιβάλλεται διπλή φορολογία, ούτε και να είναι στο απερόβλητο, γιατί κανείς δεν το θέλει αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ward. Μία ερώτηση θα ήθελα να θέσω. Με το Brexit υπάρχουν κίνδυνοι. Πρόσφατα μίλησα στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Βρετανικών Ορχιστρών έχουν κάνει μια πολύ περιστατωμένη μελέτη για το Brexit και ανέφεραν κάποια ζητήματα φορολογίας. Ποια είναι τα σχόλιά σας, θα υπάρχουν επιπτώσεις στις ορχήστρες, θα υπάρχουν επιπτώσεις και από εκεί και πέρα. Γιατί και το θέμα τι αξιοποιούμε και τι αξιολογούμε στις κοινωνίες μας. Σε καιρούς λιτότητας πρέπει να αλλάξουμε τις πολιτικές Κάποιοι ξέρουν για το New Deal. Στη δεκαετία του 30 η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφάσισε ότι θα ήταν καλή ιδέα να χρηματοδοτήσει οι καλλιτέχνες να κάνουν καλή δουλειά. Και γι' αυτό είχαμε τις υπέροχες τοιχογραφίες του Diego Rivera, ε, που τώρα είναι τουριστική ατραξιόν, αλλά και στο Κογκρέσο στην Ουάσιγκτον έχουμε αρχείο με μαρτυρίες από ανθρώπους που είχαν υπάρξει δούλοι και δεν θα είχαν ποτέ συλλεγεί αυτές οι μαρτυρίες και δεν θα υπήρχε αυτό το πολύ πλούσιο αρχείο αν οι πολιτικοί άνδρες και γυναίκες δεν είχαν πει ότι πράγματι χρειαζόμαστε αυτό στην κοινωνία μας. Ωραία λοιπόν, ο κύριος Μόλενας, για μέσα δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καταρχάς για τα αθλήματα να σας πω το εξής. Μία από τις παρατηρήσεις που κάνατε ε, ήταν ότι πολλοί ε, αθλητές δεν είναι επαγγελματίες, με την έννοια ότι δεν κερδίζουν πάρα πολλά χρήματα και ένα παράδειγμα έχουμε είναι ε, ένας καλλιτέχνης ο οποίος είναι στο αφορολόγητο και δεν πληρώνει φορό στη χώρα του γιατί δεν κάνει τόσο πολλές συμβολίες συναυλίες. Το ίδιο συμβαίνει και με ε, τους αθλητές. Έχω πελάτες που είναι παίκτες γκολφ που θέλουν να φτάσουν στην κορυφή αλλά είναι στην τρίτη κατηγορία. Δηλαδή ε, ε, ό,τι κερδίζουν σε ένα χρόνο είναι εντό του αλλά ουσιαστικά έχουν αφήσει μέρη χρήματα φορολογημένα στην Ιταλία και αλλού όπου έχουν πάει να παίξουν κόλφ. Απ' την άλλη υπάρχουν αθλητές που κερδίζουν εκατομμύρια, ελάχιστοι, λίγοι οι χώρες μπορεί να θέλουν να συνεχίσουν να, τις τους φορολογούν και αυτό είναι απολύτως κατανοητό. Δεν είναι όμως αυτή η επίσημη πολιτική. Η επίσημη πολιτική είναι ότι θέλουμε να επιτεθούμε ε, σε αυτούς που προσπαθούν να αποφύγουν τη φορολογία. Δεν ε, μιλούμε ξεκάθαρα για το θέμα του προϋπολογισμού. Στο Ενωμένο Βασίλειο το φορολόγητο είναι 11.500 στερλίνες το χρόνο. της. είπα ε, το φορολόγητο είναι 30.000 δολάρια ετησίως. Το μοντέλο του ΟΣΑ περιλαμβάνει αφορολόγητο. Άρα οι χώρες μπορεί να πούνε μία στην άλλη ότι θέλουμε να φορολογήσουμε τους μεγάλους, δεν θέλουμε να τους αφήσουμε να φύγουν. Μπορούν να βάλουν ένα τέτοιο ελάχιστο κατόφλι αφορολόγητο στη σύμβαση με τη διεθνή που θα υπογράψουν. Όχι 400 ευρώ το χρόνο, 20-30 χιλιάδες το χρόνο, γιατί έτσι απαλλάσσονται οι μικροί. Δηλαδή το 90% που αυτή τη στιγμή υφίσταται αυτή την τεράστια διάκριση και θα απελευθερωθεί έτσι το 90% των ενδιαφερομένων. Συμφωνώ με την κυρία Κώστα, η επαγγελματική ζωή είναι πολύ βία και ο κίνδυνος διπλής φορολόγησης ε, υλοποιείται υπερβολικά συχνά. Ως προς το Brexit και την έκθεση του Συλλόγου Βρετανικών Ορχιστρών μπορώ να σας πω ότι πράγματι υπάρχουν κίνδυνοι με θέματα ΦΠΑ που δεν ήταν το αντικείμενο μου σήμερα, αλλά και με τη φορολόγηση για τις παραστατικές ε, τέχνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκπίπτουν οι δαπάνες και το δικαίωμα υποβολής δηλώσεων είναι θέμα ευρωπαϊκό. Και όταν ε, φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί να γίνει καμία έκπτωση και απαλλαγή. Δεν υπάρχουν φορολογικές συνθήκες με τις άλλες χώρες ε, δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο με το Brexit θα είναι σε χειρότερη θέση από ό,τι είναι η ΕΠΑ ΕΕ σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες, γιατί υπάρχουν φορολογικές συνθήκες σε ε, σχέση με τις ε, χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΕΠΑ. ΕΕ. Μιλήσατε για την αξία των τεχνών και συμφωνώ, είναι το τελευταίο μου σχόλιο όταν μονομερώς αποφασίσουν οι χώρες να παραιτηθούν από αυτή την παρακράτηση φόρου όπως έκαναν οι το χώρο το 2007 και η Ιρλανδία στη συνέχεια, το 2006 η Ολλανδία παραιτήθηκε από 6 εκατομμύρια ευρώ φορολογικών εισοδημάτων, φορολογικών εσόδων. Και πέρσι ε, υπολογίσαμε με κάποιους Βρετανούς συναδέλφους ότι αν το κάνει μονομερός η Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, όχι στη Διεθνή Σύμβαση, θα παραιτηθεί από φορολογικά έσοδα ύψου 40 εκατομμυρίων ε, στερλινών, 40 εκατομμύρια στερλίνες, ε, λιγότερες θα εισπράξει. Όταν το κάνει κανείς μονομερός, δηλαδή δεν είναι και ένα τεράστιο ποσό, αλλά είναι καλύτερο να συμβεί διμερός γιατί μπορεί να χάνει έσοδα, αλλά δεν χρειάζεται να κάνει και επιστροφές φόρους κράτος και δεν χρειάζεται να τις δώσει αυτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Μιλούμε πάντοτε για την ενιαία αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λίγο παράδοξο το ότι συνεχίζουμε να μιλούμε για διμερείς φορολογικές ε, συμφωνίες. Παρ' όλα αυτά, ε, είναι και αυτό στοιχείο που δείχνει πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει ενοποίηση και στον τομέα της φορολογίας στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ε, εμπειρογνώμονες, τους προσκεκλημένους μας. Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσες ε, και οι συμβουλές σας και οι πληροφορίες σας και περνάμε... Καταρχάς να σας ευχαριστήσω λοιπόν για την παρουσία σας, για την, ε, για την συμβολή σας στη συζήτηση. Να σας χειροκροτήσουμε κιόλας γιατί το αξίζετε πραγματικά. Και περνάμε κατευθείαν στο σχέδιο έκθεσης διορθωτική φραγμή για την πρόσβαση στα πολιτιστικά αγαθά. Μπορείτε να καθίσετε βεβαίω να παρακολουθήσετε τη συζήτησή μας, Αν έχετε όμως ανηλυμένε υποχρεώσεις σας κατανοούμε πλήρως. Σας ευχαριστώ άλλη μια φορά για την παρουσία σας εδώ. Και δίνω κατευθείαν το λόγο στον κύριο Στογεύσκη για πέντε λεπτά, προκειμένου να μας παρουσιάσει την έκθεσή του, να μας πει τι ε, σκοπεύει να συμπεριλάβει σε, αυτή την έκθεση πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσω ε, αναφέροντας κάτι πολύ σημαντικό αρχικά. Όσον αφορά τους φραγμούς στην πρόσβαση στον πολιτισμό. Είναι πρώτη φορά που συζητούμε αυτό το θέμα από μια ολοκληρωμένη ε, σκοπιά και όχι ε, με κατακαιρματισμένο τρόπο. Δύο, δύο είναι τα βασικά και σημαντικότερα στοιχεία. Πρώτον, κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δικαίωμα να συμμετέχει στον πολιτισμό. Αυτό είναι ε, δικαίωμα που κατοχυρώνεται στις συνδίκες και Δεύτερον, ο βαθμός συμμετοχής στον πολιτισμό στον πολιτισμό αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη της Ευρώπης. Επίσης, η πολιτιστική πυκλομορφία της Ευρώπης πρέπει να προστατεύεται από το νόμο. Τέταρτον, πρόσβαση στον πολιτισμό πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Κάθε δημόσια διοίκηση έχει τρεις βασικούς στόχους που πρέπει να επιτύχει. Πρώτον, να εκπαιδεύει καλλιτέχνες. Δεύτερον, να εκπαιδεύει το κοινό. Και τρίτον, να δημιουργεί τις απαραίτητες υποδομές μέσα στις οποίες μπορεί το κοινό να συναντά τους καλλιτέχνες και το αντίστροφο. Η διαμόρφωση λοιπόν των πολιτιστικών αναγκών αποτελεί καθήκον των δημόσιων αρχών αλλά και συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης θέλω να τονίσω ότι χρειάζεται να έχουμε μια ευρύτατη αντίληψη ε, του πολιτισμού. Μιλώ για καλλιτέχνες και το καλλιτεχνικό τους έργο αλλά και τις δραστηριότητες των πολιτών. Και βεβαίως σε αυτό περιλαμβάνεται και η πολιτιστική κληρονομιά. Τώρα, έχουμε το εξή πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα ζήτησης πολιτιστικών αγαθών, όχι προσφοράς. Και οι προφορίες που ακούσαμε το απέδειξαν αυτό. Φαίνεται ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες που δεν έχουν, καμία ανάγκη να συμμετέχουν στον πολιτισμό καθόλου. Η απάντησή τους είναι δεν μας ενδιαφέρει, δεν συμμετέχουμε γιατί δεν νιώθουμε καμία ανάγκη. Φυσικά δεν υπάρχουν πολίτες που δεν συμμετέχουν καθόλου στον πολιτισμό. Με στενούς όρου κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο. Αλλά η ποιότητα και το βάθος της συμμετοχής ε, παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλη ποικιλομορφία σε όλη την Ευρώπη. Και επιπλέον στοιχείο. Η γνώση του πολιτισμού αποτελεί προϋπόθεση και βασικό δείκτη της ικανοποίησης από τη συμμετοχή στον πολιτισμό. Όσον αφορά τους φραγμούς, θέλω να τονίσω ότι η βασική φραγμή είναι οικονομική, ένα, δύο, εκπαιδευτική, δηλαδή έλλειψη γνώσεων και τρίτον, δομικά εμπόδια. Αυτά είναι τα βασικά ε, εμπόδια. Υπάρχει όμως και ένα τέταρτο εμπόδιο που είναι το τα τεχνολογικά εμπόδια. Μια τέταρτη κατηγορία εμποδίων δηλαδή. Πρώτον, λεφτά. Νομίζω ότι ήταν σαφές και από τις παρουσιάσεις που παρακολουθήσαμε ε, πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ένα σαφές φορολογικό σύστημα και πόσο μπορεί να βλάψει την καλλιτεχνική δημιουργία, η δημιουργία, ε, η ασάφεια ε, ως προς τα βρολογικά καθεστώτα. Δεύτερο, η, η εκπαίδευση στον πολιτισμό μπορεί να αποτελέσει μεγάλο εμπόδιο. Η έλλειψη εκπαίδευση, παιδείας δηλαδή στον πολιτισμό. Γι' αυτό και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και μέρημνα για την εκπαίδευση των νέων ανθρώπων προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν ε, στην πολιτιστική δημιουργία. Και παρεμπιπτόντως να αναφερθώ και σε μια ψυχολογική πτυχή του θέματος. Στην Ευρώπη υπάρχει ευρύτατη αποδοχή, είναι ευρύτατα αποδεκτό κανείς να έχει χαμηλό επίπεδο γνώσεων στον πολιτισμό. Αυτό είναι πάρα πολύ ενισχυτικό. Τρίτη κατηγορία εμποδίων, τα διαρθρωτικά, τα, τα δομικά εμπόδια. πόσο κοντά δηλαδή στο σπίτι σου ε, βρίσκεται μια βιβλιοθήκη ή ένα θέατρο. Γιατί όσο πιο κοντά είναι, τόσο πιο πιθανό είναι να συμμετέχει στην πολιτιστική ζωή. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να, αρθούν τα δομικά εμπόδια. Και τελευταία κατηγορία εμποδίων, η τεχνολογία. Γνωρίζουμε πολύ καλά τις παραδοσιακές μορφές συμμετοχής. Να πηγαίνει κανείς στο θέατρο, για παράδειγμα, ή να διαβάζει ένα βιβλίο κτλ. κτλ. Λίγα όμως στοιχεία γνωρίζουμε όσον αφορά τη συμμετοχή μέσω, στον πολιτισμό μέσω του ίντερνετ. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την ευρύτατη επισκόπηση. Και ξεκινούμε με τους σκιώδες ηγητές. Κυρία Ροντρίγκους. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Το έγγραφο αυτό μας επιτρέπει να καταλάβουμε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα θέματα. Άπτονται οριζοντίως και καθέκτος όλων των στοιχείων που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό. να ενισχυθεί το κεφάλαιο που έχει να κάνει με τα εμπόδια προς την εκπαίδευση, γιατί η εκπαίδευση είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει να υπερπηδηθούν τα εμπόδια προς τον πολιτισμό. Για να δημιουργηθούν εταιρικέ και στρατηγικές σχέσεις θα πρέπει να έχουμε πολιτιστικά προγράμματα. Εταιρικέ σχέσεις μεταξύ σχολικών ιδρυμάτων και πολιτιστικών ιδρυμάτων, γιατί όχι και διασυνοριακή συνεργασία. Για να μετριάσουμε τα εμπόδια αυτά. Και ό,τι έχει να κάνει με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Τα κράτη-μέλη να μειώσουν το κόστος για τους νέους, για τους ηλικιωμένους, για τα μέλη πολυάριθμων οικογενειών. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια και κυρίως για τις χώρες που υποφέρουν απολυτότητα να αναθεωρηθούν οι πολιτικές που έχουν να κάνουν με την επιχορήγηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων για να μην υπάρχουν πληθυσμιακές ομάδες που είναι αποκλεισμένες. Η έκθεση αναφέρει μία από τις αρνητικές παρα απαραμέτρους. Μιλούμε για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πρέπει να υπάρχουν εταιρικέ σχέσεις με τους τοπικούς πολιτιστικούς θεσμούς και τους περιφερειακούς θεσμούς. Και έτσι μπορούν να συμμετέχουν όλοι στη διαμόρφωση του αυριανού ακροατηρίου, του αυριανού κοινού να έχουμε μια ενοποιημένη στρατηγική για να υπερπηδήσουμε τα εμπόδια στα οποία, ε, τα οποία αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των εξόχως απόκεντρων περιφερειών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι πιο δραστήρια, να ενισχύσει ε, τα κίνητρα για την κινητικότητα των επαγγελματιών στον τομέα του πολιτισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μίχελς. Ευχαριστώ. Ήταν εκτεταμένη η επισκόπωση. Στατιστικές πολιτισμού, προαγωγή του πολιτισμού με δημόσια μέσα. Εγώ θέλω να ρωτήσω τι ακριβώς σκοπεύουμε να υποστηρίξουμε. Θα έχουμε να κάνουμε μια πολύ μορφή υποδομή πολιτισμού, θέατρο, σχολές τέχνης, αρχεία, βιβλιοθήκες, γκαλερί πινακοθήκες, ε, σύγχρονο έργο, πολιτιστική μνήμη. Δεύτερον, προσανατολισμοί προς, με, προς ένα είδος πολιτιστικού mainstreaming όπως αναφέρεται στις παράγραφους 4 και 5 ή αντίστοιχα ε, καινοτομία στην τέχνη. Τρίτον, δεν βλέπω ακριβώς τις προτάσεις το 9 σημείο 9 για τις επενδύσεις για το πολιτισμό και την οικονομία της δημιουργίας. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, εδώ έχουμε να κάνουμε την παραγωγή των μεγαλύτερων πολιτιστικών έργων του κόσμου. Βιβλία είναι αυτά, μουσική είναι αυτά, ε, άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Πρέπει να μιλήσουμε, πιστεύω, για τις ε, κακοπληρωμένες θέσεις εργασίας στον χώρο της τέχνης για να μπορέσει να αναπτυχθεί ένας υγιής διάλογος για τον πολιτισμό. Και, τελευταίο, στα ζητήματα της ε, εκμετάλλευσης δικαιωμάτων πνευματικών δημιουργών είναι νομίζω ανεπαρκής η έκθεση επιχειρημάτων σε σχέση με, τις, ε, με τους φορείς που συνιστούν ε, θεματοφύλακες, βιβλιοθήκες, αρχεία και ούτω καθεξής. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να βρεθεί μια διαφορετική λύση. Προσβλέπω βέβαια στην ε, συνεργασία και τις παρατηρήσεις μου τις ε, περιορίζω αυτές τις δύο, σε αυτούς τους δύο τομείς που εξέφρασε επιφυλάξη. Ευχαριστώ κυρία Μπίλτ. Ναι, ευχαριστώ. Μας προτείνεται ως εξήγηση την ε, έλλειψη μόρφωσης για τα λαϊκά στρώματα, ότι δηλαδή δεν μπορούν να καταλάβουν τι είναι τέχνη. Διαρωτώμεθα όμως και ποια είναι η προσφορά πολιτιστικού υλικού που πολλές φορές γενναιόδορες πολιτικές, δημόσιες πολιτικές υποστηρίξουν χωρίς όμως να προ... προτείνουν αυτό που θέλει ο κόσμος. Ο Ζων Βιλάρ, ο οποίος είναι ο διευθυντής του Φεστιβάλ της Αθηνιών, λέει ότι δεν παίρνει αρκετό χώρο η τέχνη, είτε η νέα, είτε η παλαιότερη, η πιο απαιτητική, τώρα ζητά, αναζητά νέα ερμηνεία. Ο ίδιος όμως φαντάζομαι ότι του ιδίου όμως φαντάζομαι ότι θα τρίζουν τα κοκαλά του διότι βλέπει ότι, βλέπουμε ότι σε ορισμένα φεστιβάλ και από τα πιο γνωστά στην Ευρώπη και τη Γαλλία είναι ανεπαρκέστατες ε, και πολύ ανεπαρκέστατες ε, οι προβολές ε, αποκλεισμένοι σε έναν elephantino πύργο ή ε, δημιουργεί και δεν έχουν καμία σχέση με τη λαϊκή τέχνη, με την τέχνη που απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Ιδιαίτερα για τη Γαλλία λοιπόν πολλά πράγματα ακόμα μένουν να γίνουν και ευχαριστώ τελεία. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Κύριε Κώστα, ένα λεπτό. Είναι πολύ ενδιαφέρον πιστεύω και ευχαριστώ τον εισηγητή. Είναι ενδιαφέρον το κείμενο της έκθεσης και μπορεί να αποτελέσει μια χρήσιμη συνεισφορά και μετά βέβαια την ακρόαση που είχαμε. Ε, τη δομή της ε, την ε, θεωρώ πολύ καλή. Ε, ωστόσο θέλω να επισημάνω τα εξής. Έχουμε κάποια στοιχεία ανεπαρκή όμως του ευρωβαριού μέτρου, έστω και να έχουμε κάποια εμβάθυνση σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Χρονιά για την Πολιτική Κληρονομιά. Άρα πρέπει να δούμε τι είδου ζήτηση υπάρχει σε παιδοπολίτη, όχι μόνο την προσφορά σε καλλιτεχνικό προϊόν και βέβαια και τα όρια, ή φραγμοί που μας απασχολούν. Πρέπει να αναλυθούν και ως προς τα πρότυπα διαχείρισης, τα συμμετοχικά πρότυπα διαχείρισης, παραδείγματι, μπορούν να είναι μια λύση, μας ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως και το δικαίωμα του πολίτη στη γνώση του πολιτιστικού προϊόντος ώστε να μπορεί να ε, ασκεί καλλιτεχνική δημιουργική δραστηριότητα αλλά και να ενημερώνεται αλλά και να έχει πρόσβαση ο ίδιος στο πολιτιστικό προϊόν. Πρόκειται για τη συμβάση του Φάρο που έχουν υπογράψει όχι όλες αλλά πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι λοιπόν εδώ ε, αλλάζουμε <coughs> τύπο διεκδίκησης και απέτησης ως προς το πολιτιστικό προϊόν. Πρέπει να το επιδιώξουμε αυτό για να ε, απαιτήσουμε το πολιτιστικό προϊόν στη θέση όχι του τουρίστα μόνο, αλλά και του πολίτη, εκείνου που μένει στη χώρα. Αυτό ισχύει για όλη την Ευρώπη και δει για την αδυναμία πρόσβαση σε γλωσσικό ή πολιτιστικό επίπεδο, ακόμα και σε χώρες που έχουν ε, προσφορά πολιτιστικού προϊόντος μόνο σε μία ή δύο γλώσσες που όμως δεν καλύπτουν την ε, ε, γλώσσα του ντόπιου πληθυσμού μεταναστών. Στο Μουσείο του Αιγυπτιακού Επαραδείγματι του, του Ορεινού έγινε κάτι το πρωτοποριακό. Έβαλαν τις ε, εξηγήσει των έργων, όχι μόνο στα Ιταλικά και τα Αγγλικά, αλλά και στην Αραβική γλώσσα και αυτό οδήγησε σε τεράστια αποδοχή από τον κόσμο, εκείνον ο οποίο θεώρησε ότι γίνεται αποδεκτό με τον τρόπο αυτό. Και νομίζω ότι εδώ μπορούμε να βελτιώσουμε σημαντικά την προσφορά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο και στον κύριο Σαμπιέρη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σα παρακαλώ όχι παραπάνω από δύο-τρία λεπτά αν γίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ακρόαση αυτή. Και θα ήθελα να τονίσω το, τη δουλειά των συναδέλφων στη Eurostat που στήριξαν αυτές τις συζητήσεις με τα στοιχεία που έχουν παράσχει. Ειδικά για την κινητικότητα και τα εμπόδια στην κινητικότητα είναι μία από τις προτεραιότητές μας. Το δουλέψαμε αυτό πέρσι και πρόπερσι. Ο καθηγητής Μόλεναρ ήταν ένας από τους καλεσμένους μας και θα συνεχίσουμε. Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα και ε, ε, έχω, πρέπει να έχουμε ένα αρκετά μεγάλο πυρήνα κρατών μελών για να υλοποιηθούν αυτές οι δραστηριότητες. Οι φορολογικές πολιτικές είναι κάτι το δύσκολο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα το ξαναβάλουμε ως προτεραιότητα όταν θα διαπραγματευτούμε ξανά ε, στο ε, Συμβούλιο. Τώρα για την έκθεση. Στηρίζω αυτά που είπε η κυρία Κώστα, γιατί τα ζητήματα είναι πολύ περίπλοκα. Και τα δεδομένα αυτό δείχνουν αν τα μελετήσει κανείς σε βάθος. Για παράδειγμα το χάσμα υπαίθρου και αστικού τοπίου δεν είναι τόσο τεράστιο ε, στα, σε ορισμένα κράτη-μέλη. Σε κάποιες ε, χώρες μέλη ε, το κατόφλι της φτώχειας είναι στα αστικό περιβάλλον και σε κάποιες άλλες χώρες το κομμάτι του πληθυσμού που είναι πολύ φτωχό είναι στην ύπεθρο και αυτό είναι πιο μεγάλο και σημαντικό ρήγμα το ρήγμα δηλαδή στα εισοδήματα των ατόμων. Ε, ε, πρέπει να βελτιώσουμε την ε, πρόσβαση στην παροχή των προϊόντων πολιτισμού και η προσέγγιση μας πρέπει να βασίζεται στην κοινότητα, όπως και το ίδιο κάναμε και με την πολιτιστική κληρονομιά. Δηλαδή πρέπει να εμπλέξουμε την τοπική κοινότητα. Η κουλτούρα, ο πολιτισμός να είναι μέρος της τοπικής κοινότητας και εκεί μπορούμε να απευθυνθούμε στους πιο ευάλωτους, σε αυτούς που ε, ε, δεν συμμετέχουν και που δεν συμμετέχουν γιατί δεν έχουν τα χρήματα, αλλά υπάρχουν και άλλοι που δεν συμμετέχουν γιατί δεν έχουν ενδιαφέρον και αυτό είναι αυτό που σκοτώνει τη συζήτηση. Πρέπει να αφυπνίσουμε, να ξυπνήσουμε το ενδιαφέρον. Θα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις προσπάθειές μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, Μπορεί και να έχετε δίκιο ότι ενδεχομένω η πολιτιστική προσφορά να μην είναι η ενδεδειγμένη για να φτάσουμε σε όλου. σω μπορεί και αυτό να, να αποτελέσει μια σκέψη που μπορεί να μα προβληματίσει. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Να δώσω τέλο το λόγο για άλλη μια φορά στον κύριο Στογεύσκη και να σα υπενθυμίσω ότι η προθεσμία υποβολή τροπολογιών είναι η Δευτέρα Μαρτίου στι 10 το πρωί και ψηφοφορία εδώ στην Επιτροπή θα γίνει στι 25 Απριλίου. Κύριε Στογεύσκη, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές και να απαντήσω εν συντομία σε όσα ακούστηκαν. Για την κυρία Ροντρίγκες, συμφωνώ απολύτως. Και εγώ υπογραμμίζω στην έκθεσή μου αυτό το εκπαιδευτικό εμπόδιο. Μιλώ για μια βασική εκπαίδευση η οποία θα επιτρέπει στον κόσμο να κατανοεί τα πολιτιστικά αγαθά. Το πώς θα μειωθούν οι δαπάνες ε, είναι ένα ζήτημα που αφορά τις ε, ε, τις ε, διοικητικές ε, αρχές. Ευτυχώς όμως φαίνονται, υπάρχουν μηνύματα από ολόκληρη την Ευρώπη που δείχνουν ότι αρχίζουν, αρχίζει να συνειδητοποιείται το γεγονός ότι τα παιδιά θα πρέπει να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα μουσεία και σε άλλα πολιτιστικά ιδρύματα. Το πρόβλημα που θέλω εγώ να αναδείξω είναι ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχουν μελέτες που πιστοποιούν ότι άνω του 50% του πληθυσμού δηλώνει ότι δεν ενδιαφέρεται για τον πολιτισμό. Και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Κυρία Μίχελς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που είπατε και, σας... και χαίρομαι πολύ για το σχόλιο αυτό. Δυστυχώς έχω περιορισμό λέξεων. Αλλά μέσω των τροπολογιών μπορούμε να εντάξουμε και κάποια ακόμα θέματα. Στα άρθρα 4 και 5 και 9 είναι αναγκαίο να υπάρξει μια επεξήγηση των όσων γράφω εγώ και είμαι αισιόδοξο ότι θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πάντως που είπατε ότι είναι πολύ μικρή η έκθεσή μου γιατί αυτό με διευκολύνει πολύ στο από εδώ και πέρα έργο μου. Κυρία Μπίλτ, σκόπιμα δεν αναφέρθηκα σε αυτόν τον ε, σε αυτόν τον πολιτισμό της ελίτ την Αβινιόν και αυτά, και αυτά τα φεστιβάλ που, που τις, τις πολιτικές εκδηλώσεις που, που αναφέρατε ξέρω ότι είναι λίγες αυτές στην Ευρώπη και με μικρή συμμετοχή ακριβώς γιατί είναι πάρα πολύ ε, μικρή συμμετοχή. Δεν, δεν, δεν τις επικρίνουμε βεβαίως αυτού του είδους τις εκδηλώσεις. Δεν τις αναφέρουμε καν όμως. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει και αυτό που θέτουμε στο επίκεντρο της προσοχής μας είναι κληρονομιά, ε, διατήρηση, συντήρηση των υποδομών. Τα βασικά. Πυκλομορφία πολιτιστική. Αυτά θέλουμε. Αλλά παρόλα αυτά σας ευχαριστώ. Επίσης, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε η κυρία Κώστα. Θεωρώ και εγώ ότι αυτή είναι ακριβώς η βασική τομή στους οποίους πρέπει να επικεντρωθούμε. Γι' αυτό και αναφέρθηκα σε αυτούς. Η σχέση μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών, η διάσταση του φύλου, η διαφορά εκεί είναι 2% ε, υπέρ των γυναικών, δηλαδή οι γυναίκες συμμετέχουν πιο πολύ στον πολιτισμό από ότι οι άνδρες. Και επίση συμφωνώ βεβαίω ότι χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία, περισσότερα δεδομένα και για τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω να ευχαριστήσω τη Eurostat. Από το 2012 έως το 2016 η Eurostat έκανε τεράστια βήματα. Πολύ υψηλή ποιότητα μάλιστα. Το ευρωβαρόμετρο και άλλα εργαλεία της Eurostat ε, καταγράφουν πλέον ε, και τον πολιτισμό και καθόλου τυχαίως δεν αναφέρω αυτό το στοιχείο και στην έκθεσή μου γιατί πιστεύω ότι ε, αξίζει να συνεχιστεί. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν όντως πολύ ενδιαφέρον τα όσα ακούσαμε σήμερα το απόγευμα όπως και η έκθεση βεβαίως 2 Μαρτίου στις 10 έχουμε την προθεσμία για την κατάσταση των τροπολογιών. Άντε λοιπόν τώρα, κουραστήκατε, να ξεκουραστείτε, το κερδίσατε μετά τις σημερινές συστήσεις, αύριο το πρωί στις 9, πάλι εδώ, στην ίδια αίθουσα. Και ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τους Δερμηνείς, λέει πολύ ευγενικά η Πρόεδρος, την ευχαριστούμε και ανταποδίδουμε.